Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, a warm welcome. Και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να καλωσορίσω τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας. Έχουμε τώρα ακρόαση για τον έλεγχο των άμεσων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζετε το γεγονός ότι πέρυσι είχαμε πολλές ε, ίδιες ε, άμεσες επενδύσεις, ε, ειδικά από μια μεγάλη ασιατική χώρα. Νομίζω γύρω στις 300 εταιρείε εξαγοράστηκαν ή και στήθηκαν από αυτή τη χώρα και ε, γι' αυτό, έγιναν έντονες συζητήσεις όσον αφορά τον έλεγχο των επενδύσεων εντός της Ένωσης και τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κομισιόν υπέβαλε σχετική πρόταση και δεν είναι δικό μου καθήκον να εξηγήσω την πρόταση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Μάλουστρομ εδώ που θα μας εξηγήσει την πρόταση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Λάγκε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά σε όσους δεν έχω δει ακόμα και σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτήν την ακρόαση στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Είναι πολύ επίκαιρη συζήτηση. Είναι θέμα που συζητείται σε πολλές χώρες και έχω έρθει σήμερα να σας μιλήσω για την πρότασή μας, για την εξέβρεση ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ελευθερία και την ασφάλιση ασφάλεια στι δημόσιε τάξει. Υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι ο καλύτερο ώρα για να φυτέψει κανείς ένα δέντρο ήταν πριν 20 χρόνια. Αμέσως επόμενη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για δεν, να κάνουμε κάτι σωστά για μια φορά, αλλά για ε, κάνουμε κάτι σωστά που θα έχει διάρκεια. Είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε και το μέλλον της Ένωσης εξαρτάται από το πώς θα προετοιμαστούμε για αυτό το μέλλον, όχι μόνο για αυτήν εδώ την πρόκληση, αλλά για όλες τις προκλήσεις που μας περιμένουν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα θεμέλια της Ένωσης. Και ε, δεν είναι εύκολο να έχουμε τη διορατικότητα για να αναγνωρίσουμε τις μελλοντικέ ευκαιρίες αλλά και τις απειλές, απλές αποφάσεις νωρίς ή πιο περίπλοκες και δύσκολες αποφάσεις αργότερα. Αυτό είναι κάτι που πάντα πρέπει να σταθμίσουμε. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ήταν σταθμισουμε πως γνωριζετε η ευρωπαικη ενωση ειναι και ηταν ανεκαθεν το πιο ανοιχτό περιβάλλον για επενδύσεις στον κόσμο. Στηρίζουμε τις ανοιχτές επενδύσεις, είναι μια βασική ε, οικονομική ελευθερία. Όμως δεν θα πρέπει να είμαστε και αφελείς, γιατί η επιθυμία για δράση στον έλεγχο των επενδύσεων είναι συνετή, αλλά είναι και ε, πιο ε, μακρόπνοη θα πρέπει να δούμε πώ θα αυξηθούν οι στρατηγικοί. Όπως είπε μάλλον και ο πρόεδρο Λάγκε, αρκετέ επενδύσει έχουν γίνει τον περασμένο χρόνο. Ορισμένε είναι κρατικέ επενδύσεις και ορισμένε άλλε στηρίζονται από ξένες ε, ε, κυβερνήσει. Όπου όμω αυτέ οι χώρε έχουν, ε, να αντιμετωπι... έχουν πολύ συγκεκριμένα ω εμπορικούς φραγμούς. Δεν είναι τόσο ανοιχτέ δηλαδή όσο είμαστε εμείς και δεν παίζουν με τους ίδιους κανόνες όπως εμείς. Έχουν λοιπόν δικά τους συμφέροντα τα οποία στηρίζουν και τα δικά τους συμφέροντα είναι κάποιες φορές, αλλά όχι πάντοτε συμβατά με τα δικά μας. Και γι' αυτό και ε, συζητάμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν για τον έλεγχο των ε, επενδύσεων. Έχουμε και ένα πάνελ ειδικών, του οποίους θα ακούσουμε γιατί είναι απαραίτητη μια τέτοια πρόταση τώρα, τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει και βέβαια μετά θα έχουμε και έρωτα απαντήσεις. Γιατί είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο τώρα, επειδή ο κόσμος έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει και οι επενδυτικές ροές. Παραδοσιακά οι επενδυτικές χώρες ήταν ε, χώρες που είχαν τις ίδιες αξίες με εμά. Όμως οι παγκόσμιες αγορές έχουν αλλάξει, και νέοι ισχυροί παίκτε αναδύονται που δεν, ε, έχουν πάντοτε, δεν τηρούν πάντα τις ίδιες προδιαγραφές ούτε τους ίδιους κανόνες και δεν παίζουν πάντοτε και θεμητά και δίκαια. Χρησιμοποιούν την πρόσβαση στις τεχνολογίες, στις υποδομές και στις πληροφορίες. Και χρειάζεται ίσως εμείς να προστατεύσουμε κάποια δικά μας ε, στοιχεία και πρέπει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ε, αλληλεξαρτώμενοι, περισσότερο από όσο το συνειδητοποιούμε. Και σημαντικές τομεί όπως η ενέργεια εξαρτώνται από ιδιαίτερες ε, ε, δεξιότητες και υπηρεσίες. Και δεν μπορούμε να αυτά να τα δώσουμε σε έναν ξένο επενδυτή χωρίς να αναλογιστούμε τον αντίκτυπο όλων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν κάθε κράτο μέλο να κατανοήσει πώ θα διαχειριστεί τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια. Αυτέ είναι ευαισθησίε, αλλά έχουμε και πιο ευάλωτα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο υποβάλαμε αυτή την πρόταση ώστε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στον έλεγχο των επενδύσεων, αν υπάρχει ήδη τέτοιο σύστημα και αν αποφασίσουν να εισάγουν τέτοιου μηχανισμού. Όπω ξέρετε, ούτε καν τα μισά κράτη-μέλη δεν έχουν τέτοιο τέτοιου μηχανισμούς αυτή τη στιγμή. Και ίσω και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, να μοιραστούμε πληροφορίε μαζί και να συνεργαστούμε. Και θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να είναι ενήμερα και να ενημερώνουν τους εταίρους τους για τέτοιους ε, επενδυτικούς εταίρους. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε μια πλατφόρμα για την ε, μοιρασιά της γνώσης, αντί να κάνουμε το ίδιο πράγμα 28 φορές, να κάνουμε κάτι και από κοινού για να εξοικονομήσουμε χρήματα και προσπάθειες και ε, ωφέλη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την πρότασή μας. Να δούμε δηλαδή ποιους μηχανισμούς έχουμε, ποιοι λειτουργούν, να βρούμε κάποια βασικά κοινά στοιχεία, να ορίσουμε τις καλύτερες πρακτικές, τη διαφάνεια, απουσία διακρίσεων, Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία, με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι στην Ένωση και που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου συστήματος ελέγχου. Οι χώρες να μπορέσουν να αναπτύξουν ε, ε, σχετικές νομοθεσίες, αλλά να έχουμε και την πεποίθηση μιας ε, κοινότητας. Και η συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών δεν σταματά εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένες γραμμές επικοινωνίας σε αυτό το τομέα και αυτό προσπαθούμε να αναπτύξουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη χώρο ώστε να συζητήσουν και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε διάφορα πράγματα. Πρώτον, συνεργασία μεταξύ των μελών, ε, ώστε να έχουμε μια, μεγαλύτερη, μια ευρύτερη εικόνα για τα, τους τρόπους ε, με τους οποίους γίνονται οι ξένες επενδύσεις, θα εντοπιστούν οι ανησυχίες, να δημιουργηθεί ένας χώρος για συζήτηση, ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών και η Κομισιόν να λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο συντονισμού όπως σας είπα, να δώσει στα κράτη-μέλη μια βάση ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Εμείς από πλευράς Κομισιόν θα διερευνήσουμε πιθανές απειλές στην ασφάλεια και σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί απειλή, να υπάρχει και μία μη δεσμευτική σύσταση και έτοιμα προς, ε, για επεξηγήσεις, αν χρειάζεται να προχωρήσει η επένδυση. Ε, η πρόταση αυτή δεν αναιρεί οποιοδήποτε δικαίωμα από τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, όταν έρχεται μια ξένη επένδυση σε μια χώρα, θα είναι αυτή η χώρα που θα ορίσει τελικά, θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι. Το, το σχέδιό μας είναι όχι να ελέγξουμε τις χώρες, αλλά να τις βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε, ούτε να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό ελέγχου. Πρόκειται για συνεργασία, για ανταλλαγή πληροφοριών και για βοήθεια παροχή βοήθειας προς τα κράτη-μέλη ώστε να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Ε, δεν θα πρόκειται για ένα εργαλείο προστατευτισμού. Φαίνεται εξάλλου από το ιστορικό μας ε, ότι είμαστε προσιλωμένοι στην ανοιχτή, ελεύθερη αγορά. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις προς τον ΩΣΑ και στον ΠΟΕ και στην οικοδόμηση μια νέα παγκόσμια τάξη, πράγμα που είναι πολύ πιο σημαντικό. Θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη στις ξένες επενδύσεις, τι χρειαζόμαστε και τι καλωσορίζουμε, δεν τι υποτιμούμε, δεν τι υποσκάπτουμε, αλλά πρέπει να μπορούμε να το συζητήσουμε περισσότερο σε ορισμένε περιπτώσει. Θέλουμε να επιτύχουμε τη μελλοντική ασφάλεια και όπως ε, ε, επειδή άρχισα με μια κινέζικη παροιμία, θα τελειώσουμε μια ελληνική παροιμία που λέει ότι μια κοινωνία προχωρά καλύτερα όταν ε, οι γέροντές της φυτεύουν δέντρα που ξέρουν πως δεν θα τους ε, ε, σκιάσουν ποτέ. Είναι δύσκολο οι πολιτικοί, οι νομοθέτες να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις πάντοτε, οι οποίες κάποιες φορές είναι πολύ γρήγορες και δεν συμφωνούν όλοι πως η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το φέλιμο. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, έγκυρες και άκυρες, αλλά η προστασία της ε, βασικής, των βασικών υποδομών είναι ένας προβληματισμός και θέλουμε να μπορέσουμε έτσι να κάπως να σχηματίσουμε και να δώσουμε μορφή στην παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι ένα καλό σημείο κίνησης. Είναι ένα σημαντικό σημαντικό βήμα μπροστά όσον αφορά ακριβώ το σχηματισμό της παγκοσμιοποίηση, βοήθεια προ τα κράτη-μέλη ώστε να λαμβάνουν τι αποφάσει του έχοντα γνώση των ε, πραγμάτων, εντοπισμό απειλών, προσαρμογή στο παγκόσμιο περιβάλλον, να προσπαθούμε να είμαστε μπροστά και έτσι να εξασφαλίσουμε πως οι πολίτες μας θα ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα ανθίζει και θα καινοτομεί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να προβλέψουμε και να οπλίσουμε την Ευρώπη ώστε να είναι επιτυχής και προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο ώστε να προχωρήσουμε. Ξέρω πως ο εισηγητής κ. Προύστα έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του μπροστά από το Συμβούλιο και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας. Ε, ευχαριστήσω και πάλι που διοργανώσατε τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Υπήρχε σαφής τάση προς το Κοινοβούλιο να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε δύο πάνελ. Το ένα θα εξετάσει τις δυσκολίες του ελέγχου των επενδύσεων και το άλλο με τα πρακτικά στοιχεία του ελέγχου. Στο πρώτο έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες. Με μεγάλη χαρά έχουμε τον Νέιμεν Μίρ μεταξύ ημών που είναι ο αναπληρωτής υφυπουργός ε, του Υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος του ΣΦΙΟΥΣ, την υπηρεσία στις ΗΠΑ που ελέγχει τις επενδύσεις. Και για πρώτη φορά έχουμε την τιμή να σας υποδεχτούμε, κύριε Μύρ, για να μας εξηγήσετε την προσέγγισή σας. Έχουμε μετά την Ιέβα ε, Γιάουντζίμε, του Υπουργείου Οικονομικών στην ε, Λετωνία. και ένα τρίτο άτομο από την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία ε, της Γαλλίας, τον κύριο Φεντερίκ Βερλέ. Καταρχήν ο κύριος Μύρο όμως για την πρώτη παρέμβαση. Σα ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Χαίρομαι που θα σα μιλήσω για τη δική μα εμπειρία για την, τον έλεγχο των επενδύσεων. Ποια είναι η προσέγγισή μα Πρέπει να καταλάβετε ότι οι ΗΠΑ ε, έχει δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε διάφορε κυβερνήσει, επί δεκαετίε να κρατήσει ένα ανοιχτό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Ε, οι ξένε επενδύσει ε, είναι υποφελεί για την οικονομία μα, από την εμπειρία μα φαίνεται αυτό, και συνεισφέρουν στο ΑΕΠ μα ε, δημιουργούν θέσει απασχόληση, εξαγωγέ και κοινοτομία. Είμαστε λοιπόν στην, συμφωνούμε στο γεωμικό σχήματος με την, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κίνδυνοι. Πριν από 30 χρόνια ξεκινήσαμε όμως να σχεδιάζουμε μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τους βασικούς κινδύνους ε, που συνεπιφέρουν οι ξένες επενδύσεις. Ε, η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανήκει στο Υπουργείο ε, Οικονομικών ε, με τη συμμετοχή πολλών Υπουργείων, συναρμόδιων Υπουργείων, είναι υπεύθυνη για αυτή τη διαδικασία. Θα σας πω για κάποιες διαδικασίες και κάποια σχόλια για το πώς αντιμετωπίσουμε το εξελισσόμενο περιβάλλον των ξενοπενδύσεων. Ξεκινούμε με την υποβολή ε, φακέλου στην Επιτροπή και τελειώνει με την ολοκλήρωση του φακέλου. Όταν ολοκληρωθεί αναθεωρούμε, ε, επανεξετάζουμε το φάκελο μέσα σε 30 μέρες. Ε, μπορούμε να δώσουμε άλλες 45 μέρες, συνολικά δηλαδή 75 μέρες για την όλη διαδικασία. Μέσα αυτό το διάστημα όλη η Επιτροπή και όσοι ασχολούνται με, την, με τις φορείς των ε, υπηρεσιών πληροφοριών ε, συναντιόμαστε σε εβδομαδιαία ε, βάση για να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Αν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, ενημερώνεται το Κογκρέσο και εάν δεν υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια, θεωρείται ότι το μέλος το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση είναι safe harbor όταν όμως υπάρχουν προβλήματα εθνικής ασφάλειας, τότε γίνεται μια γραπτή ανάλυση που αποφασίζει με βάση αυτή, αν μπορούμε να μετριάσουμε τον κίνδυνο, πώς, με τη διαπραγμάτευση, ε, ούτως ώστε να υπάρχουν μετριασμό μετριασμός του κινδύνου. Εάν δεν μπορούμε να μετριάσουμε τον κίνδυνο, τότε παραπέμπουμε το θέμα στον πρόεδρο, ο οποίος με διάταγμα ή με νόμο μπορεί να απαγορεύσει την συναλλαγή αυτή. Τώρα, κάποια χαρακτηριστικά που πιστεύουμε ότι μας βοήθησαν να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία είναι πολύ αποτελεσματική και ε, ε, σεβόμαστε τα θέματα της ασφάλειας, ε, κρατώντας ανοιχτό περιβάλλον για τις επενδύσεις, ελκυστικό κτλ. Καταρχάς, το ΣΦΙΟΥΣ ασχολείται με θέματα εθνικής ασφάλειας αμυγός. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό για να εξετάσουμε την όλη διαδικασία όλα τα θέματα ε, της εξέτασης ξεκινούν με αυτή την προσέγγιση και τελειώνουν με αυτή την προσέγγιση. Ε, καθορίζουν τις εμπορικές αποφάσεις ε, και η κυβερνητική παρέμβαση υπάρχει μόνο σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Δεύτερον, η διαδικασία αυτή δεν είναι μια τομεακή διαδικασία που απαγορεύει τις επενδύσεις. Ε, λαμβάνουμε τις αποφάσεις ανά επένδυση, επιτρέπουν τις ε, επενδύσεις που ε, είναι ε, συμβατές με την εθνική ασφάλεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ε, ο, ο φορέας μας ε, ελέγχει όλες τις επενδύσεις. Όσες επενδύσεις δεν δημιουργούν θέματα ασφάλειας, γενικά μπορούν να προχωρήσουν ε, ανεμπόδιστα. Ε, εξετάζουμε επίσης ε, αναλυτικά στοιχεία. Κάθε επένδυση ε, αναλύεται ε, με βάση την πολιτική, από εμπειρογνώμονες, από διάφορους τομείς. Αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι της εθνικής ασφάλειας ε, περιπτωσιολογικά με βάση τρεις παράγοντες. απειλή, ευαλωτότητα και συνέπειες. Η ανάλυση της απειλής εμπεριέχει μια αξιολόγηση ε, του αγοραστή να προκαλέσει βλάβη στην εθνική μας ασφάλεια και εδώ ε, συμμετέχει και, συμμετέχουν και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Επίσης, αναλύουμε τις ε, συνέπειες. Βλάβες, συνέπειες που... και τι μπορεί να εκμεταλλευτεί η συγκεκριμένη επένδυση. Αναλύουμε και τους τρεις αυτούς παράγοντες ε, και δεν εξετάζουμε καθόλου τα οικονομικά ωφέλη. Οι περισσότερες επενδύσεις που εξετάζουμε ε, στην πραγματικότητα παίρνουν το πράσινο φως, ε, χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση. Επίσης, είμαστε αναλογικοί στην προσέγγιση μας σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο. Δεν δρούμε εάν αν άλλοι φορείς είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους, τα προβλήματα και τους κινδύνους ε, της επένδυσης. δεν θέλουμε να μπλοκάρουμε την επένδυση. Προσπαθούμε, ε, αν μπορούμε, να μετριάσουμε τον κίνδυνο, ούτω ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα όσο μπορούμε. Το γεγονό ότι μια επένδυση μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο στην εθνική ασφάλεια δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα μπλοκάρουμε την επένδυση αυτή. Η μεγάλη πλειοψηφία των επενδύσεων που ελέγχει ο φορέας μας ως ε, παίρνει το πράσινο φω. Αλλά ακόμα και εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, πολύ συχνά τελικά βρίσκουμε τα μέτρα, ούτως ώστε να μετριάσουμε τον κίνδυνο της επένδυσης. Ε, είμαστε έτοιμοι να συστήσουμε στον Πρόεδρο να απαγορεύσει την επένδυση, εάν θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι αποτελεσματικά, δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Ιστορικά, ένας μικρός αριθμός ε, επενδύσεων τελικά απαγορεύεται και δεν παίρνει την έγκριση. Πέμπτος, πέμπτον, ε, η διαδικασία μας είναι αποτελεσματική και λογοδοτούμε Επίσης είναι ε, εμπιστευτική, δια νόμου δεν ε, δημοσιεύουμε καθόλου πληροφορίες, ε, όλα τα στοιχεία του φακέλου παραμένουν εμπιστευτικά, ε, εκτός από τις δράσεις φυσικά του Προέδρου. υπάρχει εμπιστοσύνη σε εμά και στην ικανότητά μας να κρατήσουμε την εμπιστευτικότητα και αυτό δίνει κίνητρα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν το φάκελό τους στους φιούς. Ε, η διαδικασία ήταν πολύ, ε, πολύ δραστήρια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, για να αντιμετωπίσουμε θέματα εθνικής ασφάλειας. Τα βασικά χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα ήταν βασικά για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους κινδύνους, ε, κρατώντας ένα εποφελές επενδυτικό περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επενδύσεις από το εξωτερικό στις ΗΠΑ το 2015 και το 2015 το ΣΦΙΟΥΣ ήταν πολύ δραστήριο. Ε, είχαμε πάρα πολλές υποθέσεις. Από το 2009 μέχρι το 2016 ε, εξετάσαμε το 7,8 των υποθέσεων και το απορρίψαμε. Ε, επίσης ε, έχουμε και εμείς ανάλογες ε, ανάλογα ερωτηματικά με αυτά που έχετε στην Ευρώπη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θέτουν οι ξένες επενδύσεις εδώ στην Ευρώπη. Ιδίω οι νέε ε, τεχνολογίες, ε, οι κρίσιμες υποδομές, ε, καθώς και επενδύσεις που στηρίζουν την πολιτική των κυβερνήσεων για να υλοποιήσει βασικούς στόχους. Θέλουμε να κρατήσουμε το ανοιχτό μας περιβάλλον και να κρατήσουμε τις βασικές μας αρχές ε, διαφάνεια, κράτος δικαίου, ε, ανοιχτή αγορά. Τα, οι βουλευτές μας, εθνικοί μας βουλευτές, έχουν υποβάλει νομοθεσία για να αναθεωρήσουν τη διαδικασία του φίους. Ε, μπορούμε όμως να, μπορεί να αλλάξει η αρμοδιότητά μας και να υπάρξουν αλλαγές στη διαδικασία, μάλλον με τη νέα νομολογία, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά που ακούσατε να σας περιγράφω δεν θα αλλάξουν. Ε, η ασφάλεια των ε, συμμάχων μας, ε, ξέρουμε ότι ενισχύει και τη δική μας ασφάλεια, οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, τι κάνετε εσείς στην Ευρώπη και η εξελίξη στην Ευρώπη. οι νόμοι που έχετε εδώ στην Ευρώπη μπορεί να έχουν άμεσες συνέπειες, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και στην αμερικανική ασφάλεια. Επιπλέον, εξετάζουμε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι για να προστατεύσουν τις τεχνολογίες και, τις, και το δυναμικό τους, Ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί να μην εξετάσετε με τον ίδιο τρόπο τις επενδύσεις ε, όπως και εμείς, αλλά πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί και το βασικό για μας είναι να έχουμε μια καλή σχέση συνεργασίας. Ε, θα συνεχίσουμε το διάλογο, τόσο ώστε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές και είμαι έτοιμος να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Και δίνω τώρα το λόγο στη Λετωνία. Chairperson. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε μέλη της Επιτροπής σας αποτελεί τιμή μου να παραβρίσκομαι σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ Πρόεδρε Λάγκη για την ε, διοργάνωση αυτής της σημερινή ακρόαση. Ε, οι ε, ξένε επενδύσει καθίστανται όλο ένα και πιο σημαντικέ λόγω τη γενικότερη κατάσταση παγκοσμιοποίηση. Και εγώ στο πλαίσιο τη παρουσίασή μου θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Στον μηχανισμό του ελέγχου των ξένων επενδύσεων στη Λετωνία, καθώ ε, θα αναφερθώ και στι ε, προτάσει ε, που κάνουμε εμεί σε σχέση με τα όσα πρότεινε η Επιτροπή. Κατά τη δική μα άποψη, είναι σημαντικό να γίνει σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία, έτσι ώστε να σα εξηγήσω και ποια είναι η θέση τη Λετωνία σε αυτό το πλαίσιο. Καταρχήν να σα εξηγήσω ποια είναι η θέση σε σχέση με τι εξάνε επενδύσει τη Λετωνία. Εμεί είμαστε μια μικρή ανοιχτή κοινωνία και έχουμε αναγνωρίσει το όφελο που μπορούν να αποφέρουν αυτέ οι εξάνε επενδύσει. Ωστόσο, το ύψο του είναι σχετικά μέτριο. Για παράδειγμα, κατά τα τελευταία τρία έτη, ε, οι άμεσε ξένε επενδύσει ανήλθαν σε περίπου 3% του ΑΕΠ. Ε, και λόγω των πολιτικών σοκ ε, που δέχθηκε η χώρα μας ε, δεν ήταν δυνατόν να αυξηθεί ο σχετικός ρυθμός των, ξένων επενδύσεων. Τώρα, η Ε, υπήρχε συγκεκριμένη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία από ξένες επενδύσεις, αλλά επειδή χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στην ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία, ε, εφαρμόστηκαν νέε νέες διατάξεις που είχαν αντίστοιχο αντίκτυπο στην ελκυστικότητα, στην ελκυστικότητα της αγοράς μας. Μέσω τώρα ε, ε, μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική και αντίστοιχων ε, ενεργειών από την γείτονα χώρα μα είδαμε ε, πως υπάρχει ένας υπαρκτός ε, κίνδυνος ε, για τη δημόσια ασφάλεια της χώρας μας και γι' αυτό αποφασίσαμε να προβούμε σε νομοθετικά μέτρα, συμμορφώνουμε πάντα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβήκαμε σε μια νομική ανάλυση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποιο θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος μιας, ενός τέτοιου νόμου στις επενδύσεις, ποια είναι τα νομικά πλαίσια που ισχύουν σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία ε, και το ε, ποια είναι, ποιο είναι το υφιστάμενο νομικό ε, πλαίσιο σε εμά. Επίσης εξετάσαμε τις δυνατότητες νομική προσφυγή και ποιο ήταν ο υφιστάμενο νόμο. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέταση που κάναμε, τον Μάρτιο του 2017, 13 Μαρτίου, πέρασε, υιοθετήθηκε δηλαδή ο νέος νόμος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται ε, σε επενδύσεις, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εθνική ασφάλεια, ε, την κρίσιμη υποδομή επίπεδου Β σε κρατικό επίπεδο ή για, την ευρωπαϊκή, ε, για τις ευρωπαϊκές κρίσιμες υποδομές. Υπάρχουν 26 επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν αυτές τις ε, προϋποθέσεις του νόμου Εθνική ασφαλείας ε, και ε, λογίζονται ως επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Θα ήθελα τώρα να εξηγήσω στο κοινό σας το πόσο προσεκτικοί προσπαθήσαμε να είμαστε προκειμένου να επιτύχουμε την ισορροπία ανάμεσα Αφενό στην ανάγκη του να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλεια και από την άλλη πλευρά να παραμείνουμε ελκυστικοί απέναντι στις ξένες επενδύσει. Θα ήθελα τώρα να σα εξηγήσω τις δικέ μας προτάσεις σε σχέση με την πρώτα που συζητείτε και στην ε, ομάδα εργασία του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Όπω ανέφερε σωστά ο πρόεδρο Juncker στην ομιλία του State of the Union, ε, δεν είναι κανένα από εμά ένα ε, αφελή ελεύθερα εμπορευόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να προστατεύσουμε τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο χρειαζόμαστε τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Ευχαριστούμε λοιπόν την Επιτροπή για την υποβολή αυτή τη πρόταση, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσει αρκετό χρόνο στις συζητήσεις αν είχε συνοδευτεί αυτή η πρόταση από μια αξιολόγηση αντικτύπου. Ίσως να φαίνεται δηλαδή κάτι το περιττό, κάτι το γραφειοκρατικό μια τέτοια αξιολόγηση αντικτύπου στο πλαίσιο ακριβώ και των τεχνολογιών που υπάρχουν σήμερα. Ωστόσο, η διοργανική συμφωνία που ισχύει ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τη Ένωση και την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την καλύτερη νομοθεσία ε, που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2016 και αυτή δεν είναι κάτι το τυπικό. Έχει συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή την βελτίωση της διαδικασίας νομοπαραγωγής. Η εν λόγω λοιπόν διοργανική συμφωνία αναφέρει με σαφήνεια ότι τα τρία αυτά θεσμικά όργανα συμφώνησαν ε, σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα των αξιολογήσεων αντικτύπου για την βελτίωση των νομοθετικών προτάσεων τη Επιτροπή. Ε, τέτοιου είδου αξιολογήσει αντικτύπου υπάρχουν για να βοηθούν ακριβώ τα τρία θεσμικά όργανα να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένε αποφάσει. Α, τώρα, μια σειρά από κράτη-μέλη ε, συμφώνησαν ε, ως πως το ότι θα πρέπει να δοθεί ε, συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να πάντοτε να έχουμε κατά το πόσο σημαντικό είναι ακριβώς να εστιάσουμε στην καλύτερη ε, νομοθεσία. Ε, εμείς λοιπόν χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση, αλλά υπάρχουν μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα. Καταρχήν, νομική βάση. βασίζεται η πρόταση στη νομική βάση του άρθρου 207 παράγραφος 2. Ε, το εν λόγω άρθρο αναφέρεται ρήτα στην εμπορική πολιτική. Αλλά ο έλεγχος των ξέων επενδύσεων αποτελεί εμπορική πολιτική ή όχι. Είναι κάτι το οποίο ε, παραμένει προσεζήτηση. Επίσης, το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει μία παράγραφο 6, η οποία αναφέρεται στην εχώρηση της αρμοδιότητας σε ό,τι αφορά τον τομέα της εμπορικής πολιτικής και ορίζει ότι δεν παρισφρέει στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωση και κρατών μελών. Αυτό μα οδηγεί στο δεύτερο πρόβλημα η δηλαδή πρόταση ε, έχει τη μορφή κανονισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι άμεσα εφαρμοστέ από τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν μία σειρά από που περιλαμβάνονται στη μη δεσμευτική γνωμοδότηση της Επιτροπής, ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά και τον ορισμό τους, ε, του screening, αυτό του ελέγχου, ουσιαστικά δεν, δεν συνάδει με αυτήν την νομική μορφή τη πρόταση τη επιτροπή, δηλαδή ως κανονισμό. Ή θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν, να μην είναι δηλαδή πλέον κανονισμό. Θα πρέπει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα ε, πλαίσιο συνεργασίας για τα κράτη-μέλη. Γιατί ένα πλαίσιο συνεργασίας είναι ακριβώς εκείνο που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ θα υπάρχουν όμως ταυτόχρονα και δεσμευτικές ε, γνωμοδοτήσεις. Ούτως ή άλλως ε, γνωρίζουμε ε, καλά ότι υπάρχει μεγάλη συνέντευξη μεταξύ των κρατών μελών. Το εν λόγω δηλαδή πλαίσιο δεν θα χρησιμοποιούνταν μεταξύ των κρατών μελών για να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλα κράτη-μέλη. Άλλοι αποφασιστικοί παράγοντες ο καθορισμό των αποφασιστικών παραγόντων σε ό,τι αφορά δηλαδή τον έλεγχο ξένων επενδύσεων σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να επαφέται στα κράτη-μέλη. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε, οι οποίε συλλέγονται για αυτέ τι ξένες επενδύσει, αυτέ ε, ε, αυτές συλλέγονται πάντοτε από τι εθνικέ υπηρεσίε ε, πληροφοριών και θεωρούνται ω κρατικά μυστικά. Οπότε δεν μπορούν εύκολα να διαβιβάζονται σε άλλου. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε λοιπόν τώρα ένα δίκτυο των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής σας, ε, νομίζω πως στους επόμενους έξι μήνες στο πλαίσιο της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας αλλά και η συζήτηση που θα κάνετε σήμερα εδώ θα βοηθήσουν την ομάδα εργασίας να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν ε, τα όσα γνωρίζουμε σε επίπεδο εμπειρία τεχνογνωσίας αλλά και τα όσα μπορούμε να επιτύχουμε σε επίπεδο τεχνολογία έτσι ώστε να επιτύχουμε το κατάλληλο, την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στι προτεραιότητέ μας λαμβάνοντα ε, πάντοτε υπόψη τις αρχές τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα, ε, όπω αυτέ έχουν κατοχυρωθεί στι συνθήκε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σαφέ μήνυμα, λέει ο πρόεδρο και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρίκη από Καλημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με καλέσατε για να μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το μηχανισμό ελέγχου των ξένων επενδύσεων στη Γαλλία. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ποια είναι η βάση της διαδικασίας μας, εν συνεχεία να σας πω ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής τη διαδικασία ε, για την ε, εξέταση των αιτήσεων και εκχώρηση άδεια και στο τέλος θα σας πω ποια είναι η άποψη της γαλλικής ε, κυβέρνησης για την πρόταση της Κομισιόν. Η βάση της διαδικασίας είναι ότι έχουμε μια αρχή και κάποιες εξαιρέσεις. Η αρχή ποια είναι η ελευθερία των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Γαλλίας και των ξένων χωρών, του εξωτερικού και οι εξαιρέσει είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται σε μια πρώτερη άδεια των ξένων επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς περιορισμένους όπως είναι η εθνική άμυνα ε, που μπορεί να διαταράξουν την δημόσια τάξη και όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την εγγύηση της ομαλής λειτουργίας της χώρας. Όλα αυτά ε, με σεβασμό ε, των ευρωπαϊκών συνθήκων έχουμε τρία κριτήρια σορευτικά. Καταρχάς, Έχουμε τη διαδικασία αδειοδότησης, την, προέλευση του επενδυτή, τη φύση της δραστηριότητας και ποια είναι η εταιρεία στόχος στη Γαλλία της επένδυσής του. Κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα στους επενδυτές που, έχουν, που προέρχονται από τον ΕΟΧ και τον υπόλοιπο κόσμο, καταρχάς. Η φύση της δραστηριότητας ή της επιχείρησης, καταρχάς όταν υπάρχει έλεγχος ε, μιας εταιρείας, ε, γίνεται εξέταση. Ε, όταν έχουμε την εταιρική έδρα στη Γαλλία, ε, τους ελέγχουμε επίσης και για τους επενδυτές εκτός ΕΟΧ, ε, όταν ξεπερνάμε το 33,3% ε, κατοχής κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου, πάντα επίσης γίνεται έλεγχος. Τώρα, η δραστηριότητα που ελέγχεται αφορά μπορεί να είναι δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την δημόσια τάξη ή τα εθνικά συμφέροντα ή την εθνική άμυνα. Και έχουμε και ένα κανονισμό που περιορίζει το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων που προανέφερα. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις όπου ο επενδυτής προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως σας είπα, και υπάρχουν διάφοροι τομείς οι οποίοι αναφέρονται, την κρυπτογράφηση, όταν μια εταιρεία στόχος ε, έχει μυστικά που σχετίζονται με την εθνική άμυνα, παραγωγή όπλων, εξοπλισμού, ε, πυρίτιδας κτλ. Όταν έχουμε με, δραστηρι... που η δραστηριότητά τους ε, ενδιαφέρει το Υπουργείο Άμυνας και όταν η παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων είναι ουσιαστική για την ε, εξασφάλιση της δημόσιας ε, τάξης ή της εθνικής άμυνας. Δηλαδή, ε, παροχή και ανεφοδιασμό σε ενέργεια, σε νερό, υπηρεσίες μεταφορών, εκμετάλλευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάσταση, εγκαταστάσεις που είναι σημαντικές για την άμυνα και την προστασία της δημόσιας υγείας για τις επενδύσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες και μόνο. Καλύπτουμε τις δραστηριότητες στον τομέα των, των τυχερών παιχνιδιών, ε, παθογενών ιών, επίσης ε, υλικού για την παρακολούθηση τηλεφωνικών υποκλοπών και παρακολουθήσεων, αξιολόγηση και πιστοποίηση της ασφάλειας ε, λόγω των, ε, της παροχής τεχνολογικών προϊόντων, ε, επίσης τεχνολογίες ε, διτής χρήσεως. Ποια είναι η διαδικασία τώρα. Τρεις φάσεις ε, διακρίνουμε. Η πρώτη φάση είναι η υποδοχή της, υποβολή, υποβολή μάλλον της αίτησης σε κάποιο Υπουργείο, κυρίως του Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει να γίνει αίτηση για ε, για πρώτερη άδεια ή επίσης μπορεί ε, το ενδιαφέρομενο να μας ζητήσει από τις γαλλικές αρχές να του πούν αν ή όχι ανήκει στην κατηγορία ε, που καλύπτεται από φορολογικές συμφωνίες. Τα λεγόμενα «ρεσκρίστα» στα γαλλικά, φορολογικές συμφωνίες. Η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών είναι υπεύθυνη με την ε, βοήθεια των διαφόρων Υπουργείων ανάλογα με το θέμα και τον τομέα. Η τρίτη φάση είναι η κοινοποίηση της, απόφαση ε, απόφασης μέσα σε δύο μήνες από τη στιγμή υποδοχής του πλήρους φακέλου στο βαθμό που βεβαίω η απουσία ε, απόφαση σημαίνει σιωπηλή άδεια. Ο Υπουργός δίνει την απάντηση τελικά είτε η επιχείρηση δεν, δεν ανήκει σε, στην κατηγορία που πρέπει να υποβληθεί άδεια ή μπορεί να υποβληθεί ε, απλή άδεια ή άδεια με προϋποθέσεις. Ή μπορούμε να αρνηθούμε την επένδυση σε περίπτωση που αιτιολογήσει την άρνηση αυτή ο αρμόδιος υπουργός. Οι επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες με προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές προϋποθέσεις. Αφορούν τη διατήρηση μέσω του της επένδυσης, της διαιώνησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων ε, ή της τεχνογνωσίας της εταιρείας στόχου, ε, ακαιρεότητα, συνέχεια και αδιάκοπτη συνέχεια του ανεφοδιασμού, προστασία της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντα υπόψη επίση και τι συμβατικέ υποχρεώσει τη επιχείρηση που εξαγοράστηκε. Η άρνηση τώρα τη άδεια έχουμε δύο λόγου. Ε, έχουμε τεκμήρια ότι η επένδυση ε, με την επένδυση μάλλον ε, γίνεται ουσιαστική παράβαση σε κάποιους νόμους. Έχουμε να κάνουμε με διαφθορά, λαθρεμπόριο, τρομοκρατία, αμφιβολίες για τον επενδυτή δηλαδή ή δεν έχουμε τα στοιχεία ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι διασφαλίζουμε την εθνική ασφάλεια ε, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουμε, μπορούμε να δώσουμε άδεια με προϋποθέσεις. Εάν δεν τηρούν οι προϋποθέσεις μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις οικονομικές, τελωνιακές και ποινικέ. Πολύ σύντομα τώρα θα σας παρουσιάσω την θέση των γαλλικών αρχών σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν, μια και το θέλαμε αυτό και την... θέλαμε αυτή την πρόταση και την υποστηρίζουμε. Είμαστε στη διάθεσή σα για οποιασδήποτε ερωτήσει. Τρει uh, uh, Τρεις πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις ε, όσον αφορά τον έλεγχο των ε, επενδύσεων. Τώρα έχουμε μισή ώρα για ερωτήσεις. Να θυμίσω σε όλους ότι πρόκειται για ακρόαση, όχι για ε, χρόνο και συζήτησης. Είναι χρόνος ερωτήσεων προς τους εμπειρογνώμονές μας. Πρώτα, για 1,5 λεπτό θα ακούσουμε τον εισηγητή και μετά οι υπόλοιποι όσοι θέλουν να θέσουν ερωτήσεις θα έχουν το λόγο για ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Προύστ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε τόσο γρήγορα και γιατί δείχνετε και πάλι την ικανότητά σας να ακούτε και να κάνετε διάλογο ακόμα και σε ακαθόδη ζητήματα. Έχω δύο ερωτήσεις και δύο-τρεις ερωτήσεις στους διάφορους ε, ομιλητές που θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ, κυρίως στον κύριο Μύρ που έρχεται από μακριά ε, μέσα σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο, ξέρουμε, στις ΗΠΑ. Προς εσάς, Επίτροπε, είπατε 12 χώρες έχουν ήδη φτιάξει σχετικούς μηχανισμούς, αλλά έχετε κάποια ενημέρωση από τις εμπειρίες που έχουν αυτές οι χώρες με τη λειτουργία αυτών των μηχανισμών. Για παράδειγμα, μειώνονται οι επενδύσεις, οι ξένες επενδύσεις σε αυτές τις χώρες, ε, βέβαια γνωρίζοντας ε, και λέγοντας ότι δεν είμαστε κατά των ξένων επενδύσεων, αλλά ε, είμαστε κατά των παράξενων επενδύσεων. Μιλήσατε επίσης για πριν από λίγο για ένα είδος ε, μοιρασιά συντονισμού, γιατί όντως εγώ συμφωνώ με τη δική σας ανάλυση για το θέμα ότι εφόσον θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, η ευρωπαϊκή διάσταση είναι η κατάλληλη για να μπορούμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια μας. Τι μπορεί να μας εγγυηθεί λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει πραγματικά Ε, θα μπορεί όντως να συνδυάσει τις πληροφορίες ε, οι οποίες πρέπει να είναι όμως καλής ποιότητας για να υπάρχει πραγματική ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη. Και έπειτα θα ήθελα να γνωρίζω τι σημαίνει ε, ο ότι έχετε ένα μηχανισμό διήθησης ε, φιλτραρίσματος ε, σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα. Επίση, ξέρουμε ότι ορισμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν περίπλοκα συστήματα ε, δημοσιονομικά, προσπαθούν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να κρύψουν ποιος είναι ο, ο αρχικός επενδυτής με διάφορα δημοσιονομικά οικοδομήματα. Πώς ε, παίρνετε την τελική πληροφορία λοιπόν και έπειτα για τις επαφές και αυτό περισσότερο προς τον κύριο Μύρ. Έρχεστε σε επαφή με την άλλη χώρα όταν μια επένδυση αγγίζει μια επιχείρηση στην επικρατεία σας και για παράδειγμα μια αμερικανική εταιρεία έχει ε, ε μετοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω τώρα τους κοιόδης ηγητές αν έχουν ερωτήσεις. Κύριε Σταμπάτη, θέλετε να θέσετε ερώτηση. Συμφωνώ με τα όσα μας είπε η επίτροπο, Πραγματικά ήταν ισορροπημένα και ανταποκρίνεται ε, και στις ε, απόψεις ε, του ΕΣΕΡ. πραγματικά ο κόσμος μας σήμερα είναι ένα ανοιχτό μόρφωμα εντός εισαγωγικών όπου οι ξένες επενδύσεις, οι διάφορες μπορούν ε, να λαμβάνουν χώρα, αλλά βέβαια υπάρχουν εκεί μία σειρά από μεθοδεύσει και σκοπιμότητες ε, απέναντι στι οποίες θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε ε, και μας ενημέρωσε και ο συνάδελφος από τις ΗΠΑ το πώς υπερασπίζονται εκεί τα συμφέροντά τους ε, και νομίζω πως ε, ε, εδώ τίθεται και ένα ζήτημα επικουρικότητας ότι δηλαδή υπάρχουν και ειδικοί σε εθνικό επίπεδο και από εκεί και μετά και σε υπερεθνικό επίπεδο αλλά σίγουρα είναι σημαντικό να γίνεται ένας διάλογος εδώ ανάμεσα στα κυρίαρχα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ε, εκείνο που θα ήθελα να ξέρω είναι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις σχετικά με τις εμπειρίες των επιμέρους χωρών ως προς το όφελος τελικά ή όχι τέτοιων επενδύσεων για το σύνολο της οικονομίας. Ή υπάρχουν εκθέσεις, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά επενδύσεις οι οποίες έχουν στόχο μόνο και μόνο την άντληση τεχνογνωσίας από τη συγκεκριμένη χώρα. Οπότε θα ήθελα να γνωρίζω, έχουν συνταχθεί τέτοιου είδου εκθέσεις. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο έχει το λόγο ω αστιώδη εισηγητή, ε, θα ήθελα να προσθέσω ένα ερώτημα ε, το οποίο απευθύνω και στου τρει εδώ μιλητέ του πάνελ καθώς μας εξέδεσαν διαφορετικά θέματα ο καθένας. Ε, η στοχοθέτηση αυτών των επενδύσεων, η ποιότητά τους και η επίπτωση που έχουν στην τοπική οικονομία είναι ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δηλαδή, δημιουργία θέσεων εργασία, προστασία του περιβάλλοντο τέτοιου είδου κριτήρια λαμβάνονται με βάση τη δική σας εθνική εμπειρία είναι ε, στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη και στο πλαίσιο ενός ε, screening σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Ξεκινήσατε με μια, με μια, γαλλική, ναι, με μια κινέζικη παροιμία και τελειώσατε με μια ελληνική παροιμία. Αυτό μου θυμίζει τον Πειραιά, το λιμάνι του Πειραιά. Τι γίνεται με αυτή τη στρατηγική επένδυση. Αυτός, αυτό το λιμάνι είχε μία πολύ ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία που έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία του. Ε, Όμω η ελληνική κυβέρνηση ήταν αναγκασμένη να ζητήσει από έναν επενδυτή να πάρει στα χέρια ένα ουσιαστικό στοιχείο τη ελληνική οικονομία. Άρα αυτό έχει να κάνει με την εθνική κυριαρχία τη Ελλάδα. Και, και χρησιμοποιήθηκε ε, η επένδυση αυτή στον Πειραιά τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προσπαθούσε να πείσει τα κράτη-μέλη να έχουν πραγματικά μέτρα αντι-dumping κατά των φωτοβολταϊκών τόξων της Κίνας. Υπάρχει λοιπόν από τη μία ε, τα δημόσια οικονομικά, από την άλλη έχουμε επενδύσει που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία, γιατί μπαίνουν πολύ περισσότερα χρήματα κτλ. Και τι κάνει ένα κράτο όταν δέχεται τρομακτικέ πιέσει. μια πρώτη ερώτηση στον Αμερικάνο φίλο μας που τον ευχαριστώ και που ήρθε εδώ και που είναι από τον... Μην ξεχνάτε ότι ε, το γραφείο για τις αιτήσει ασύλου είναι δίπλα εδώ. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην αμερικανική πολιτική ε, και στην ε, πολιτική σας για τις δημόσιες προμήθειες. Έχετε μια στάση πολύ περιοριστική που μειώνει την δράση ας πούμε, και, ε, το μερίδιο των ξένων επενδυτών. Και μια ερώτηση προς την Επίτροπη. Καταλαβαίνω που είναι η συζήτηση στην Ευρώπη. Μου κάνει εντύπωση η δηλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη σήμερα επιτέθηκε στην ε, Apple, στην Google ε, μέσω της κυρίας Βεστάγκερ ε, είναι γιατί είναι όλη η Ευρώπη από πίσω παρά την ομοφωνία αυτή, γιατί δεν πάτε πιο πέρα, γιατί δεν έχετε μια πραγματική ομοφωνία για να προστατεύσετε ας πούμε τα κράτη ας πούμε και απέναντι σε ξένους επενδυτές που έχουν τεράστια επιρροή. Ευχαριστώ. Θα είμαι όλοι σας στις παρεμβάσεις σας αναφερθήκατε στη λέξη κλειδί ασφάλεια. Ε, πώς μπορεί να ορίσει κανείς αυτό το πλαίσιο, αυτό το, τον όρο, αυτή την έννοια της ασφάλειας. Υπάρχει δηλαδή και μια οικονομική χρειά εδώ, οπότε θα ήθελα να ακούσω από σας ε, πώς ορίζετε την ασφάλεια. Ε, και από εκεί και μετά. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Ζαντόμολης τώρα, Άκουσα ε, την ίδια παρέμβαση που έκανε και σε ένα άλλο φόρουμ ε, σήμερα. Και ε, θα πρέπει να πω ότι εκείνο που δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ακριβώς ένας τέτοιος κίνδυνος όπως αυτός προέκυψε με την επένδυση στο λιμάνι του Πειραιά. Και σας ζητώ συγγνώμη εκ των προτείνων, αλλά έχω μια πτήση την οποία θα πρέπει να πάρω και θα αποχωρήσω κάποιος. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ πολύ Επίτροπε για την ε, παρέμβασή σας και ευχαριστώ και όλους τους ε, ε, ομιλητέ. Εγώ πιστεύω πως είναι ένα καλό έγγραφο, μια καλή αρχή. Καταρχάς έπρεπε να μπει αυτό το θέμα στη μερίσια διάταξη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει ένα μηχανισμό που θα ρυθμίζει τι ξένε άμεσε επενδύσει για την ασφάλειά μας και όχι μόνο για την ασφάλειά μας σε θέματα εθνικής άμυνας αλλά και για ό,τι αφορά τις απειλές σε τεχνολογικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια, υποβάλω μια ερώτηση στην ε, εκπρόσωπο ε, της Λετωνίας. Εσείς ε, είπατε ότι αυτή η οδηγία σας ανησυχεί μήπως δεν συμβαδίζει με την καλύτερη νομοθεσία. Και εγώ ρωτώ ως προς τι, γιατί ο ρόλος ε, της πρότασης αυτής είναι ε, μια στενότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κρατημέλη. Αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκεται και ε, θεσπίζει και ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Από πού εσείς λέτε ότι είναι κατά της καλύτερης νομοθεσίας εφόσον αυτή είναι η αρχή. Και άλλη μια ερώτηση για τον εκπρόσωπο τον είπα. Πώς μπορούμε εκ των προτέρων να καθορίσουμε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ή απειλή για το μίσο που είναι πραγματικά περίπλοκη. Πώς μετράτε τον αντίκτυπο, ποια μεθοδολογία έχετε, ποια κριτήρια χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε τον αντίκτυπο στην ασφάλεια. Ευχαριστώ κυρία Αντρικένα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε κάποιες ερωτήσεις προς την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ και πολύ μου αρέσανε οι παροιμίες σας, ε, οι κινέζικοι και οι ελληνικοί. Δεν πιστεύετε ότι μια ε, απόφαση ευρωπαϊκής διάστασης θα είναι εξαιρετικά μικρή και λιγοστή ε, σε σχέση με ε, σχετικούς μηχανισμούς που υπάρχουν ήδη σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων είπα η Ιαπωνία που προσπαθούν να περιορίσουν τις ξένες επενδύσεις γιατί όταν βλέπω την πρόταση όταν τη διαβάζω είναι μια συμβιβαστική μέση οδός. Το δεύτερο ερώτηση βεβαίως αυτό θα συζητηθεί στο Συμβούλιο και το πραγματικό, η πραγματική δοκιμασία θα είναι ε, στο Συμβούλιο του 2018 πρέπει να περάσει το κανονισμό με ειδική πλειοψηφία. Μπορεί δηλαδή, μάλλον αν λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει στις ε, νότιες ε, και χώρες της Ένωσης και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί τελικά αυτή η πρόταση να είτε να απορριφθεί τελείως είτε να χαλαρώσει πολύ. Και τελευταία μου ερώτηση αφορά τον ορισμό των στρατηγικών και σημασία τομέων. για τις νέες τεχνολογίες στους γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς όπως ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ την Επίτροπο και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές, λέει η κυρία Μόσκα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, την πρώτη ήδη την έθιξαν κάποιοι συνάδελφοι. πώ θα καταστήσουμε αποτελεσματικό αυτόν τον κανονισμό, δεδομένου ότι η Κομισιόν έχει μόνο το ρόλο εποπτείας ε, σε σχέση με τις γενικές δραστηριότητε που ήδη ασκούν τα κρατημέλη και πιο συγκεκριμένα, και αυτό το έθεξε ο εισηγητής, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ποιοτικέ πληροφορίε ώστε να τι ανταλλάξουμε. Για τη στιγμή που το θέμα αυτή τη πρόταση είναι να εντοπίζεται το ευρωπαϊκό συμφέρον, αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει ποιότη πληροφοριών που να ξεπερνά κατά κάποιο τρόπο τι διαφορές και τους διχασμούς ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δεδομένου ότι πρέπει να, να καταλάβουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ή θα πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι και για την προστασία ορισμένων επενδύσεων που είναι ε, ε, ε, επικίνδυνες ή διαφορετικά οι μεμονωμένες οι χώρες είναι πιο αδύναμες στο να υπερασπιστούν τις τους τομείς τους πιο ευαίσθητους. Και έπειτα κάτι ακόμα, συλλογή στοιχείων σε σχέση με το τι έγινε αφού έχει εισαχθεί ένας μηχανισμός ελέγχου σε κάποια κράτη, να δούμε δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο και τέλος τι σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε αυτή την πρόταση και την ε, συνέχιση και την, προ... την ε, πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων με την Κίνα για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage κυρία Χέρς, τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο ερώτημά μου το απευθύνω προς την Επίτροπο. Ε, αυτή την περίοδο γνωρίζω πως η Επιτροπή συγκεντρώνει τα μοντέλα που ισχύουν στα διαφορετικά κράτη-μέλη για να ε, γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει τελικά. Ε, αποκρισταλώνεται σιγά σιγά κάποια βέλτιστη πρακτική στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή διαπιστώνεται ότι το ένα ή το άλλο κράτος μέλος πραγματικά έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό σύστημα, ένα ικανοποιητικό μοντέλο. Ή αν όχι δεν έχετε δηλαδή ακόμα ολοκληρώσει αυτή την αξιολόγηση, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Δεύτερο ερώτημα, αυτό το απευθύνω στον ε, Αμερικανό φίλο μας, τον κύριο Μύρη. Ποια είναι η σύνθεση αυτής της Επιτροπής ε, CFIUS, γιατί αναφερθήκατε στο γεγονός ότι εδώ λαμβάνονται υπόψη και βέβαια ε, ζητήματα εθνική ασφάλειας, άρα έχετε εκπροσώπους από τους διάφορους κλάδου, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα τη ασφάλεια, αλλά ειδικότερα στον ψηφιακό τομέα και στην ψηφιοποίηση, θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη του και τα όσα ενδέχεται να ε, παίξουν ρόλο στο μέλλον. Δηλαδή μια επιχείρηση τη σήμερα ημέρα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά σε πέντε έτη από τώρα να εξελιχθεί σε ένα big player, δηλαδή ένα σημαντικό παίκτη εντό εισαγωγικών στην ε, αγορά. Οπότε ε, ποια είναι η σύνθεση αυτής της Επιτροπής. Συμμετέχουν εκεί μέλη τα οποία λαμβάνουν ε, υπόψη ε, συγκεκριμένε ε, διαστάσεις, για παράδειγμα την επένδυση συγκεκριμένων κονδυλίων σε ερευνητικού σκοπούς και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας και να σας πω πως πιστεύω μεγάλη είναι η σημασία της ύπαρξης ενός τέτοιου συστήματος και κυρίως το να έχουμε μια ευρωπαϊκή σκοπιά. Εγώ θα ήθελα να έχω πληροφορίες για το κατά πόσο υπάρχει μια αξιολόγηση ήδη από ευρωπαϊκή σκοπιά για τα όσα δηλαδή έχουν ε, ήδη φτιάξει τα διάφορα κράτη-μέλη. Είπατε, καμιά δεκαριά πως έχουν ε, μηχανισμούς ελέγχου. Πρέπει να σχηματίζονται κάποιες στάσεις ε, με θέληση ορισμένα κράτη να δεχτούν επενδύσεις για ορισμένους τομείς. Ξέρουμε κάτι περισσότερο για τις στρατηγικές αυτών των χωρών. Υπάρχουν κάποιες στάσεις γενικές που θα μας επιτρέψουν να προσαρμόσουμε τα κείμενά μας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο τον συνεισηγητή από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την ΟΚΕ, τον κύριο Μπάμλε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθετηθώ εδώ εκ μέρους ε, της ΕΟΚΕ αλλά και εκ μέρους ε, της ε, Επιτροπής των Περιφερειών βέβαια ασχολούμαστε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο με αυτό το ζήτημα και σα ε, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και επίση λοιπόν θεωρούμε πω ε, οι ξένε επενδύσει είναι σημαντικέ ε, για την ανάπτυξη και την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασία. και κατά συνέπεια σε γενικέ γραμμέ, επί της αρχής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στι ξένε επενδύσει από τρίτε χώρε. Ωστόσο αντιλαμβανόμαστε και εμεί του κινδύνου που μπορούν να προκύψουν και κατά συνέπεια είμαστε κι εμεί υπέρ τη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου screening των επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρία ζητήματα. Καταρχήν στο ζήτημα της αρμοδιότητας των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σημείο πεδίο εφαρμογή, αν θέλετε, ενό τέτοιου μηχανισμού, δηλαδή σε τι είδου επενδύσει και σε ποιου κλάδου θα μπορεί να εφαρμόζεται αυτό ο μηχανισμό ελέγχου. Και τρίτο, πώ θα διαμορφωθεί αυτό ο μηχανισμό με τρόπο που να μην αποτελέσει τροχοπέδι για επενδύσεις οι οποίες ε, συμβάλλουν στην ε, αύξηση της ευημερία και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επειδή τώρα έχει γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση σε ό,τι αφορά τη ΣΕΤΑ και άλλε συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου, νομίζω πως ε, μετά και από την ε, νομοδότηση του ε, Δικαστηρίου της Ένωσης σε σχέση με τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει εδώ αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τρίτων χωρών στα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρώ πω υπάρχει εδώ ζήτημα αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια το επιχείρημα ε, τη ε, που έχουν αναφέρει κάποιοι συνάδελφοι δεν ισχύει ε, σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, ακούσαμε ε, βέβαια και κάποια, για κάποια συστήματα όπω αυτό στη Γαλλία, τα οποία πράγματι λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα τη έννοια ε, τη δημόσια ασφάλεια ε, και τάξη, νομίζω πω ναι, πρόκειται για ζήτημα εθνική αρμοδιότητα και κατά συνέπεια εάν θέλουμε κανονισμό θα πρέπει να οριστεί επακριβώς το τι εννοούμε με αυτήν την εθνική ασφάλεια και τάξη έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί. Πάντως θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος ευρωπαϊκός ε, μηχανισμός, ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά κρίσιμες ε, υποδομές ίδρυυση, ηλεκτροδότηση και ούτω καθεξής. Και από εκεί και μετά, όταν έχουμε επενδυτές από κρατικά ελεγχόμενες ή κρατικές επιχειρήσεις, εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικό μηχανισμός, μια ειδική διαδικασία ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι τεχνολογίες κλειδιά δεν περνούν στα χέρια άλλων χωρών χωρίς τουλάχιστον να έχει γίνει η απαραίτητη επένδυση, ο απαραίτητο δηλαδή ύψος. Νομίζω πως θα πρέπει ο μηχανισμός μας να κινηθεί με βάση τις γενικές γραμμές της Επιτροπής Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω Πρόεδρο. Έχετε δίκιο δικά σε αυτό το τελευταίο σημείο που, στο οποίο αναφερθήκατε. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν προ την Επίτροπο και στου εμπειρογνώμονε. Ε, σε Σίλβια, πρώτα έχει εσύ το λόγο. Ε, οι ερωτήσει σα δείχνουν πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχετε για αυτά τα θέματα. Όπω είπαν και οι Αμερικανοί φίλοι μα, στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70. Δεν είναι κάτι που αναπτύσσεται μία νυχτή είσε σε μερικές εβδομάδες θα χρειαστεί χρόνος. Υπάρχει μια ομάδα συντονισμού των κρατών μελών που συνέρχεται, θα συνέλθει το Μάρτιο για να συζητήσει για πρώτη φορά το θέμα αυτό. Η Κομισιόν ετοιμάζει μια έκθεση για τις ε, άμεσες ξένες επενδύσεις που θα παρουσιαστεί στα... αργότερα μέσα στο 2018. Ήταν δύσκολο να λάβουμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη ε, αν μπορείτε να κάνετε κάτι στις χώρες σας για να πιέσετε ούτως ώστε να μας δοθούν πληροφορίες, καλό θα ήταν. Γιατί πριν ε, κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να έχουμε την πλήρη εικόνα, όλα τα στοιχεία. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας δώσουν πληροφορίες. Και μερικά δεν επιθυμούν να μας τις δώσουν. Έχουμε λίγα παραδείγματα από αυτές τις 12 χώρες που έχουν ε, νομοθεσία για τον έλεγχο, αλλά μοιάζει να μην έχει χρησιμοποιηθεί πολύ συχνά σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει, ε, επιμακρών μάλιστα, αλλά μόνο πρόσφατα άρχισαν να κάνουν μια πολιτική συζήτηση γύρω από το θέμα, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Είναι σημαντικό αλλά ευαίσθητο θέμα. Έχει συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπάρχουν στρατόπεδα στο Συμβούλιο. Ε, προσπαθούμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσουμε να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτού που δεν θέλουν τίποτα σε κάποιου, και σε κάποιου που θέλουν ακόμα κάτι πιο φιλόδοξο. Αυτό που είδαμε από την υποβολή, από την στιγμή που η πρόταση, υποβολήθηκε η πρόταση τέλη καλοκαιριού ότι αυξήθηκε η δραστηριότητα ε, στις διάφορες χώρες. Σεμινάρια, δραστηριότητες, συμμετείχαμε κι εμείς για να μιλήσουμε και να ακούσουμε κιόλα. Και η συζήτηση είναι όλο και πιο έντονη. Ακόμα και στις χώρες εκείνες που είναι πιο απρόθυμες ε, που είναι πιο, υπάρχει μεγαλύτερο σκεπτικισμό. Ε, όλοι να γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα από την νομοθεσία και το αν θα υπάρξει νομοθεσία, πρέπει να το συζητήσουμε τουλάχιστον το θέμα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στι διάφορε χώρε. Τώρα, είναι αργά, μήπω, ίσω. Ε, Εμεί ετοιμάσαμε την έκθεση σε χρόνο ρεκόρ και θα την παρουσιάσουμε μέχρι τα τέλη του 2018. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει το να αρχίσει τουλάχιστον η συζήτηση ε, μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν σημεία επαφή, ούτως ώστε άτυπα τουλάχιστον να αρχίσει συνεργασία. Στην πρόταση της Κομισιόν ορίζουμε τις, ε, το, το κρίτικο στρατηγικό συμφέρον, ε, τις κρίσιμες υποδομές, ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού, ε, ορισμένες χώρες έχουν ευρύτερο ορισμό των κρίσιμων υποδομών. Ε, εμείς θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε φυσικά αυτό τα κρατημέλη. Τι σημαίνει αυτή η όρη. Φυσικά αυτό είναι ουδέτερο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες χώρες. Υπάρχουν ε, το, ο Γαλιλαίος και κάποια, ε, κάποιες άλλες υποδομές που είναι κρίσιμες ε, για την Ευρώπη, επενδύουμε πολλά λεφτά και είναι λογικό η Κομισιόν να υπαγρυπνά για αυτές τις επενδύσεις. Τώρα, το αν θα υπάρξουν και άλλες εταιρείε ή επιχειρήσεις, αυτό καλύπτεται πλήρως από τη νομική βάση που προτείνουμε. Ε, το ίδιο που χρησιμοποιείται και για τα, τον εξοπλισμό διτής χρήσης ή τα αγαθά της χρήσης. Για την Κίνα τώρα. Ε, διαπραγματευόμαστε και, συζητόμαστε, και συζητάμε με την Κίνα για μια επενδυτική συμφωνία εδώ και καιρό. Και προσπαθούμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ισοτιμία με την Κίνα. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσουν οι Κινέζοι στην Ευρώπη από το αντίθετο, να επενδύσουμε εμεί στην Κίνα. Συζητάμε αυτά τα θέματα. Δεν προχωρούμε με το ρυθμό που θα θέλαμε. Δυστυχώ, θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα με του Κινέζους ομολογού μα, αλλά αυτό το θέμα ε, που συζητάμε σήμερα δεν έχει συζητηθεί με την Κίνα. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι, είμαστε στην αρχή του εγχειρήματο. Το πιο βασικό είναι να ξεκινήσει η συζήτηση, να συνεχιστεί η συζήτηση και να συλλέξουμε όσο να τον περισσότερες πληροφορίες, να αξιολογήσουμε ό,τι μπορούμε να αξιολογήσουμε και να επανέλθουμε με την ε, έκθεση και ελπίζουμε οι συζητήσεις να συνεχίσουν ε, να λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο. Ξέρω που, θα, που μπλοκάρει το πράγμα, που λύγει το πράγμα, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη ότι θα προχωρήσει. Και τώρα, ε, με αντίστροφη σειρά, οι ομιλητές του πάνελ να απαντήσουν. Ο κύριος Χιγκέ θα απαντήσει πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου κάναν ε, ερωτήσεις για το εύρος του μηχανισμού. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία. Δύο άτομα εργάζονται ε, με πλήρη απασχόληση και υπάρχει ένας θυματάρχης που είναι υπεύθυνο. Από την εμπειρία που έχουμε και ε, λόγω της ύπαρξης του ίδιου του μηχανισμού ε, υπάρχει ε, σίγουρα ένας αποτρεπτικός χαρακτήρας για κάποιες ξένες επενδύσεις. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχει. Η διαδικασία είναι δύο μήνες από τη στιγμή που θα λάβουμε τον πλήρη φάκελο. Θα πρέπει δηλαδή να, έχει, να είναι πλούσιο φάκελο, να έχει περισσότερε δυνατέ πληροφορίε και έχει, υπάρχει ένα χρόνο δύο μήνε που τρέχει. Δεν, μας, σταματάμε μόνο στι πληροφορίε που μα δίνει ο επενδυτή. Συνεργαζόμαστε με τι διάφορε υπηρεσίε και φορεί, καθώ και με υπηρεσίε μα στο εξωτερικό. Παραδείγματο χάρη, ε, ρωτάμε για τη φήμη του ΑΒ επενδυτή, παραδείγματο χάρη. Ε, το σύνολο λοιπόν των υπηρεσιών μας το Υπουργείο Άμυνας, ας πούμε, και όλες οι εξαρτώμενες υπηρεσίες και φορείς συνεισφέρουν τόσο ώστε να επιταχύνουν την ε, διεκπαιρέωση του φακέλου. Τώρα, για τον ορισμό της ε, ασφάλειας. Μου φέρνει στο μυαλό τον ορισμό που έδινε ο μεγάλος νομικός, ε, αμερικανός νομικός για την πορνογραφία. Έχουμε μία, ένα ορισμό εξελικτικό για την ασφάλεια. Πριν από 150 χρόνια, ας πούμε, είχαμε ένα μηχανισμό που κάλυπτε, ας πούμε, την κτηνοτροφία ύπων, Φερρυπίν. Αυτό ήτανε. Τώρα σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, ε, ανατομέα κτλ. Και, και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη εμπεριέχεται ε, στον ορισμό αυτό. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη πανελίστρια. Θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Ροντρίγκες. Ίσως ε, να υπήρξε μια παρανόηση το ανώσαρτα. αυτά. Είπα ότι λόγω της ε, διοργανικής ε, συμφωνίας κάθε νέα νομοθετική πρόταση θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από αξιολόγηση αντικτύπου. Κάτι που δεν συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά δηλαδή δεν συνάδει με τα όσα συμφωνήθηκαν στο επίπεδο της διοργανικής συμφωνίας. Ε, και ότι με αυτόν τον τρόπο δηλαδή η Επιτροπή δεν συμμορφώθηκε με αυτή τη διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Και εμεί ε, από την πλευρά του Συμβουλίου ε, ασχοληθήκαμε για τρεις, ε, σε τρει συνεδριάσει τη ομάδα εργασία με αυτό το ζήτημα τη αξιολόγηση αντικτύπου. Και ζητήσαμε ακριβώ ακόμα και εκ των υστέρων από την Επιτροπή μια τέτοια αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, αν όχι πλήρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βασικότερα στοιχεία. τώρα, τώρα. σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό του ελέγχου των επενδύσεων. Ε, σίγουρα πως ε, ε, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της ασφάλειας για όλους μας, γιατί ήδη αυξάνονται οι σχετικές επενδύσεις με μέτρους ρυθμούς Και βέβαια ε, αυτή η ε, ε, ελκυστικότητα αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ξένες επενδύσεις είναι, έχει ακόμα πιο σημαντικές επιπτώσεις για τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ένωσης. Ακόμα δηλαδή και με αυτήν την αύξηση του 3% εμεί παραμένουμε φιλόδοξοι να φτάσουμε στο 5% αλλά βέβαια θα δούμε ποιο θα είναι ο αντίκτυπο ε, του κανονισμού σε αυτές τις ε, ξένε επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως ε, ό,τι και αν προβλέψουμε στο πλαίσιο δηλαδή, του μελλοντικού μηχανισμού θα πρέπει να παραμείνουν οι δυνατότητες για επενδύσεις και στο μέλλον. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος έχει το λόγο. Ναι, τέθηκαν κάποια ερωτήματα ω προ το πώ προβαίνουμε στι αξιολογήσει μα και πώ ορίζουμε την εθνική ασφάλεια, το national security. Η ασφάλεια δεν ορίζεται στη δική μα εντολή, οπότε την ορίζουμε ανάλογα δηλαδή με τι εξελίξει, ανάλογα με, τις, με τα διάφορα τροτά σημεία μα. Ο ορισμός δηλαδή είναι αρκετά ευρύς έτσι ώστε αυτές, αυτή την περίοδο να περιλαμβάνει ζητήματα για παράδειγμα υποδομής τηλεπικοινωνιών ή άλλων υποδομών όπου η κατασκευή ή η καταστροφή τέτοια υποδομή θα μπορούσε να είχε ε, σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και στην ανθρώπινη ζωή. Επίση, ε, ε, περιλαμβάνει και ζητήματα ευαίσθητων πληροφοριών πληροφορίες οι οποίες ε, εάν διαρρεύσουν μπορούν για παράδειγμα να ε, έχουν ανετικό αντίκτυπο για τις ενόπλες ε, δυνάμεις μας γενικότερα για το προσωπικό μας. Είναι λοιπόν ευρύ ορισμό της εθνικής ασφάλειας και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό συμφέρον των ΗΠΑ. οι επιχειρήσεις ε, δηλαδή αποφασίζουν φυσικά στο πλαίσιο μιας επένδυσης κατά πόσο η εν λέγω επένδυση είναι προς το συμφέρον τους ή όχι. Τώρα, ως προς το πώς ε, αποφασίζουμε, ε, ως προς το κατά πόσο μια επένδυση αφορά ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή όχι, πράγματι οι επενδύσεις γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκες τα τελευταία χρόνια και λόγω της αυξημένης περιπλοκότητας των συναλλαγών, αλλά και επειδή ε, κάποιες από τις τεχνολογίες ε, που ισχύουν ε, και υπάρχουν σήμερα είχαν αναπτυχθεί κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς πριν από 20 χρόνια. Και οι μελλοντικές τεχνολογίες θα προβλέπουν και θα περιλαμβάνουν τέτοιου είδους ικανότητα αμυντική και ικανότητες σε σχέση με την ηθική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν αυτό καθιστά πιο περίπλοκο το έργο μας, δηλαδή του να να διαπιστώσουμε ποιε τεχνολογίε εκείνε που έχουν και μια τέτοια διάσταση που αφορά στην εθνική ασφάλεια. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε σε αυτέ τι περιπτώσει είναι να έχουμε πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη από όλου του τομεί τη κυβέρνησή μα. Έχουμε καταρχήν ε, το Υπουργείο Οικονομικών ε, που ασχολείται ακριβώ με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε, χρηματοδότηση τρομοκρατία και άλλες δραστηριότητε οικονομικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικού. Από εκεί και μετά έχουμε το Υπουργείο Άμυνα και όλου του τεχνικού και όλου του ειδικού σε σχέση με τι σχετικέ ικανότητε. Έχουμε μετά το Υπουργείο Ενέργεια ε, με την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη όχι μόνο σε ό,τι αφορά ε, τι υποδομέ ενέργεια αλλά και σε ό,τι αφορά ε, ζητήματα πυρηνική ενέργεια αλλά και ζητήματα ημεαγωγών. Μετά έχουμε εκείνο του Κογκρέσου όπου υπάρχουν μια σειρά από πολιτικοί μηχανικοί που ασχολούνται με κάθε είδου τεχνολογία ασφαλεία από εκεί και μετά ε, και το State Department αλλά και εκπροσώπους από τον εμπορικό ε, τομέα έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι όταν εξετάζουμε μια συναλλαγή εντοπίζουμε πράγματι όλα τα ζητήματα εθνική ασφάλεια και ταυτόχρονα βέβαια παραμένουμε εντό τη εντολή μα, δηλαδή να ασχολούμαστε αμυγό με ακριβώ ζητήματα εθνική ασφάλεια. Προσπαθούμε λοιπόν να συγκεντρώνουμε την απαραίτητη προγνωμοσύνη από όλα τα τμήματα τη κυβέρνηση και να γίνεται η κατάλληλη εξέταση από το αρμόδιο ακριβώ ε, τμήμα. Σε τελική ανάλυση βέβαια κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίζει σε ποιο βαθμό θέλει να εξετάσει περισσότερο ή λιγότερο διεξοδικά την εκάστοτε επένδυση. ειδικότερες, ειδικότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που εξετάζουμε ε, των ε, αμερικανικών επιχειρήσεων αυτή την περίοδο, σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερη, καλύτερη εξέταση. Ε, και επειδή προβλέπεται προθεσμία 25 ημερών, ε, προφανώς η λόγω διαδικασία είναι ταχύτατη ε, μέσα στην κυβέρνησή μας, αλλά ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία, ότι δηλαδή γίνεται ο κατάλληλος διεξοδικός έλεγχος, αλλά από την άλλη πλευρά δίνεται και ο κατάλληλος χρόνος στα διαφορετικά τμήματα έτσι ώστε να προβούν στην απαραίτητη εξέταση, στην απαραίτητη αξιολόγηση. Τώρα, τέθηκαν κάποια ερωτήματα ω προ τη συνεργασία μα ε, με άλλε χώρε. Ναι, εξετάζουμε τα όσα συμβαίνουν τόσο εντό τη επικράτειά μα όσο και εκτό αυτή, έτσι ώστε να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε μια κοινή κατανόηση τη ασφάλεια και να αναγνωρίσουμε προβλήματα που ε, ανακύπτουν, ακόμα και αν δεν εμπίπτουν αμυγό στην δική μα ε, δικαιοδοσία. Πάντω, η προστασία των ικανοτήτων και ε, τεχνολογιών εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει κέρια σημασία και για την προστασία των δικών μας αντίστοιχων συμφερόντων στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, και ακριβώς η, πρόσφατη θέτηση σχετικής νομοθεσίας στις Ηνωμένε Πολιτείε λαμβάνει αυτή τη διάσταση υπόψη γιατί Ε, προβλέπει ότι ε, δεν ε, εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή τη εξέταση των επενδύσεων επενδύσει που λαμβάνουν χώρα σε χώρες οι οποίε ακριβώ διαθέτουν ένα αντίστοιχο μηχανισμό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε αυτέ τι περιπτώσει βασιζόμαστε στον μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων αυτών των άλλων χώρων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, τον κύριο Αμέρη. Λάβαμε εδώ λοιπόν μια γενική επισκόπηση των διαφορετικών ζητημάτων και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ το οποίο εξετάζει πιο συγκεκριμένα την πρακτική εφαρμογή του, του ελέγχου των επενδύσεων και έχουμε και εδώ μαζί μας ε, κάποιους συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες ε, για πέντε λεπτά ο καθένας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΩΣΑ, έχουμε δύο εκπροσώπους, οπότε θα λάβουν συνολικά 8 λεπτά. Ε, ο ΩΣΑ μια ενδιαφέρουσα μελέτη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 ε, αφοσιωμένη σε ένα ανοιχτό επενδυτικό κλίμα, δηλαδή υπάρχει αναγνώριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη μας και είμαστε 35 τον αριθμό, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ένωσης, που είναι μέλη του ΩΣΑ. Αναγνωρίζουν λοιπόν ότι είναι προς το συμφέρον των χωρών να διατηρούν ένα, μια ανοιχτή επενδυτική πολιτική. Και θεωρούμε τις επενδύσεις ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, για αυξημένη ευημερία και ε, ως μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ταυτόχρονα όμως ο ΣΑ αναγνωρίζει ότι οι χώρες μέλη έχουν το δικαίωμα να προστατέψουν ε, την εθνική τους ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, το δημόσιο συμφέρον απέναντι στις, ε, ερχόμενες, στις εισερχόμενες επενδύσεις. Άρα μπορούν να ελέγχουν, να περιορίζουν τις ξένες επενδύσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται και είναι ένας από τους κύριους κανόνες του ΣΑ που έχει αναφερθεί και από τον πρόεδρο του CFIUS. Ότι αυτό πρέπει να γίνεται επί τη βάση συγκεκριμένων προτύπων, πρώτον διαφάνεια, δεύτερον προβλεψιμότητα, τρίτον αναλογικότητα και τέλος λογοδοσία. Επί τη βάση λοιπόν των ε, μέσων που έχει στη διάθεση το ΩΣΑ, η γραμματεία που εμείς αντιπροσωπεύουμε, η γραμματεία της Επιτροπής Επενδύσεων, ε, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα και αυτό οδήγησε, όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, στην εκπόνηση μιας έκθεσης που δημοσιεύθηκε πριν από 1,5 χρόνο και που είναι μια έρευνα όχι μόνο για τις εξελίξεις πολιτικών στις, στον τομέα αυτών ή στις 35 χώρες τόσο, αλλά το ξεπερνάμε και αυτό, γιατί έχουμε ένα φόρουμ στο Παρίσι όπου συγκεντρώνουμε πάνω από 55 χώρες, που είναι και χώρες όπως η Κίνα, η Ιδονησία και άλλες, και εκεί συζητάμε τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Δεν θα σας παρουσιάσω τα κεντρικά απορίσματα αυτής της έρευνας, διότι ο συνάδελφος Γιωακήμ θα το κάνει και θα δείτε ότι η έκθεση που έχουμε δημοσιεύσει μπορεί να απαντήσει κάποια από τα ερωτήματα που ήδη εγερθήκαν ε, ε, στο πρώτο τμήμα της συζήτησης. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αυξανόμενη τάση για μηχανισμούς ελέγχου με επί τη βάση της εθνικής ασφάλειας. για τις χώρες μέλη του ΩΣΑ πάντοτε μιλάω. Μισές εξ αυτών έχουν ήδη θεσπίσει τέτοιους μηχανισμούς. Και ίσως αυτό που είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς είναι ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν θεσπιστεί, έχουν ενισχυθεί στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Και έχουμε και πρόσφατες εξελίξεις από τη Λετωνία. Η Γερμανία έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις πριν λίγους μήνες. Και άλλες χώρες σκέφτονται είτε να ενισχύσουν αυτούς τους μηχανισμούς που ήδη έχουν, είτε να συστήσουν νέους. Ε, το θέμα αποκτά σημασία δηλαδή όσον αφορά τα θέματα εθνικής ασφάλειας και με χαρά συμβάλλουμε σε αυτήν τη συζήτηση για να σας φέρουμε, δώσουμε τα βασικά πορίσματα αυτής της μελέτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια για τη δουλειά μας. Έχουμε φέρει ε, τη μελέτη μας, έχουμε φέρει κάποια αντίτυπα, είναι στην έξοδο. Να συνοψίσω τα κύρια πορίσματα. Έχουμε εξετάσει 60 χώρες περίπου και από τις 60 περίπου το 1 τρίτο έχουν ε, ε, εισάγει πολιτικές για να αποτρέψουν ε, θέματα εθνικής, προβλήματα μάλλον εθνικής ασφάλειας. Από τις χώρες που έχουν εγκαταστήσει τέτοιες πολιτικές έχουν διαφορετικές πολιτικές η καθεμία. Καμία δεν συμπίπτει με την άλλη. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι σε θετική ε, θέση. Ε, αν δείτε την ελληνική και την κινέζικη παροιμία, γιατί έχετε πολλές ε, περιπτώσεις στις γειτονικές σας χώρες για να μελετήσετε τι λειτουργεί καλύτερα. Τώρα, να σας πω ποια είναι η ποικιλομορφία όλων αυτών. Έχουμε να διακρίνουμε τρεις ομάδες. Οι χώρες που δεν έχουν τίποτα, οι χώρες που είναι στην άλλη άκρη του φάσματος όπου δηλαδή έχουν, έχουν πάρει πολύ σοβαρά υπόψη την υπόθεση αυτή και ακούσαμε ένα παράδειγμα και στη μέση υπάρχουν διάφορες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που ε, έχουν προβλέψει και επιτρέπουν την ε, απαγόρευση κάποιων επενδύσεων. Τώρα, αυτό που διακρίνει είναι ο προπολογισμό, το θεσμική μορφή και οι δυνατότητες που έχουν προϋπολογισμός. Η ΕΠΑ δαπανούν αρκετά εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για το μηχανισμό ελέγχου. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ε, δαπανά αρκετές χιλιάδες ευρώ για αυτό το μηχανισμό. Ε, χίλιες φορές παραπάνω δηλαδή δαπανά μια χώρα σε σχέση με μια άλλη μεγάλη οικονομία της Ένωσης. Ε, θεσμική μορφή. Κάποιες χώρες εργάζονται με την κοινωνία με, την, με τον τομέα μάλλον των πληθυμιστικών πληροφοριών και προσπαθούν να συνεργαστούν και με άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν ακόμα διαλέξει μια μέση εδώ και άρα οι δυνατότητες αυτών των μοντέλων είναι είτε να ανοιχνεύσουν αυτό μάλλον που καταφέρνει ο μηχανισμός των ΙΠΑ ε, και άλλοι μηχανισμοί όπου κοστίζουν εκατομμύρια και άλλοι μηχανισμοί μπορούν να εμποδίσουν σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, γνωστό πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούν να εντοπίσουν πρόβλημα το οποίο να μην διαφαίνεται ήδη με κάποιο τρόπο. Το θέμα δεν είναι λοιπόν αν θες να ασκήσεις κάποια πολιτική, αλλά το ποια πολιτική είναι η καλή. Και αυτή είναι μια ερώτηση που μου έχει ήδη Το κράτος δικαίου απαιτεί να υπάρχουν προβλέψιμοι κανόνες σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο γνωστό πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό συνάδει προς ε, την ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων ενό θεσμού που θα λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με προβλέψιμους, όπως είπαμε, κανόνες ή νόμους. Επόμενο ερώτημα είναι θες να ταπανίσεις εκατομμύρια ή χιλιάδες. Θες δηλαδή να ξεπεράσεις τη δυνατότητα απλής ενέργειας όταν γνωρίζεις ήδη κάτι ή θες να μπορείς και να προβλέψεις, να ανοιχνεύσεις. Δεν γνωρίζουμε δυστυχώς και κανείς δεν γνωρίζει μάλλον γιατί οι βασικοί δείκτες απόδοσης δεν υπάρχουν ακόμα δεν, και μάλλον δεν θα υπάρξουν. Πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, απετράπησαν οι κίνδυνοι στον κόσμο κάπου με βάση κάποια από αυτά τα συστήματα. Δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν πλέον πληροφορίες. Έπειτα, ποιοι κίνδυνοι δεν αποφεύθηκαν παρότι υπήρχε ε, κάποιος μηχανισμός ελέγχου. Η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών δεν είναι γνωστή. Και έπειτα, άλλη ερώτηση που ε, απασχολεί κάποιες χώρες. Ποιες ε, επενδύσεις ε, έχουν αποτραπεί ενώ θα ήταν επιθυμητές και μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός ελέγχου. Ξέρουμε πως υπάρχουν κάποιες ε, απαγορεύσεις, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, άρα και κάποιο κόστος και πιστεύουμε πως η δυνατότητα αποτροπής, μάλλον η αποτροπή λόγω της ύπαρξης μηχανισμού ελέγχου είναι σχετικά μικρή. Έπειτα η ελαστικότητα είναι περιορισμένη. Αν ας πούμε θέλει κανείς να αγοράσει έναν γερμανό κατασκευαστή ρομπότ, μόνο στη Γερμανία μπορεί να το αγοράσει. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους δυνατότητες θέλουμε να, να έχει αυτός ο μηχανισμός και τι προϋπολογισμό ε, θέλεις να ε, δαπανίσεις και έπειτα μπορείς να επιλέξεις από ε, τους διάφορους αυτούς μηχανισμούς που ήδη υπάρχουν μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι ε, πρόβλημα αυτό. Κώστα Καν, Διευθυντή Θεσμικών Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, εφεξή ΕΤΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, Πρόεδρε, για να σας δώσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για αυτό το σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γενικά θετικές, θετικές δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό ακριβώς και τις μετράμε τόσο πολύ. Ε, προσπαθούμε να δούμε τι κάνουμε για να τις προσελκύσουμε τις ξένες επενδύσεις. Η τράπεζα με περηφάνεια λέει ότι το 1 τρίτο των ομολόγων της τράπεζας αγοράζονται από επενδυτές ξένους, μη Ευρωπαίους και θεωρούμε ότι είναι σημάδι εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία και δέσμευση στην ε, ανάπτυξή της. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΤΕ ανήκει στα κράτη-μέλη και χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις, ε, άλλες και υλικές, για την υποστήριξη των θέσεων απασχόληση. Υποστηρίζουμε project που εφαρμόζουν τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και προωθούν τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα project υπόκεινται σε, στην αρχή τη δέουσα επιμέλεια. Όχι μόνο στα, σε ό,τι τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά πρότυπα, αλλά τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κρατικά κυβερνητικά δηλαδή, καθώς και την ε, συνεισφορά στις, ε, στην υλοποίηση των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος της τράπεζας ε, περιέχει μια αναθεώρηση της, του καθεστώτος ιδιοκτησίας του επενδυτή, ούτω ώστε να υπάρχει κίνδυνο, διαφθορά, ξεπλήματο χρήματο κτλ. Και έχουμε και μια διαφθορά, διαδικασία του άρθρου 19, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε project, δηλαδή κάθε έργο το οποίο εξετάζει το Συμβούλιο μας θα πρέπει να έχει τη γραπτή έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Η Κομισιόν επίσης εκπροσωπείται καθώς και τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται ε, μέσω της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εκφίν και της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει μια ευθυγράμμιση λοιπόν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει και το σχέδιο καονισμού, το έχουμε λάβει υπόψη και πρέπει να υπάρχει ε, ισορροπία ανάμεσα στην, ε, στο να υπάρχει μια ανοιχτή ευρωπαϊκή οικονομία στις ξένες επενδύσεις αλλά και προστασία των βασικών ε, συμφερόντων των κρατών μελών. Οι τομεί που ανέφερε η Κομισιόν, οι κρίσιμες υποδομές Φερρυπίν και η κρίσιμη τεχνολογία είναι τομεί που η ΕΤΕ ε, υποστηρίζει τις επενδύσεις. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ε, Καινοτομία είναι βασικό στόχος. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για το πώς σκοπεύουν να διενεργήσουν αυτόν τον έλεγχο για να καταλάβουμε το πώς θα εφαρμοστεί τελικά στην πράξη. Θέλουμε να πούμε ότι ο έλεγχος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει πολύ περίπλοκος, γιατί για να είμαστε ανταγωνιστικοί ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να κρατήσουμε και την νομική ασφάλεια για τους επενδυτές, ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν ένα σαφές πλαίσιο και να μην υπάρχουν ε, περιττές καθυστερήσεις στη διαδικασία ε, έγκρισης. Όταν ξεκίνησε το σχέδιο Juncker, ένα βασικό στοιχείο ήταν να μην υπάρχουν φραγμοί στις επενδύσεις. Εάν θέλουμε τέτοιον ευρωπαϊκό συντονισμό για τον έλεγχο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες ή ανεπιθύμητα εμπόδια στις επενδύσεις. Όταν μιλάμε για τους φραγμούς, μην ξεχνάμε και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες όταν προσπαθούν να επενδύσουν στο εξωτερικό. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την οικονομική διπλωματία και αναθεωρούμε και εξετάζουμε το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε την διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σεβασμό των κανόνων του ΠΟΕ. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος και θέλουμε η ε, ανοιχτή ευρωπαϊκή οικονομία να συνοδεύεται από ανοιχτές οικονομίες ε, στις χώρες εταίρους. Μια τελευταία παρατήρηση που δεν συνδέεται τόσο πολύ με τον έλεγχο των επενδύσεων, ε, αλλά στο πώς θα έχουμε και τα οικονομικά προϊόντα για να υποστηρίξουμε αυτούς τους στρατηγικούς τομείς. Έχουμε αναπτύξει καλά ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα για νεοφύης επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα όταν ε, γιγαντωθούν αυτές οι, επιχειρήσεις ε, και γίνουν στόχο στόχος επενδυτών ή μεταναστεύσουν ή μετεγκατασταθούν ας πούμε, στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, στι πιο κρίσιμες στιγμές ε, η Ευρώπη δεν είναι παρούσα και τελικά οι θέσει απασχόληση μετακινούνται και φεύγουν από την Ευρώπη. Ε, αυτό το φαινόμενο σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν δρέπει τους καρπούς ε, από το, τη γιγάντωση αυτών των ε, πιο καινοτόμων ας πούμε, νεοφιών ε, επιχειρήσεων που τελικά περνάνε σε άλλη φάση στο εξωτερικό κτλ. Ε, και εκεί ε, τις παίρνουν ε, ξένοι επενδυτές. Ε, Παραδείγματο χάρη η γερμανική εταιρεία Κούκα, εταιρεία ρομποτικής. Ε, πρέπει να δούμε αυτό το θέμα της φάσης ε, της ορίμασης του κεφαλαίου και να δούμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να καλύψουμε αυτά κενά, ούτως ώστε να δρέψουμε και εμείς τους καρπούς. Ίσως με την κεφαλαιακή ένωση της Ευρωπαϊκής, ε, με την ένωση των κεφαλαίων δηλαδή, θα πετύχουμε περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Από το Hudson Institute, ο Γιώνας Παραλουπλάς, να έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με κάλεσε σήμερα εδώ. Ε, και ε, ζητώ συγγνώμη εκ των πρώτων από τους διερμηνείς ε, γιατί είναι λίγο βραχνή η φωνή μου. Είχα ένα ακρολόγημα, κόρσα κάτι στο αεροπλάνο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτής Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, ξένων επενδύσεων, ειδικότερα από την Κίνα, ε, είναι κάτι που με έχει απασχολήσει για αρκετό καιρό. Είχα ε, συμμετάσχει στο σχετικό Think Tank, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τι Ξένε Σχέσει και ήμουν ένα από του συντάκτε σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά την αύξηση αυτών των κινέζικων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είχα ήδη από τότε προτείνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων και εδώ στη δική σας επιτροπή είχα αναφερθεί ε, στη σημασία του να υπάρξει ένας τέτοιος ε, μηχανισμός ε, και θεωρώ κατάλληλη χρονική συγκυρία ότι συζητείται τώρα αυτός ο μηχανισμός και ελπίζω να εφαρμοστεί στο εγγύ μέλλον. Ε, συμφωνώ με τα όσα είπε ο πρόεδρο ε, Γιούγκερ ότι δεν ε, είμαστε αφελεί ελευθερεμπορευόμενοι. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται στα στρατηγικά τη συμφέροντα και όταν υπάρχει η εξαγορά μια σημαντική επιχείρηση ή μια, μια σημαντική επένδυση από μια κρατική επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διαφάνεια και ο κατάλληλο έλεγχο. Και εδώ πέρα βέβαια αναφερόμαστε ειδικότερα στι κινέζικε επιχειρήσει, οι οποίε έχουν αυξηθεί σημαντικά με βάση δηλαδή μια έκθεση τη Rasmussen Global. Υπάρξει, έχει υπάρξει το 2016 αύξηση κατά 77% των κινέζικων επενδύσεων. Κυρίως αυτές ε, αφορούν ε, επενδύσεις ε, στις, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες και συνάδουμε τη την γενικότερη στρατηγική της Κίνας Made in China 2025 και δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα σε ό,τι αφορά τις κινέζικες επιχειρήσεις. Ε, και βέβαια, λαμβάνοντα υπόψη ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν είναι συμμαχό μα, ενέχεται από ένα πολιτικό κόμμα και είναι ε, μια ολοένα και ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, θα πρέπει να, να σκεφτούμε και τα ζητήματα που προκύπτουν σε επίπεδο ασφάλεια ε, και ειδικότερα μέσω τη εξαγορά που γίνεται με εξαγορέ και συγχωνεύσει. Γιατί βέβαια, εάν προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε εκ των υστέρων, θα βρεθούμε σε αντίστοιχη κατάσταση με αυτή τη υπερβολική, τη υπέρμετρη εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το φυσικό ρωσικό αέριο. Ε, ποια είναι λοιπόν τα κυριότερα επιχειρήματα υπέρ τη δημιουργία ενό τέτοιου μηχανισμού ελέγχου των επενδύσεων. Καταρχήν πρόκειται για σύνεση και όχι προστατευτισμό. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ευθυγραμμιστεί με τα όσα ε, κάνουν ήδη άλλες ε, χώρες ανά τον κόσμο. Δηλαδή η δημιουργία ενό τέτοιου μηχανισμού ελέγχου των επενδύσεων δεν συνιστά προστατευτισμό. Αποτελεί κοινή λογική και ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδά και η Ιαπωνία εφαρμόζουν τέτοιου είδου συστήματα, αλλά και η ίδια η Κίνα διαθέτει το δικό τη σύστημα ελέγχου των ξένων επενδύσεων. Ε, τώρα, καθώ εργάζομαι αυτή την περίοδο σε ένα αμερικανικό think tank, το Hudson Institute, παρακολουθώ την ε, συζήτηση που γίνεται εκεί και θα ήθελα να σα δώσω ε, ε, κάποια ε, παραδείγματα εδώ. Ο, ο κύριο Αεμίρ από την ε, Συμφίουσα αναφέρθηκε στο ποιο είναι το σκεπτικό και ε, θεωρούμε πως ε, αντίστοιχα με τη Συμφίουσα θα πρέπει να υπάρξουν τα, αντίστοιχα στοιχεία δηλαδή. Η πρόταση της Επιτροπής σε αυτή την περίοδο ουσιαστικά εμ, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προβλέπουν σωσιατικό έλεγχο χωρί να βρίσκεται κάτι πιο συγκεκριμένα. Εμεί ε, θεωρούμε πω ε, θα πρέπει να βασιστεί το νέο σύστημα στο Σεφυρίους που είναι και το πιο προχωρημένο πρότυπο τη σήμερα ημέρα. Ε, και από εκεί και μετά θα ήθελα να αναφερθώ στο πώ ε, ο έλεγχο των επενδύσεων θα μπορούσε να προωθήσει τις, ε, διαταδικό συντονισμό σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Υπήρξαν μια σειρά από πρόσφατε περιπτώσει. Για παράδειγμα, ε, πριν από την εξαγορά τη γερμανική Κούκα από την κινέζικη Μεντέα, η Κούκα έπρεπε να απαλλαγεί από τον κλάδο των Systems Aerospace, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη διαστημική έρευνα, μετά από σχετική έρευνα που έγινε από την CFUC. Για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα τη Extron, μια γερμανική που εξαγοράστηκε από κινέζικη, ε, υπήρξε εδώ μια σχετική εκτελεστική απόφαση του Προέδρου Ομπάμα το Δεκέμβριο του 2016 ε, καθώς υπήρξε μια σχετική εξέταση από την πλευρά τη ΣΥΦΙΟΥΣ και καθώ η Έξτον είχε και κάποιες θηγατρικές στι ΗΠΑ είχε δικαιοδοσία η ε, ΣΥΦΙΟΥΣ. Ε, τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 12 κράτη-μέλη ε, διαθέτουν ένα μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων. Ε, στην πρόσφατη τώρα Εθνική ε, Στρατηγική Ασφαλεία ε, των ΗΠΑ αναφέρεται ρητά και ανησυχία σε ό,τι αφορά τι κινέζικε επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται δηλαδή ότι εδραιώνεται στρατηγικά η στην Ευρώπη επενδύοντα σε ε, υποδομές και σε ευαίσθητες τεχνολογίες. Άρα λοιπόν η δημιουργία ενός ε, μηχανισμού ελέγχου των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε ακριβώς να ε, αποβεί προς όφελος και του συντονισμού ε, μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαϊκής Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνο μου, αλλά ήθελα να θίξω και τα γενικότερα ζητήματα τη ευθυγράμμιση των πολιτικών ΕΕ και Κίνα. Αλλά θα αναφερθώ μόνο σε αυτό λέγοντα ότι ε, πέραν του ίδιου του ελέγχου ε, των επενδύσεων και του σχετικού μηχανισμού υπάρχουν και ευρύτερα ζητήματα όπω αυτό τη αμοιβαιότητα ε, σε ό,τι αφορά ακριβώ τη δυνατότητα επενδύσεων. Αυτά από την πλευρά μου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η Λουίζα Σάντος τώρα, διευθύντρια για διεθνείς σχέσεις της Business Europe την οποία βέβαια γνωρίζω ήδη πολύ καλά. Λοιπόν, Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι στην Business Europe ακόμα είμαστε στην ε, οριστικοποίηση της θέσης μας όσον αφορά τις, ε, τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων, αλλά θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ιδέες και να θέσω και κάποιες ερωτήσεις, καθώς και να τονίσω κάποιες πτυχές που ανάλογα με την πρόταση το, την έκταση της πρότασης μπορεί να, να είναι τελικά θετικά στοιχεία ή και λιγότερο θετικά. Καταρχάς θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η πρόταση είναι ε, κατάλληλη. Όταν μιλάμε για επενδύσεις είναι σημαντικό να έχουμε μια γενική εικόνα και προοπτική για τις πολιτικές τις επενδυτικές στην Ένωση πριν αρχίσουμε να υιοθετούμε μέτρα για κάποιον τομέα. Ίσως για αυτό είναι ένας από τους λόγους ε, που θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια μελέτη αντικτύπου πριν την υποβολή της πρότασης, δηλαδή να δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους οι διάφορες προτάσεις. Οι άλλοι ομιλητές δε ε, επαναλαμβάνουν και επαναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά ότι θέλουμε η Ευρώπη να μείνει ανοιχτή στις επενδύσεις και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο ανταγωνισμός των, για τις επενδύσεις αυξάνεται, όλο είναι και περισσότερες χώρες ασκούν πολύ επιθετικές πολιτικές για να προωθήσουν ε, και να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις ε, με διάφορα μέσα, όπως και με τη φορολογία. Μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας της ΣΥΠΑ, που σίγουρα θα προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε λοιπόν αυτή την πτυχή. Και είναι σημαντικό <coughs> να το έχουμε υπόψη μας ε, και έπειτα χωρίς να θέλουμε να στιγματίσουμε κάποια χώρα και δεν θέλω να στιγματίσω την Κίνα εδώ, αλλά γιατί είναι σαφές και με άλλες χώρες ότι θεωρούμαστε και νομίζω πως όλοι εδώ θα συμφωνήσουν ότι η Ευρώπη είναι πολύ ανοιχτή αγορά όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις και αυτό, πράγμα που δεν ισχύει σε όλες τις χώρες. Τώρα, ο έλεγχος είναι ένας τρόπος εξορρόπησης κατάστασης, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ξέρουμε πως έχουμε περιορισμούς για το πεδίο εφαρμογής, για, δηλαδή μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί καταρχάς υπάρχει το θέμα εθνικής μονοδιότητας, υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας, αλλά υπάρχει και το θέμα του σεβασμού των διεθνών μας δεσμεύσεων σε διάφορα φόρα όπως ο ΣΑΙ ο Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ακριβώς τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτή την πρόταση. Είναι η βελτίωση της πρόσβασης μας στις αγορές, είναι το να αυξήσουμε τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και εδώ βεβαίως πολλά μπορούν να γίνουν. Έχουμε σήμερα διάφορα συστήματα, όπως είπαν πολλοί έχουμε λιγότερες χώρες από τις μισές που έχουν ήδη φτιάξει έναν μηχανισμό ελέγχου και οι περισσότερες δεν, ξέρουν, δεν έχουν τίποτα. Τώρα, η πρόταση μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, να μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερες πληροφορίες, να γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει με τις ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Αυτή τη στιγμή η πρόταση είναι μόνο επιθελοντικής βάσης, με την έννοια ότι δεν μπορεί να αναγκάσει τις χώρες να δώσουν τις πληροφορίες και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κατανοήσουμε. Επίσης δεν μπορεί να εξαναγκάσει τις χώρες που δεν έχουν σύστημα να φτιάξουν ένα. Και όσον αφορά τις πληροφορίες και το επίπεδο πληροφοριών που θα απαιτηθεί ή θα ζητηθεί από τις χώρες, είναι σημαντικό να ε, δούμε ακριβώς τι είδους πληροφορίες θα δίνουν οι χώρες, πώς θα εξορροπήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες που έχουν ήδη screening, άρα περισσότερες πληροφορίες ενώ οι άλλοι δεν έχουν τίποτα, που δεν έχουν φτιάξει κάποιο μηχανισμό, έχουν ε, συνήθως λιγότερες πληροφορίες. Και όταν πρόκειται για πληροφορίες, για μας βεβαίως τις εταιρείε είναι πολύ σημαντικό να ε, προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Σε πολλέ περιπτώσει υπάρχει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, όχι μόνο εκτό Ευρώπη αλλά και εντό. Άρα λοιπόν, αν οι πληροφορίε για μία επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με έναν ανταγωνιστή, τότε μπορεί να κινδυνεύει ολόκληρη η επιχείρηση. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που δίνονται. Και έπειτα, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα λειτουργεί με την έννοια ότι είναι αποτελεσματικό, είναι αποδοτικό και ταυτόχρονα παρέχει καλό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κάποιες από τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή, ώστε να εξασφαλίσουμε πως η ερμηνεία που θα είναι η βάση για τη συλλογή των πληροφοριών και για το screening θα είναι εναρμονισμένη εντός της Ένωσης. Αυτές είναι λοιπόν κάποιες πρώτες παρατηρήσεις. Τέλος... η Καρ από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ευχαριστώ. Στην ETUC είμαστε, έχουμε την ίδια θέση με το Business Europe. Δεν έχουμε δηλαδή μια επίσημη θέση ακόμα <clears throat> για την πρόταση της Κομισιόν, όμως καλωσορίζουμε τη συζήτηση αυτή για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και καλωσορίζουμε επίσης την πρόταση για μια ενδελεχή ανάλυση μέχρι το τέλος του 2018. Δεν θεωρούμε ότι ο έλεγχος των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς ήμασταν υπέρ του ελέγχου εδώ και πολύ καιρό. Θέλαμε να υπάρχει μάλιστα ε, μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και ο έλεγχος είναι μια ψηφίδα της πολιτικής αυτής. Καλωσορίζουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου του 2017 για την οικοδόμηση ενός φιλόδοξου, μιας φιλόδοξης ε, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανία, ε, για την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Υποστηρίζουμε την έκκληση προς την Κομισιόν για να υποστηρίξει τον ηγετικό ρόλο των γυναικών και να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανισότητες ε, στους μισθούς και στις θέσεις και στην ιεραρχία. Την κοινή επιστολή της 28 Ιουλίου από πολλά κράτη-μέλη προς την Κομισιόν που έχει κάποια θετικά στοιχεία για τις εξαγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εάν δεν έχει ο επενδυτής ουσιαστική ανεξάρτητη δραστηριότητα πέρα από αυτής της εξαγοράς. Διάφορα κράτη-μέλη επίσης έχουν διαδικασίες ελέγχου που εστιάζουν πολύ λογικό στις εθνικές προτεραιότητές τους. Όμως θεωρούμε ότι η ανάγκη να εξασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ των διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων και μεταξύ των, διαφο... των απόψεων των διαφορετικών υπηρεσιών της Κομισιόν είναι πολύ σημαντική. Καλωσορίζουμε επίσης τα όσα είπε η Επίτροπος Μάλστρομ ότι πρέπει, υπάρχει η επιθυμία να υπάρξει ένα ισότιμο πλαίσιο με τις τρίτες χώρες ό,τι αφορά τις ε, συνθήκες επενδύσεων. Αυτό είναι σημαντικό, θεωρούμε. Και τονίζουμε επίσης το στοιχείο της αμοιβαιότητας. Με συντομή αναφερθήκαμε και σε αυτό. Ζητούμε όμως οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι να εμπλακούν στη δουλειά της ομάδας συντονισμού που αναφέρει η πρόταση αυτή. Η ανακοίνωση μιλάει για τέσσερις κρατικές ε, επιχειρήσεις ε, πολύ ενδιαφέρουσες για, την, για τον έλεγχο. Όλοι οι Κινέζοι επενδυτές είναι υπό τον έλεγχο των κρατικών αρχών, ανεξάρτητα από την τυπική και επίσημη σχέση τους με ε, την κυβέρνηση. Πριν από δύο χρόνια ε, η TUC έκανε μια μελέτη για τις ε, κινέζικες επενδύσεις και την ε, κινέζικη πολιτική επενδύσεων στην Κίνα, καθώς και τις συνθήκες που προσφέρει στους εργαζόμενους. Παραδείγματο χάρη, λαμβάνουμε υπόψη τι έγινε στον Πειραιά. για τις λογικές συμβάσεις, τις συνθήκες εργασίας, τη μείωση των θέσεων απασχόλησης που συνέβησαν εκεί. Επίσης, σας ευχαριστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι στην Κίνα οι αποφάσεις επενδυτικές παίρνονται σε υψηλότατο επίπεδο και η πρωτοβουλία ε, για τη ζώνη και την οδό ε, είναι κάτι που το αποφασίζει η κυβέρνηση. Τώρα, για τον έλεγχο των επενδύσεων για λόγου ε, δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν να μα δοθούν περισσότερε πληροφορίε για το τι καλύπτουν αυτοί οι όροι. Η βιώσιμη ανάπτυξη, τα εργασιακά και το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να καλύπτονται. Και κυρίως ζητάμε η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή η καταστροφή θέσεων απασχόλησης, καθώς και η ποιότητά τους όχι μόνο η, η ποσότητά τους, να αξιολογούνται στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου. Το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και το θέμα τη προστασία των επενδυτών, που δεν καλύπτεται από την ανακοίνωση. Και δεν θα μιλήσω τώρα γι' αυτό βέβαια. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνοδεύει την ευθύνη που έχουν οι επενδυτέ. Να μην το βλέπουμε αποκομμένο δηλαδή. Άκουσα και του προηγούμενους ομιλητέ με προσοχή και η ιδέα που ακούστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων με τις επενδυστικές της αποφάσεις ε, βάζει κάποιες προϋποθέσεις στις ε, δικές μας επενδύσεις. Γιατί να μην βάζουμε Προποθέσει και στι ξένε επενδύσει, Ξένε επενδύσεις οι οποίε επηρεάζουν τι αξίε μα και τον τρόπο ζωή μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν διαφορετικέ προοπτικέ, διαφορετικέ οπτικέ γωνίε και έχουμε περιορισμένο τώρα χρόνο στη διάθεσή μα για ερωτήσει. Οπότε όσοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, ε, να θέσουν ερωτήματα και να τα θέσουν συγκεκριμένα στους ομιλητές. Ε, κύριε Προύστη, ναι. Ένα λεπτό καθένας. Έχω δύο ερωτήσει, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τον ΩΣΑ και για την Business Europe, γιατί όντω αυτή η ακρόαση δεν έχει στόχο να μπει μέσα στην ε, έκθεση, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, γεωπολιτικές ε, Υπάρχουν δυνάμεις που έχουν δείξει τρόπες. Ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει το μεταπητικό σχέδιο της, της Κίνας μέχρι το 2025. Μπορούμε να μιλήσουμε για το δρόμο του μεταξύ. Έχουν αποφασίσει μέσω και έχει πρόθεσμα να κυριαρχήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο σε συγκεκριμένους τομείς. Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Σάντος, μιλήσατε για μελέτη αντικτύπου και εγώ θετικά το δέχτηκα το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ Πολλέ μελέτε αντικτύπου, γιατί στον επιχειρηματικό κόσμο αυτό που έχει σημασία είναι η ε, δυνατότητα αντίδραση. Και αν χάσαμε στα φωτοβολταϊκά είναι γιατί δεν αντιδράσαμε αρκετά γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σήμερα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί στι ανάγκε των επιχειρήσεων για τι τις προστατεύσει καλύτερα. Τώρα, ε, το θέμα είναι ποιου τομεί θα θεωρήσουμε ασφαλεία ή ευαίσθητου κτλ. Γιατί μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Να φτάσουμε όμω ένα κείμενο πριν το τέλο του χρόνου, γιατί όλε οι άλλε χώρε και το είπατε όλοι, ήδη έχουν αυτό το σύστημα ε, διήθηση ε, και ελέγχου και η Ευρώπη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Η Κίνα έχει, η ΕΠΑ έχει. Ε, μόνο η Ευρώπη δεν έχει αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει μονομένα, αλλά το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και νομίζω πως η διευρωπαϊκή διάσταση είναι ατού. Για την Business Europe να ρωτήσω λοιπόν, δεν πιστεύετε πως ένα κράτος μέλος που έχει ένα μηχανισμό ελέγχου δεν είναι ατού για τους ε, ξένους επενδυτές, γιατί εφόσον υπάρχει τέτοιος μηχανισμός, είναι μια νομική ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο. Γιατί εμένα μου φαίνεται πως είναι μάλλον πιο ενδιαφέρον. Εγώ το Δεκέμβριο πήγα στις ΗΠΑ και αυτό μπόρεσα να διαπιστώσω σε σχέση με το ε, CFIUS. Τώρα, για τον ΩΣΑ θέλω να ρωτήσω. Πιστεύετε πως ένας μηχανισμός ελέγχου των επενδύσεων επιτρέπει να προβλέψουμε την προστασία των μελλοντικών τεχνολογιών ή δεν έχουμε αρκετά προβλέψει. Ευχαριστώ. Πρώτον, ε, ο κύριος Ζαντό, έχετε δίκιο κυρία Κάρ ότι ο βιομηχανικός και οικονομικός ε, και, ε, κυριαρχία η εθνική είναι αναχρονισμός και παραλογισμός στο σημερινό κόσμο και αυτό μας εμποδίζει να είμαστε πιο συμπαγεί στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον εκπρόσωπο του Νίλσον Ινστιτούτου για, για να μου, θέλω να μου εξηγήσετε ποιες είναι οι αποτυχίες αυτού του μηχανισμού. Γιατί σπάρουμε ένα παράδειγμα. Η επένδυση της ε, κινέζικης εταιρείας CGN, της πυρηνικής ε, ε εταιρείας στο Point. ήταν βέβαια για πειρατεία, για βιομηχανική πειρατεία στις ΗΠΑ. Η Τερέζα Μέη έρχεται λοιπόν στην εξουσία και λέει έχουμε πρόβλημα ε, και, και ενεργειακής κυριαρχίας με αυτή την εταιρεία. Και τελικά μετά από την πίεση της Γαλλίας και ίσως και των Κινέζων αυτός ο επενδυτής παρέμεινε. Gazprom dans certains pays sur les nationaux. Ε, για την Gazprom ας πούμε. Και εκεί αφήνουμε να μπει ο λύκος μέσα στο κοπάδι των αρνιών. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε και αρνάκια, αλλά ούτε και οι Ρώσοι είναι μονολίκοι, αλλά εν περιπτώσει. Για να... Και μετά έχουμε εκείνο το ταμείο του, εκείνο το νόμιλο του Κουβέιτ που έρχεται και επενδύει. Ναι, λέτε όμως ότι πρέπει να είναι δημοκρατίες, ε, στρατηγικοί τομείς όπως ο Πυρνικός ε, είναι ε, στρατηγικής αλλά έρχεται όμως το κουβέτ και παίρνει μετοχές στην Αρέβα. Ε, πού λοιπόν απέτυχε το σύστημα και ο έλεγχος, ο κύριος Σερμπάτη. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε εκπροσώπους ε, του ΩΣΑ. Η λέξη κλειδί είναι ο έλεγχος, το screening, δηλαδή πώς εξετάζουμε τις ξένες επενδύσεις, ε, πώς μπορούμε δηλαδή να ανακαλύψουμε σε ποιο βαθμό πράγματι αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα τέτοιου είδου επενδύσει. Εσεί έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία σε σχέση με, αυτόν, με αυτή τη διαδικασία ελέγχου. Θα μπορούσε λοιπόν με βάση αυτή την εμπειρία να αναπτυχθεί ένα μοντέλο με βάση το οποίο θα κινούνται τα κράτη-μέλη όταν θα ελέγχουν ακριβώς ε, ε, κατά πόσο μία επένδυση αντίκειται στα εθνικά του συμφέροντα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σόλτς. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ε, στην ΤΟΚ, αλλά και στην Business Έχουμε λοιπόν ε, παγκόσμιες αλυσίδε παραγωγή αξία ε, και έχουμε βέβαια και διάφορα συμπλεκόμενα μεταξύ τους ε, συμφέροντα και ιδιοκτησίες και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνεται με ρεαλιστικό τρόπο ένα investment screening, ένα έλεγχο των επενδύσεων, διατηρώντα ταυτόχρονα βέβαια την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αναφέρθηκα και μία σειρά από ζητήματα σε σχέση με μεγάλες τρίτες χώρες που επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν στον έλεγχο των επενδύσεων. Γιατί ε, σε ένα τέτοιο μηχανισμό δεν περιλαμβάνεται ε, και ακριβώς ε, η διάδικαση ενεργοποίησης, δραστηριοποίησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ελέγχου των επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και ε, έναν αντίστοιχο μηχανισμό ανάληψης ίδιας πρωτοβουλία. Ε, και ποια είναι η τοποθέτηση σε σχέση με αυτό το Business Europe και τη ΕΤΟ. θα ακούσω. Ναι, ε, από την δική μου πλευρά, προς τον ΟΣΕΤ και προς την ΕΤΟ. Α, όχι, ξέχασα τον α, ε, συνάδελφο. Κύριο Ντάκμα, θα έχετε λόγο. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, οι άμεσε ξένε επενδύσει περίθαλψη στην αρμοδιότητα της Ένωσης ε, στο πλαίσιο της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Στο δικό μου βιβλίο, το οποίο έγραψα πριν από δύο χρόνια, δεν υπήρχαν ε, πολλά παραδείγματα ελέγχου, για να μην το πω εμ, παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδου επενδύσει. Οπότε θα ήθελα να ξέρω τι υπάρχει ήδη σήμερα μέρα σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους ελέγχους και ε, θα ήθελα να ακούσω πόσα παραδείγματα υπάρχουν, δηλαδή ε, απτές πραγματικές περιπτώσεις ε, στο παρελθόν τέτοιου ελέγχου. Οπότε συμφωνείτε ή διαφωνείτε ως προς το ότι ε, υπερβολικός έλεγχος των επενδύσεων ουσιαστικά θα μπορούσε να αποβεί προς ε, εις βάρος των επενδύσεων και όχι προς οφελούς τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ερώτημα από την πλευρά μου προς τον Έτου και τον ΩΣΑ. Αυτός ο έλεγχος των επενδύσεων θα πρέπει ε, να περιλαμβάνει στα κριτήρια της αξιολόγησης και την ποιότητα της επένδυσης. Για παράδειγμα, αν εξετάσω τα παραδείγματα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Volvo είχαμε μια τέτοια άμεση ξένη επένδυση, η οποία όμω περιέκοψε ε, την έρευνα και το, τον όγκο της παραγωγής. Με αποτέλεσμα βέβαια η Volvo τελικά να ε, μην υπάρχει πλέον. Ε, Τώρα βλέπουμε ένα διαφορετικό, μια διαφορετική ε, προσέγγιση. Οπότε το ερώτημά μου είναι θα πρέπει μέσα στο screen να περιλαμβάνεται και η ποιότητα της επένδυσης ως κριτήριο. Και υπάρχει ενδεχομένω και κάποια εμπειρία στη δική. Τώρα λοιπόν να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές ε, των πάνελ. Με αντίθετη σειρά, Ελίνα λοιπόν πρώτη έχει το λόγο. Uh, the, the question of why isn't uh, the... Γιατί Δεν υπάρχει τιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δράσει. Δεν ξέρω, ρωτήστε την Κομισιόν. Γιατί για κάποια εμπορικά θέματα εμείς γράφουμε επιστολές στην Επιστροπή για να απαντήσει επί χρόνια. Και όμως δεν αλλάζει η στάση της. Τώρα, για το αν ο έλεγχος των επενδύσεων γίνεται και με ποιες προϋποθέσεις, σας παραπέμπω στη μελέτη στην οποία αναφέρθηκα, σε ό,τι αφορά κυρίω τι ε, κοινωνικέ επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν δυνατότητε να θέσουμε τις προϋποθέσεις όταν ετοιμάζουμε τις συμφωνίες. Υπάρχει ένα παράδειγμα συγκεκριμένο για το Χίνκλι, ας πούμε. Και για τα θέματα του εργατικού δυναμικού. Τι ποσοστό των ε, εργαζόμενων από την τοπική κοινωνία πρέπει να χρησιμοποιείται Παραδείγματο χάρη στην, στην περίπτωση του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά. Δεν υπήρχαν καθόλου προϋποθέσεις για, για να γίνει κινέζικη επένδυση και το χρησιμοποίησε ο Κινέζο επενδυτή για να εξαρθρώσει τη δομή που υπήρχε ήδη. Και τελικά έχουν 200 ε, εργαζόμενους, όλοι έχουν διοικητικές θέσεις, ενώ οι, οι εργάτες ουσιαστικά που δουλεύουν επί τόπου ε, είναι εξωτερικοί συνεργαζόμενοι, έχουν 10 με 15 θέσεις, ε, μέρες άδειε. Ε, οι βραδινές βάρδιες, οι αργίες, Βασικά όλα αυτά θα πρέπει να μπαίνουν ε, στη συμφωνία όταν υπογράφεται. Ευχαριστώ. Για το θέμα του εισηγητή για την ασφάλεια δικαίου και για το αν οι επιχειρήσεις δεν είναι ικανοποιημένες. Όχι. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το πλαίσιο είναι πιο σαφές. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις ε, για να υπάρξει μηχανισμό ελέγχου εφόσον θέλουν να το χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ξέρουμε ποιε είναι οι αρχέ πια. Ε, βάσει των οποίων λειτουργεί ο μηχανισμό διαφάνεια, τη δυνατότητα ε, ένδικων μέσων και την ανάγκη αντικειμενικών κριτηρίων. Είναι σημαντικό αυτό και φυσικά συμφωνούμε. Όταν μιλάμε τώρα για τη μελέτη αντικτύπου, μιλάμε γι' αυτό για να ξέρουμε σε ποιο βαθμό η πρόταση μπορεί να προχωρήσει και για να είμαστε σίγουροι ότι υλοποιεί τους στόχους. Αυτή ήταν η ιδέα. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, πληροφορίε για τις ξένες επενδύσεις και ό,τι συμβαίνει τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητάμε αυτό γιατί θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει στην πράξη. Αλλά και γιατί συμφωνούμε βεβαίω. Ένα σημείο που νομίζω ακούστηκε και πριν και που τονίζω και εγώ, είναι σημαντικό στη διαδικασία αυτή να υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, διαφορετικές προτεραιότητες στα κράτη-μέλη και με αυτή την πρόταση δεν θα πρέπει να βάλουμε και ένα νέο στοιχείο που θα καθυστερεί τις διαδικασίες, γιατί τότε μπορεί να αποτραπούν κάποιες επενδύσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Και αυτό είναι σημαντικό για το θέμα της απασχόλησης και το... τα εργασιακά. Ε, όπως είπε και η Λίνα, αυτά σε πολλές περιπτώσεις είναι τμήμα των συμβάσεων εδώ όμως μιλάμε για τα έργα τα ίδια. Ε, και συχνά ε, σε αυτά τα project ε, το κράτος έχει σημαντική, σημαντικό ρόλο και παρέμβαση. Φυσικά όταν τα έργα είναι μικρά είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Γιατί μερικές φορές έχουμε ε, φορείς δημοσίου ιδιωτικού σε κάποια έργα. Ή μερικές φορές, ας πούμε, σε κάποιες εταιρείες υπάρχει έντονη κρατική παρουσία ε, τότε το κράτος μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα για τις ιδιωτικές συμβάσεις βεβαίως το πράγμα ε, α, επαφίεται ας πούμε στη βούληση των δύο μερών. Γιώνας. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές για τις ερωτήσεις σας. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Εγώ αυτό που προ... προσπάθησα να πω ήταν ότι όσο ταχύτερα γίνει ε, ένας έλεγχος ε, των επενδύσεων από τη δική μας πλευρά, τόσο το καλύτερο και αναφέρθηκε αυτό σε ό,τι αφορά την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, Κούκα. Ε, δηλαδή και εδώ πάλι σε ό,τι αφορά την περίπτωση τη Κούκα η συζήτηση ξεκίνησε από το βιβλίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό τι μα καταδεικνύει ότι χρειαζόμαστε το δικό μα σύστημα ελέγχου των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει και περισσότερο συντονισμό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Συνεννόηση δηλαδή μεταξύ των χωρών. Ποιε πληροφορίε έχει η μία και ποιε οι άλλοι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και δυστυχώ διαπιστώνουμε ότι ακριβώς οι Αμερικανοί ανησυχούν με το τι συμβαίνει εδώ στην Ευρώπη, ότι δεν υπάρχει ένας, μια τέτοια συντονισμένη απάντηση. όσα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες του μέλλοντος, Ε, νομίζω πως είναι ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν ε, χρειάζεται να το καλύψουμε σήμερα. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οπότε ε, τα ωφέλη μιας επένδυσης και το τι αποτελείται η τεχνολογία του μέλλοντος και τι όχι, είναι διαφορετικά ζητήματα. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε από αυτού σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα μοντέλο με βέλτιστε πρακτικέ, εδώ θα πρέπει εσεί να κάνετε τη σχετική επιλογή. Δηλαδή, θα πρέπει να δείτε ποιε είναι οι ικανότητε ενό τέτοιου συστήματο ε, που επιθυμείτε, ποιου πόρου θα έχετε στη διάθεσή σα και ποιο επίπεδο ελέγχου των επενδύσεων είναι εκείνο που θεωρείται απαραίτητο. Ε, αυτές είναι αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής και όχι αποφάσεις σε επίπεδο ε, εμπειρογνωμόνων. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές και κάποιες κακές πρακτικές, αλλά οι καλές πρακτικές που θα επιλέξετε εξαρτώνται ακριβώς από τις αξίες και τις προτεραιότητες που εσείς θα θέσετε. Σας ευχαριστώ. Ε, νομίζω πως θα πρέπει να αποσχολήσετε το διπλωματικό σώμα. Ο κύριο Προύστο, για να κλείσουμε την ακρόαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο και όλους τους ομιλητές και σας Πρόεδρε που οργανώσατε αυτή την ακρόαση, πολύ τεχνική. Όλες οι παρεμβάσεις ε, ήταν αλληλοσυμπληρούμενες και θα μου επιτρέψουν να απαντήσω στις βασικές τρεις, στις βασικές τρεις ερωτήσεις που πρέπει να θέσουμε ως νομοθέτες στον εαυτό μας. Πώς θα συνεχίσουμε να προσελκύουμε ξένες επενδύσεις πρώτον. Δεύτερον, πώς θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ξένων επενδύσεων προστατεύοντας τους στρατηγικούς τομείς της Ένωσης. Τρίτον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοχλό ούτως ώστε να ανοίξουμε τις ξένες αγορές της ευρωπαϊκής επενδύσεις. Όπως είπατε, η Ευρώπη είναι ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις και αυτό σημαίνει οικονομικός δυναμισμός και ανάπτυξη. Οι, που έχουν, οι χώρες που έχουν ε, έλεγχο των επενδύσεων δεν σημαίνει ότι είναι κλειστέ στις επενδύσεις. Λοιπόν, θυμίζω τα όσα μας είπε ο κ. Σμιρ από την Αμερική, που υπάρχει αυτό το εργαλείο από το 1975 στι ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή διάσταση ε, είναι καινοφανής, αλλά υπάρχει κάποια εθνική εμπειρία σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Η Λετωνία και η Γαλλία σας παρουσίασαν σήμερα ε, ενδιαφέρουσα στοιχεία του δικού του συστήματος. Αυτά τα εργαλεία που σας παρουσιάστηκαν έχουν ε, και κενά, αλλά είναι ισορροπημένα, προβλέψιμα και υπάρχουν και προβλέπουν και ένδεικα μέτρα μέσα. Ε, οι χώρες ε, που έχουν έναν τέτοιο μηχανισμό δεν βλέπετε ότι έχουν έλλειμμα ε, επενδύσεων γιατί το φιλτράρισμα και ο έλεγχος είναι πολύ περιορισμένος. Οι επενδύσεις εξαρτώνται από το πολιτικό κλίμα, από τις πρωτοβουλίες που γίνονται στο τοπικό επίπεδο και κυρίως από τα πλεονεκτήματα πολύ περισσότερο από ότι ένα μηχανισμό ελέγχου. Ε, και επίση, μην ξεχνάτε την επίπτωση που μπορεί να έχει μια επιχείρηση σε άλλου τομεί στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Ακριβώ γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση. Η εξαγορά μια επιχείρηση μπορεί να έχει επιπτώσει στη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην άλλη άκρη τη Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον να ανταλλάσσουμε πληροφορίε, ε, όπω είπε και η κυρία Καρ, γιατί συμφωνώ με την αποψή τη, για τα κοινωνικά θέματα και τα περιβαλλοντικά θέματα. Σε ένα τόσο γρήγορο. Ε, ασταθή κόσμο, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι γίνεται στην άλλη άκρη τη Ευρώπη, σε επιχειρήσει μα, γιατί πραγματικά είναι μειονέκτημα, για να μην πω λάθο. Χωρί να θέλουμε να ε, φτάσουμε στο κίνδυνο μηδέν, πούμε, στον ελληνικό κίνδυνο, τουλάχιστον να το μειώσουμε. Ε, νομίζω ότι θα χάσουμε αν δεν το κάνουμε. Τελειώνω. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά όλου του ομιλητέ τέθηκαν σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάρα πολλά ερωτήματα. Ε, μπορώ να σας πω ότι πολλά από αυτά είναι καινούρια και για το Κοινοβούλιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κρατήστε όμως ότι υπάρχει μια εμπειρία τουλάχιστον στα κράτη-μέλη και σε όλο τον πλανήτη. Ε, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να βοηθηθούμε, για να βρούμε ένα μηχανισμό ισορροπημένο, αναλογικό και κυρίως, και τονίζω και υπογραμμίζω, αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες και ορισμένοι από εσά κάνατε και μακρύ ταξίδι για να έρθετε ως εδώ. Ήταν όλα αυτά πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν ε, μια ακρόαση που μας βοήθησε να κατανοήσουμε περισσότερο την κατάσταση. Θα συνεχίσουμε την εργασία μας. Το Φεβρουάριο θα έχουμε ένα έγγραφο εργασία από τον εισηγητή μας και καλή επιτυχία σε όλους. So, now we switch to... Τώρα περνάμε στο σημείο 23 της ημερησίας μας διάταξης ε, Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας με την Ιαπωνία. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο και τώρα η Επίτροπος θα μας παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και όλοι όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν εισήχως, παρακαλώ. Please be quiet. Work is still going on. Παρακαλώ ησυχία, οι υπόλοιποι δουλεύουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να φύγετε ησύχως. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να συνεχίσουμε. Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές. Όπως γνωρίζετε, στις 8 ε, Δεκεμβρίου πέρυσι ανακοινώσαμε την ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας για οικονομική εταιρική σχέση και αμέσως μετά δημοσιεύσαμε τη συμφωνία ώστε να την μελετήσετε ε, online. Βεβαίως πρόκειται για μέγα επίτευγμα για την Ιαπωνία και για την Ευρώπη έχει μεγάλη οικονομική αξία, αλλά είναι και στρατηγική σημασία, καθώ στέλνει μήνυμα στον κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία είναι ε, τιμέ να στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία επί τη βάση μια ε, δίκαιων και ρυθμισμένων αγορών αποφεύγοντας ε, το πειρασμό του προστατευτισμού αλλά και την άναρχη απελευθέρωση. Η οικονομική αυτή συμφωνία είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο συνολικές ε, ε, ε, συμφωνίες που έχουμε συνάψει ποτέ. Απελευθερώνει τους δασμούς 90% για τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα προστατεύει πάνω από 200 γεωγραφικές ενδείξεις ευρωπαϊκές και επίσης καταργούνται διάφορες μη διάφοροι μη δεσμολογικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς. Πρόκειται για 600 εκατομμύρια κόσμο, περίπου 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ανοίγονται διάφορες ε, δυνατότητες εμπορικές ε, που θα ενισχύσουν τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας και βεβαίως θα ενισχύσουν τη συνεργασία εν γέννη μεταξύ της Ένωσης και της Ιαπωνίας γιατί δεν ενώνονται μόνο αγορές αλλά και οι λαοί και αυτό ενισχύει την κοινή μας ανταγωνιστικότητα αλλά και τις προσπάθειες συνεργασίας για αριθμιστική ευθυγράμμιση με τα διεθνή στάνταρα. Τον Ιούλιο αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο αυτής της συμφωνίας από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου σε Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, γιατί αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τη φύση της συμφωνίας. Πρόκειται για μια νέα οικονομική σχέση ανάμεσα στην Ένωση και την Ιαπωνία και όχι μόνο το τέλος μιας διαπραγματευτικής διαδικασία. Να σα δώσω λίγες λεπτομέρειες. Ξέρω πως έχετε ενημερωθεί ε, προηγούμενα. Από τον Ιούλιο, όταν ολοκληρώσαμε επί τις αρχές τη συμφωνία, που σας ενημέρωσα αμέσω μετά και σας παρουσίασα τη συμφωνία, έγινε πολλή δουλειά τεχνικής φύσης, μετάφραση των νομικών κειμένων ε, στις αρχές που συμφωνήσαμε. Ολοκληρώσαμε την επαλήθευση των προγραμμάτων για την πρόσβαση στην αγορά, για την αγαθά, τους διαγωνισμού, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες. Ολοκληρώσαμε και το κεφάλαιο για τη διαφάνεια. Επίσης, βελτιώσαμε το κείμενο σε μεγάλο βαθμό για το κεφάλαιο εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Ενισχύσαμε δηλαδή τη δέσμευσή μας στην κοινή στη Συμφωνία του Παρισσού για τις κλιματικές αλλαγές. Πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει αυτό σε συμφωνία εμπορική. Εισάγαμε ένα εμπορικό μηχανισμό σε αυτό το κεφάλαιο και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για το Ευρωκοινοβούλιο και ίσως ε, να παρατηρήσατε ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων. Αυτό είναι ο μόνος τομέας όπου δεν μπορέσαμε να βρούμε συμφωνία με τους Ιάπωνες φίλους μας το Δεκέμβριο. Και αυτή η συμφωνία βασίζεται στο σύστημα της ε, επίλυσης των διαφορών. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε στο παλαιό σύστημα SDS μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία μόνο με βάση το επενδυτικό δικαστήριο. Και οι Ιάπωνες είναι πιο προσιλωμένοι στο παλιό σύστημα ISTS που λένε ότι για εκείνους έχει λειτουργήσει καλά συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις για να βρούμε μια λύση εδώ. Θα ξανασυζητήσουμε σε μια-δύο εβδομάδες. Έχουμε κάνει πρόοδο προσπαθώντας να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και έχουμε συμφωνήσει. Επειδή έχουμε συμφωνήσει για όλα τα άλλα, θα ήταν κρίμα να καθυστερήσουμε τη συμφωνία μόνο λόγω αυτού. Σύντομα λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να αρχίσει να ε, ισχύει όσο γίνεται πιο σύντομα και οι Άπωνες συμφωνούν μαζί μας. Έχουμε λοιπόν λάβει μέτρα ε, για να συντομεύσουμε τις διαδικασίες. Έχουμε, ε, οριστικοποιούμε την νομικό έλεγχο και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες αυτό όπως απαιτείται. Και μετά ελπίζουμε να υποβάλουμε τη συμφωνία στο Συμβούλιο του Άνοιξη για να μπορέσουμε να την ε, υπογράψουμε ήδη το καλοκαίρι και θα σας σταλεί αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Την εξετάστε και ελπίζουμε να την εγκρίνετε και αν όλα πάνε κατευχήν θα αρχίσει να ισχύει στα τέλη του έτου τους ή στις αρχές του επόμενου. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα είναι το μπαλάκι στο δικό σας γήπεδο ε, και βασιζόμαστε σε εσάς ώστε να προωθηθούν σε ένα νέο επίπεδο οι σχέσεις μεταξύ Ένωσης και η Σε Ευχαριστώ όλους σας και ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές που συνεργαστήκαμε πολύ καλά ε, μαζί και προσβλέπουμε ε, στη συνέχιση της ε, αγαστής αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή, Επίτροπε. Είμαστε περιορισμένοι χρονικά, έχουμε ένα μισάωρο. Παρακαλώ να υποβάλλετε τα πιο σημαντικά ερωτήματα που έχετε και περιοριστείτε ο εισηγητής στο δίλεπτο και οι υπόλοιποι στο μονόλεπτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα συνάδελφοι. Ευχαριστώ Επίτροπε Λέω ο Σίλβα Περαϊρά. Ε, συγχαρητήρια για την ε, ολοκλήρωση αυτών των πολύ σημαντικών διαπραγματεύσεων. Είναι η πιο σημαντική διμερή εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντική οικονομικά και στρατηγικά. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υπογράψει το τελικό κείμενο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συνένεσή του, ναι ή όχι, ε, αφού εξετάσει το κείμενο του, της συμφωνίας, τη συγκατάθεσή του μάλλον. Και ελπίζουμε αυτό να γίνει ε, και είμαστε σίγουροι θα γίνει πριν από τις, εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα βασικά αποτελέσματα για το γεωργικό τομέα, που πάντα είναι πολύ ευαίσθητος Βλέπουμε ε, για τις εξαγωγές ε, αγιορικών προϊόντων να εξάγονται χωρίς δασμό. Ευρωπαϊκό κρασί, ας πούμε. Ε, δεν θα υπάρχουν δασμοί ε, μόλις τεθεί ε, σε εφαρμογή συμφωνία. Θα υπάρχουν ποσοστώσεις σε τομείς όμως σημαντικούς για την Ιαπωνία. Για τις γεωγραφικές ενδείξεις είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Το καλύτερο που είχαμε ποτέ, νομίζω. Ε, πετύχαμε κάτι παραπάνω από τη ΣΥΤΑ, ε, στον τομέα αυτό, στι γεωργικές ενδείξεις δηλαδή, για τα μη δασμολογικά μέτρα, ε, ε, συνδρομικό τομέα, υπάρχει η ρήτρα της επιχειρησιακής ασφάλειας η οποία έχει ακυρωθεί πλέον, να τονίσω και τα αποτελέσματα όμως σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καλωσορίζω το γεγονός ότι στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων ε, μία ρήτρα αναθεώρηση για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού τελικά μπόρεσε να συμφωνηθεί και να εισαχθεί στο κεφάλαιο. Για την κλιματική αλλαγή έχουμε επίσης πετύχει αποτελέσματα καλύτερα από τη ΣΕΤΑ. Θα θέλαμε όμως μια πιο ισχυρή διατύπωση για τα όσα λέει η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό έχει να κάνει με τις αντιστάσεις των ε, Ιαπωνέζων παρά οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι μπήκε δηλαδή. Κλείνοντας, ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα μπορέσει να συνεισφέρει αποτελεσματικά για ένα εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες και για μια πολύ φιλόδοξη εμπορική ατζέντα. Φυσικά θα συζητήσουμε το κείμενο αυτό καθεαυτό. Πολύ σημαντικές συζητήσεις στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Δέκα ομιλητές θέλουν το λόγο. Α, 11-12. Ένα λεπτό καθένα το πολύ, γιατί η Επίτροπο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να σα απαντήσει. Ένα λεπτό. Ε, λέγονται πολλά, ο Γουαλέσα, για το εμπόριο και το περιβάλλον, το επενδυτικό. Δεν υπάρχει διμερή συμφωνία για τις επενδύσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Ιαπωνίας. Και ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που θα θέλαν να χωριστεί το εμπόριο από τις επενδύσεις. Πόσο σημαντικό είναι για την Επιτροπή να υπάρχει η προστασία των επενδύσεων. Υπάρχει ευελιξία από την Κομισιόν. Ε, περιμένοντας μια επενδυτική συμφωνία ε, και μια χωριστή συμφωνία για τις επενδύσεις, τι κάνει η Κομισιόν στο μεταξύ. Επίσης αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο. Για τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Θα τεθούν σε εφαρμογή πριν από τη συμφωνία με την Ιαπωνία ή όχι, ή μετά. Ε, έχετε πάρα πολλά πάντως να κάνετε. Σας συγχαίρω για το αποτέλεσμα. Ο κύριος ή ε, από τη δική μα πλευρά ω φιλελεύθεροι επιχαίρουμε ε, την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων και αντιλαμβανόμαστε ε, το δυναμικό μια τέτοια συμφωνία. Ήδη αναφέρθηκαν τα όσα συμφωνήθηκαν σε επίπεδο γεωγραφικών ενδείξεων αλλά και δημοσίων συμβάσεων. Πράγματι αποτελούν όλα αυτά καλή βάση για περαιτέρω διαπραγμάτευση. και εγώ θα ήθελα να ακούσω λίγα παραπάνω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων. Ε, δηλαδή, ρεαλιστικά θα προλάβει να γίνει κάτι εδώ, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον υπό την Πολυγαρική Προεδρία ή όχι. Στο εγγύς μέλλον δηλαδή θα ξεκινήσετε και επίσης σε σχέση με τις ροές πληροφοριών και την προστασία των δεδομένων αναφέρθηκαν κάποια ε, Σχόλιο ότι υπήρξαν κάποια προβληματάκια εκεί. Ισχύει αυτό ή όχι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ο κ. Καμάλα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε και σε είδη. Ε, επειδή δεν έχω αρκετό χρόνο, να περάσω κατευθείαν στα ερωτήματά μου καθώς οι ροές των πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την συμφωνία και υπάρχει και η προθεσμία των τριών ετών για την αναθεώρηση, έχει εξετάσει τη ρήτρα της επάρκειας αυτό το που Provision ε, η Επιτροπή. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά ε, την παράλληλη ε, συμφωνία, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, είναι, θα μπορούσε να είναι πιο αποδεκτή από την Ασία. Και από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, γιατί δεν περιλήφθηκαν ε, γιατί είχαμε τα ζητήματα με τις, ε, με τις των πληροφοριών, ε, δηλαδή στη ΣΥΤΑ είχαν περιληφθεί, αλλά όχι εδώ. Γιατί υπήρξαν κάποιοι διαφορετικοί λόγοι ή ήταν τα δεδομένα. Και μετά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των επενδύσεων. Εάν τελικά λάβουμε, συμπεριλάβουμε και αυτή την πρόταση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την πολυμερή επίλυση επενδυτικών να διαφωνώ και τι επενδύσει εδώ, τι ακριβώ θα μπορούμε να αναμένουμε. Ευχαριστώ κύριο Ζαντόχη. Ευχαριστώ κυρία Πίτροπε. Πρώτη ερώτηση. Μιλάτε για το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πάντοτε το συζητάμε, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι είναι το μόνο κεφάλαιο το οποίο δεν, δεν, δεν συνοδεύεται από διατάξεις περικυρώσεων όπως όλα τα άλλα. Και επίσης, καθώς ξέρετε ότι έχουμε κάποια προβληματάκια με την Ιαπωνία, είτε για τη ξυλία, εισαγωγή παράνομες ξυλίες στην Ιαπωνία, ενώ εμείς έχουμε αναπτύξει το φλεκ που είναι πρότυπο. Έχουμε προβλήματα με την αλληλεία. Αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού που τα έχει όλα και τίποτα. Μπορεί να, να αναφερόμαστε εκεί, αλλά δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό εκεί. Δεύτερο, για τα ε, προσωπικά στοιχεία, αλλά αυτό υπόθηκε γιατί υιοθετήσαμε θέση για τα προσωπικά στοιχεία στις εμπορικές συμφωνίες. Και τώρα, για Τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την ποιότητα, για το θέμα της διαφάνειας και θέλω να ξέρω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα όσα θα αναπτύξουμε εμείς στην Ευρώπη κατά της ε, φοροδιαφυγής ε, και υπέρ της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα, δεν θα το διακυβεύσει αυτή η συμφωνία με την ε, Ιαπωνία. Σόλτς. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Όπως ε, α, ήδη αναφέρθηκε επανειλημμένα το κεφάλαιο σε σχέση με τις επενδύσεις, εγώ θα ήθελα ε, να το σχετίσω με την οικονομική σταθερότητα στις χώρες μας. Ε, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με το γενικότερο ζήτημα τη μεταχείρισης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ε, Πώ λοιπόν θα ρυθμίσετε αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τι επενδύσει, μετά, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή το κεφάλαιο σε σχέση με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν μια σειρά από α, κενά παραθυράκια των εισαγωγικών στη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις ε, για την υποχρεωτική κοινοποίηση και τα όσα δηλαδή προβλέπονται εδώ σε ό,τι αφορά την δέουσα κοινοποίηση. Εδώ ε, θεωρούμε δηλαδή πως δεν είναι πλήρη τα όσα προβλέπονται. Όταν θα οριστικοποιήσουμε το κεφάλαιο ή μια συμφωνία τέλος πάντων σε ό,τι αφορά τις ροές πληροφοριών, θα υπάρξει, θα ληφθούν και αυτά τα ζητήματα υπόψη. Με άλλα λόγια, δηλαδή, θα είναι μια δυναμική συμφωνία, θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μα στο μέλλον τέτοιου είδου δεδομένα. Ευχαριστώ, λέω ο πρόεδρο, ο κύριο Σαχαντήλ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και κυρία Επίτροπε, νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως είναι σημαντική από γεωπολιτική άποψη η σύναψη αυτή τη συμφωνία καθώ θα βάλει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίκεντρο του ελεύθερου εμπορίου σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε απομακρύνονται από αυτό. Είναι λοιπόν σωστή η χρονική συγκυρία, αλλά λαμβάνοντα υπόψη όλο αυτό το πλαίσιο ανακύπτει για μένα το ε, ίδιο ερώτημα όπω αυτό που έθεσε ο κύριο Βαλέσα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ή να ξεχνούμε και άλλε. Ε, συμφωνίες τις οποίε ε, προετοιμάζουμε αυτή την περίοδο, για παράδειγμα αυτές ε, τις συμφωνίες δηλαδή ελευθεροπορίου με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Δηλαδή, τι λέτε ουσιαστικά, προτεραιότητα πρώτα στην Ιαπωνία και μετά Σιγκαπούρη και Βιετνάμ ή θα σεβαστείτε το γεγονός ότι αυτές οι συμφωνίες δηλαδή με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει ε, ω προ τη διαπραγμάτευση νωρίτερα και θα πρέπει να οριστικοποιηθούν ταχύτερα. Μαρία Ρένα, η θέση του Συμβουλίου καταρχά ό,τι αφορά το διαχωρισμό ε, ανάμεσα στην ε, συμφωνία την εμπορική και την επενδυτική. Ε, εσείς λέτε ότι θα τις διαχωρίσετε. Υπάρχει σαφή θέση του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Δεύτερον, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Ζαντό και αυτά που είπε ο κ. Σόλτ για το κεφάλαιο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και την ανταλλαγή δεδομένων προσωπική αφήσεω. Ε, γιατί αυτά που διαπραγματευόμαστε στην Ιαπωνία, ή μάλλον αυτά που διαπραγματεύομαστε στην Ιαπωνία, να μην ε, αποδυναμώσουν τη θέση εδώ στην Ευρώπη. Έπειτα, το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, ξέρουμε ότι στην Ιαπωνία, σε ό,τι αφορά την παράνομη ξυλία και και την παράνομη αλία, η Ιαπωνία δεν σέβεται τι διεθνεί συνθήκε. Το να μην έχουμε κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να μην έχουμε και κυρώσει αυτή την ε, συμφωνία είναι μια αμαρτία, γιατί υπάρχουν ήδη δυσκολίε με την Ιαπωνία. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με κυρώσει. Τέλο, η Ιαπωνία έχει μια πολύ ενσωματωμένη ε, οικονομία στην Ασιατική Ήπειρο. Με ε, ελάφρυνση των κανόνων προέλευση. Θα είναι λοιπόν πολύ ανταγωνιστική όταν έχουμε και στοιχεία παραγωγής που παράγονται αλλού, σε άλλες ασιατικές χώρες. Τι γίνεται λοιπόν, έχετε στοιχεία για τι κάνουμε, γιατί στην, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο οι οικονομίες μας δεν είναι τόσο ενσωματωμένες όσο στην Ασιατική Ήπειρο. Κύριος Χάινς. Κυρία. Ε, το δικό μου γενικό ερώτημα είναι το εξή. Γιατί ε, το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιλαμβάνεται και αυτό στο μηχανισμό επίλυση των διαφορών. Ε, από εκεί και μετά αυτή η ρήτρα αναθεώρηση, το review clause, πώ ακριβώ θα εφαρμοστεί στην πράξη. Και μετά, Ε, όλες τις, ε, τις, τα, τα επιμέρους τμήματα θα πρέπει όλα αυτά να κυρωθούν ε, προτού κατακυρωθεί και οριστικοποιηθεί η συνολική συμφωνία ή όχι. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, πώς ακριβώς προτείνετε να διασφαλίσετε ότι θα παραμείνει η ίδια προστασία αυτών των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καλή τύχη, κυρία Επίτροπε, για αυτή την πολύ ε, σημαντική συμφωνία με την τέταρτη πιο σημαντική οικονομία του κόσμου. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα ανοιχτό εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες. Ε, θα κερδίζουμε ένα δισεκατομμύριο ε, ευρώ το χρόνο λόγω του ανοίγματο της αγοράς. Ε, με ωφέλη για τους καταναλωτές και σας συγχαίρω για το χρονοδιάγραμμα που πετύχατε. αυτή η συμφωνία θα ανοίξει πόρτες στον τομέα των εξαγωγών. Τι και να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις. Ε, θα, ε, ευχόμαστε καλή τύχη στην κύρια διαπραγματεύτρια. Θα θέλαμε τα, ίδια πράγματα να τα πετύχουμε και συμφωνία με το Μερκοσούρ. Πιστεύετε ότι αυτός ο μηχανισμός προστασίας της επενδύσεως και το θέμα της επίλυσης των διαφορών για τις επενδύσεις μπορεί να περιπλέξει την, το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει, ε, ούτως ώστε να καθυστερήσει η επικύρωση της συμφωνίας αυτής ε, και η σύμφωνη γνώμη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριο Ντάρτμουντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και Ελβετίας ετέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 2009. Η Επίτροπος ε, είπε στην αρχή ότι αυτό μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή κάποια στιγμή στι αρχέ του 2020. Δεν ξέρουμε ακόμα αν το κοινοβούλιο τη Βαλωνία, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να πει και αυτό την άποψή του, α πούμε, όπω έκανε για άλλε εμπορικέ συμφωνίε. Ξέρω και το ερώτημά μου, από την εμπειρία σα. Είναι ευκολότερο, πιο απλό, μια χώρα μόνη τη να συμφωνήσει για εμπορικά θέματα από ότι είναι για ένα μπλοκ, α πούμε, 27-28 χωρών που έχουν τελείω διαφορετικέ οικονομίε και τελείω διαφορετικά συμφέροντα να καταλήξουν συμφωνία με μια τρίτη χώρα. Έχετε μια συγκεκριμένη χώρα στο μυαλό σα. Ε, μπορείτε να το εικάσετε. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω πάντως. Αλέσια. Ναι, και εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία ε, από κάθε άποψη γεωπολιτική, στρατηγική αυτής της συμφωνίας. Ε, μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά ε, το γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Μέσα στη συμφωνία υπάρχει μια προστασία υποδεέστερη σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, και θέλω διευκρίνηση γι' αυτό, έτσι, υπάρχουν παρεκκλήσεις για κάποια ε, γαλακτοκομικά προϊόντα που επιτρέπουν ή μάλλον που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτά που έχουμε πετύχει ε, στα πλαίσια της συμφωνίας που τον Καναδά, με τη ΣΕΤΑ. Δηλαδή, μπορούν να καταχωρηθούν γενώσιμα ονόματα, όπως Παρμεζάν, ας πούμε, ε, Παρμετζάνο Ρετζάνο, και παράλληλα μπορούν να τιμωρηθούν συμπεριφορές που δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την προέλευση αυτών των προϊόντων. Αν η συμφωνία είναι ίδια με του Καναδά, τότε η προστασία είναι καλή. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση, μπορεί να τιμωρηθούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο γαλακτοκομικό τομέα. Παράλληλα, μπορεί να τιμωρηθούν όχι τόσο αυτά που παράγονται στην Ιαπωνία, γιατί ούτως ή άλλως η Ιαπωνία δεν παράγει πολύ τέτοια προϊόντα, αλλά μέσω προϊόντων τρίτων χωρών που είναι ε, παρόντα στην Ιαπωνέζικη αγορά. Μέσω αυτών μπορούν να τιμωρηθούν τα δικά μας προϊόντα τελικά. Thank you. Um, voorzitter. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για την νέα παράγραφο σε σχέση με την προστασία του κλίματος, όπου γίνεται λόγος για συνεργασία κατά των κλιματικών αλλαγών. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε πως είναι μια παράγραφος που θα χρησιμοποιηθεί και για τις άλλες δύο συμφωνίες με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη και πώς ε, σκέφτεστε να υλοποιήσετε αυτές τις φιλοδοξίες. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα καταλήξουμε σε μία αύξηση των εκπομπών. Πώς θα εγγυηθείτε ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα τα οποία απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και ότι δεν θα ε, σταλούν και πάλι σε μια ενδεχόμενη διατησία. Και έπειτα... Είναι μια χαμένη ευκαιρία το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν συμπεριέλαβε στη συμφωνία την Λία Φάλαινας, ε, τη φαλαινοθυρία, γιατί και αυτό σημαίνει η προστασία του περιβάλλοντος. Ε, λάβατε μια αναφορά με 260 υπογραφές, χιλιάδες υπογραφές ε, κατά της φαλαινοθυρίας. Θα, η αξιοπιστία της Ευρώπης θα αυξανόταν, αν είχε συμπεριληφθεί εδώ και το θέμα αυτό. Επίτροπο, σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα για τις επενδύσεις. Έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχουν εθνικές διμερείς ε, συμφωνίες ε, ανάμεσα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και την Ιαπωνία σήμερα. Ο στόχος να έχουμε ένα κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων με την Ιαπωνία και είναι κάτι που μας ζήτησαν και τα κράτη-μέλη. Αλλά επειδή δεν μπορέσαμε μέσα στο νέο μοντέλο να το περιλάβουμε. Όταν συμφωνήθηκαν όλα τα άλλα, σκεφτήκαμε αυτό λίγο να το αναβάλουμε και να σας παρουσιάσουμε αυτή τη συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει την προστασία των επενδύσεων όπως σήμερα ε, ε, θα θέλαμε θα σας, θα σας υποβληθεί και θα σημαίνει προστασία των επενδύσεων μόνο για την Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε καταλήψει την ιδέα. Συζητάμε με τους Ιάπωνες φίλους, προσπαθούμε να τους το εξηγήσουμε, να καταλάβουμε πώς το έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Επίσης, ταυτόχρονα ε, συνομιλούμε με τους Ιάπωνες για το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο που προχωράει, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να οργανωθεί και πιστεύω πως θα υπάρξουν νέες συζητήσει ανάμεσά μας και τους Ιάπωνες αργότερα και θα σας ενημερώσω για το πώς προχωρούν. Πάντως προβλέπουμε να σας υποβάλουμε την, την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και όταν θα έχει αυτό θα ολοκληρωθεί θα έχουμε μια άλλη μειχτή συμφωνία αν περιλαμβάνει Okay και την προστασία των επενδύσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε χαλαρώσει άλλε εμπορικέ συμφωνίε. Όπω είπε και ο κύριο Λαφράγκα, τώρα διαπραγματευόμαστε με, το τη Μερκοσούρ και είναι εδώ η κυρία Γκαλίνα, επικεφαλή των διαπραγματεύσεων και με το Μεξικό. Και έχουμε ολοκληρώσει και τι συμφωνίε με τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Κάποια τεχνικά ζητήματα μένουν να μεταφραστούν για την συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Λόγω τη αλλαγή για το επενδυτικό δικαστήριο είναι ίσονο σημασία και ελπίζω πω θα μπορέσουμε και αυτήν τη συμφωνία να σα την υποβάλουμε το, την Άνοιξη. Η συμφωνία με το Βιετνάμ καθυστερεί στη μετάφραση και όχι εξαιτία μα, αλλά λόγω του ότι οι Βιετναμέζοι θέλαν λίγο περισσότερο χρόνο για ορισμένα ζητήματα. Ελπίζουμε πως η μετάφραση αυτή θα ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα και σίγουρα θα θέλαμε και αυτή να σας την υποβάλουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν το έχουμε ξεχάσει πάντως, αυτό είναι βέβαιο. Όπως ξέρετε, παίρνουν, παίρνει κάποιο χρόνο η μετάφραση. Για την προστασία των δεδομένων και την καταλληλότητα. Ε, τώρα ολοκληρώνουμε στην Επιτροπή την πρόταση που θα συζητήσουμε μαζί σας και με τα κράτη-μέλη όπως γνωρίζετε είναι λεπτό, ε, λεπτή εξέβρεση ισορροπίας ανάμεσα στο εμπόριο και στα στοιχεία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρηση στη συμφωνία με την Ιαπωνία. Δεν είναι ανοιχτή, δηλαδή όλα. Υπάρχει ρήτρα αναθεώρηση και η συνάδελφο Γιούροβα συζητά με τους Ιάπωνες φίλου μας για την καταλότερα τη προστασία ε, των δεδομένων. Έχουν ε, αυστηρές νομοθεσίες παρόμοιες με αυτές που θα αρχίσουν να ισχύουν τον Μάιο και μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Ιαπωνία γι' αυτό, πράγμα που θα διευκολύνει το εμπόριο. Με σεβασμό στην... στα πρότυπά μας. Οι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε υπάρχουν στη συμφωνία, δεν αποκλείονται. Για το θέμα τη φοροδιαφυγή και τη διαφάνεια είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Συνεργαζόμαστε με του Ιάπωνε στο ΝΟΣΑ και στο G20 όπου η συνεργασία είναι ικανοποιητική και θα συνεχίσει να είναι. Το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης ή του περιβάλλοντος όχι. Βεβαίως είναι υποχρεωτικό και μπορεί να ενισχυθεί, αλλά δεν προβλέπονται κυρώσει. Δεν προβλέπονται κυρώσει στα πρότυπα συμφωνία. Όπω το γνωρίζετε όμω όλοι και έχω έρθει επανειλημμένα εδώ και έχω συνομιλήσει και μεμονωμένα με κάποιους από εσά, εργαζόμαστε ώστε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κεφάλαιο αυτό και την εφαρμογή του. Κυρώσεις είναι μια επιλογή. Η συζήτηση αυτή λοιπόν δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ρήτρα αναθεώρησης μέσα στη συμφωνία. Κυρία Αρένα, ρωτήσατε γιατί... Α, φύγατε. Για το θέμα της αρχιτεκτονικής, στην, έχουμε την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία και διαπραγματευόμαστε χωριστά για την προστασία των επενδύσεων. Υπάρχει διαχωρισμός εκεί. Για το γενικό θέμα της αρχιτεκτονικής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση από το Συμβούλιο ακόμα. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές. Θα συζητηθεί και στο επόμενο Συμβούλιο. Κύριε Ντάτμοφ, ναι, βεβαίως είναι ευκολότερο για δύο χώρες να έρθουν σε μια συμφωνία από ότι μια χώρα και μια, ένα σύνολο άλλων. Ευκολότερο είναι να συμφωνήσουμε εγώ και εσείς, ίσως πάλι όχι, από ότι αν είμαστε περισσότεροι για να συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι όμως βέβαια η ποιότητα της συμφωνίας και με την Ένωση 28 χώρες είμαστε ακόμη και η Ιαπωνία είμαστε μαζί το 30% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Φοβερές δυνατότητες ανοίγονται. Μια χώρα, οποιαδήποτε μία μόνη χώρα που θα διαπραγματευτεί με την Ιαπωνία μόνη της θα βρει μια συμφωνία βέβαια, αλλά θα είναι λιγότερο ε, εκτεταμένη. Και βεβαίως ε, η διαπραγματευτική ισχύς πίσω από όλα αυτά είναι ε, μεγαλύτερη όταν έχουμε μια αγορά και εκπροσωπούμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων. Προστατεύουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ε, συμφωνία με την Ιαπωνία. Περιλαμβάνονται περισσότερες ε, γεωγραφικές ενδείξεις από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Θα υπάρξουν λίγες μόνο, νομίζω μόνο τέσσερις που θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Θα μπουν σταδιακά δηλαδή, αλλά για τις υπόλοιπες θα είναι η ίδια διαδικασία, οπότε και μάλιστα ολοκληρώνεται ο κατάλογος στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει λοιπόν περίοδος ε, σταδιακής ένταξης ορισμένων γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά όλες οι άλλες και αυτές που αναφέρατε όπως η Παρμεζάνα θα, θα, θα περιλαμβάνονται και θα προστατεύονται όπως κάνουμε πάντοτε. Γιατί η φαλαινοθήρια ε, βεβαίως είναι ένα φρικτό πράγμα που συμβαίνει με τις φάλαινες και το έχουμε αυτό σαφώς τονίσει στους Ιάπωνες φίλους μας. Η εμπορική φαλαινοθυρία απαγορεύεται στα κράτη-μέλη, ε, όλα τα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες σε διεθνή φόρα και έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές στην Ιαπωνία και στους υπόλοιπους ότι όλα τα είδη φάλαινας προστατεύονται από την οδηγία Habitat. Και οι εισαγωγές και εξαγωγές απαγορεύονται. Και γι' αυτό και δεν το περιλάβαμε στο στην εμπορική συμφωνία, γιατί δεν είναι αντικείμενο εμπορίο. Εμείς συμμετέχουμε σε διάφορα φόρα ε, για να πάψει αυτή η φρικτή συνήθεια. Νομίζω πως αυτές ήταν πάνω κάτω οι ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Και έπειτα υπάρχει μια αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού που είναι σημαντική. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι πολύ ευρεία και όχι πολύ λεπτομερής και συγκεκριμένη. Όμως εργαζόμαστε σε αυτό το πνεύμα προς αυτή την κατεύθυνση με τους Ιάπωνες στο εμπόριο αλλά και στους άλλους τομείς διευκολύνουμε το εμπόριο στα, για τα αγαθά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και αυξάνουμε τη συνεργασία όσον αφορά το πρασίνισμα των οικονομιών μας ε, και στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας αλλά και στο πλαίσιο της ε, συνεργασίας που έχουμε με αυτή τη χώρα να θέλουμε πολλά και ανταλλάσσουμε καλές εμπειρίες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις ερωτήσεις σας και θα επανέλθουμε για να σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, εξ αρχής παρακολουθεί αυτέ τι διαπραγματεύσει και η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι θα συνεχίσουμε να θέτουμε ερωτήσει μέχρι το τέλο τη διαδικασία, Μέχρι ότου, δηλαδή, να χρειαστεί να λάβουμε την τελική μας απόφαση για αυτή την ε, συμφωνία. Βασιζόμαστε λοιπόν στην εργασία μαζί σα. Να μην σα εκπλήξει παρακαλώ, αν σα θέσουμε και άλλε ερωτήσει. Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. So, now we switch to another interesting... Uh, Περνάμε σε μια άλλη ενδιαφέρουσα περιοχή του πλανήτη καθώς ασχοληθούμε με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μας με τη Μερκοσούρ. Ε, όπως γνωρίζετε είχαμε, σκοπεύαμε αρχικά ε, στο πλαίσιο ε, τη πολιτική διάθεση ε, του ΠΟΕ τον Πουένο Άρη να ολοκληρώσουμε τι σχετικέ διαπραγματεύσει με του Μερκοσούρ. Δεν τα καταφέραμε τελικά. Οπότε θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ω προ τι διαπραγματεύσει μα. Και γι' αυτό εδώ καλώς ορίζω θερμά τους εκπροσώπους εδώ της Μερκοσούρ και ιδιαίτερα την αυτού εξοχότητα τον κύριο Γκαούτο Βίλμαν πρέσβη της ε, παραγωγή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και ο προεδρεύων αυτή την περίοδο της Μαρκοσούρ. Από την πλευρά της Επιτροπής έχουμε την ίδια Γαλλή τη διαπραγματευτικής ομάδας, την κυρία Σάντρα Καλίνα, πολύ γνωστή εδώ μεταξύ μας. Ναι, σας διακρίνω ότι στο βάθος Ε, και γνωρίζω ότι είναι κανένα μακρηγορή, οπότε επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να την παρακαλέσω να εστιάσει μόνο στα σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους, ε, γιατί για πρώτη φορά προσέρχομαι στην δική σας ε, επιτροπή. Ας περάσω όμως τώρα στο Λοιπόν, είχαμε την συζήτηση και τη συνάντηση στο Buenos Aires όπου καταφέραμε να συζητήσουμε και τα ζητήματα και να σημειώσουμε πρόοδο ε, και να σας αναφέρω συγκεκριμένα ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους επιτύχαμε πρόοδο και επίσης η ανταλλαγή απόψεων έγινε σε μεγάλο βαθμό γιατί υπήρξαν και συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο ε, όπου διεφάνει ότι πράγματι ερχόμαστε τώρα σιγά σιγά στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης και αυτό είναι θετικό ε, γιατί μετά από αυτήν την τελική αν θέλετε ευθεία των διαπραγματεύσεων θα παραμείνουν πολύ λίγες εκκρεμότητες. Άρα λοιπόν σε αυτά τα κύρια ζητήματα θα ήθελα να περιοριστώ. Η Μερκοσούρ ε, ολοκλήρωσε, ενοποίησε αν θέλετε την πρότασή της, οπότε έφτασε δηλαδή το 90% στον Buenos Aires, πράγμα το οποίο προφανώς είναι ευπρόσδεκτο και νομίζω έχουμε φτάσει στο 90% απελευθέρωση δηλαδή ε, όπως προτείνεται από την πλευρά της Μερκοσούρ και αυτό είναι σημαντικό. Όπως σας είπα τώρα, έχουμε σημειώσει πρόοδος ε, ότι φορά τα επιμέρους ε, έγγραφα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά εκείνο για τις υπηρεσίες αλλά και σε ό,τι αφορά το εμπόριο αγαθών. Σημαντικές λοιπόν πρόοδες σε σχέση με αυτά τα δύο έγγραφα και το πιο σημαντικό είναι ότι οι επικεφαλείς ε, διέταξαν όλα τα κείμενα αυτά, στο σύνολό τους δηλαδή. Και το κάναμε αυτό στον Buenos Aires, έτσι ε, ώστε να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς το τι παραμένει ως εκκρεμότητα. Και βέβαια σεβαστήκαμε επίσης ε, και τον ευαίσθητο χαρακτήρα των επιμέρους ζητημάτων, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των ε, προτέρων πόσες δυσκολίες μπορούν να προκύψουν από μία και μόνη λεπτομέρεια. Τώρα, μετά από εκείνη τη συνάντηση, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι και οι δύο πλευρέ να συνεχίσουμε τι εσωτερικέ μα διεργασίε, αλλά να προβούμε και μετά και σε μια νέα συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο έτσι ώστε να περάσουμε ακριβώς στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Ε, το σημαντικό θα είναι βέβαια σε αυτή την τελική ευθεία η πρόσβαση στην αγορά, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ορισμένα στοιχεία του κανονιστικού πλαισίου τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτά λοιπόν πολύ σύντομα, ενημερωτικά. Ο πιο σημαντικός τομέας, στον οποίο ακόμα παραμένει σημαντική δουλειά που θα πρέπει να γίνει σε ε, τεχνικό επίπεδο, παρότι έχουμε δει δηλαδή το ε, πακέτο, είναι ε, κανόνες προέλευσης, τα rules of origins. Εδώ έγινε πολύ κατατοπιστική συζήτηση, γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι τα ζητήματα εκείνα τα οποία χρήζουν, αν θέλετε, περισσότερε προσπάθειε και όπου θα χρειαστεί δηλαδή να κάνουν περισσότερε προσπάθειε οι υπουργοί μα για να γεφυρώσουμε εδώ τι διαφορέ μα. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο των αγαθών, να πούμε ότι πραγματικά σε ό,τι αφορά το base rate φτάσαμε σε μια τελική συμφωνία και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί ακριβώ καταδεικνύει ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση τη διαπραγμάτευση με βάση το χρονοδιάγραμμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε ε, και την εγκατάσταση. Ε, αυτό το σημείο αλλά και οι ναυτιλιακέ μεταφορές αποτελούν σημεία προτεραιότητα για μα και υπήρξαν εδώ στοιχεία τα οποία αφορούν και τις ε, τηλεπικοινωνίες. Εδώ το Μερκοσούρ είχε θέσει κάποια ζητήματα και ε, καταφέραμε βέβαια εμείς απλώς να διταχθούμε και τα καταφέραμε οπότε ε, είναι καλό το γεγονό ότι υπήρξε πρόοδο σε ό,τι αφορά τι τηλεπικοινωνίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, οι εμπειρογνώμονε θα πρέπει ακόμα να συνεχίσουν τη συζήτηση, γιατί ακόμα ε, η συζήτηση είναι προκατακτική θα έλεγα. Τώρα σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και εδώ επιτύχαμε ε, πολύ ικανοποιητική πρόοδο, λίγες εκκρεμότητες παραμένουν ε, επί των οποίων θα χρειαστεί να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις, αλλά Όπως ε, είπα ήδη και στο παρελθόν, αυτό το κεφάλαιο ε, δεν ήταν το δυσκολότερο, καθώς αυτή η εταιρεία κοσούλ δηλαδή ενδιαφέρεται πραγματικά και ίδια πάρα πολύ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, Ένα τομέα τώρα στον οποίο υπάρχουν, υπάρχει ακόμα κάποια διάσταση απόψεων, δύο βασικά τομείς είναι καταρχήν το TBT, όπου έχουμε το σύντημα των αυτοκινήτων, το, το παράτημα δηλαδή σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων φυσικά, εδώ σας αναφέρω τα πιο σημαντικά ζητήματα και από εκεί και μετά έχουμε ε, την ιδιωτική ε, διοκτησία. Ε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, θυμάμαι ότι απεστάλλεται μια επιστολή από την πλευρά των βουλευτών και πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι εδώ προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα όσα έχουμε προβλέψει σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση, τα γνώσουμε και οτιδήποτε άλλο έχουμε προβλέψει δηλαδή και σε επίπεδο FDM. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα την γενετική ιδιοκτησία, εδώ βέβαια εμπίπτουν και τα, των γεωγραφικών ενδείξεων και υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν αλλά αφορούν κυρίως σε ονομασίες. Και συνεχίζουμε την εργασία, την εξαιρετική εργασία που είχαμε με τους εταίρους μας από τη Μερκοσούρ. Λίγα δηλαδή ακόμα στοιχεία παραμένουν για να επιληθούν σε ό,τι αφορά τι γεωγραφικέ ενδείξει. Αυτά δεν θέλω να σα απασχολήσω με περαιτέρω λεπτομέρειε. Είμαι στη διάθεσή σα για περαιτέρω ερωτήσει και όπω σα είπα, στις 30 του μήνα προβλέπεται να λάβει η χώρα επόμενη υπουργική διάσκεψη έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε και αυτή την τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Αλαφράνκο, εισηγητής. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι χαίρομαι που η κυρία Γκαλίνα μας υπενθύμησε ότι ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων ε, ε, συμπεριέλαβε και συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο και ήρθαν εδώ οι αρμόδιοι επίτροποι. Ε, η δική μου πολιτική ομάδα, ε, τα άκουσα όλα αυτά, συζητήσαμε την Επίστροπο Μάλστρομ, μας δώσανε όλες τις πληροφορίες για το θέμα αυτό. Αυτό που λείπει είναι ο Επίτροπος Γεωργίας που, αφορά, που είναι υπεύθυνος για ένα πολύ ευαίσθητο τομέα των διαπραγματεύσεων δεν ήρθε εδώ για να μα δώσει εξηγήσει ε, από το Δεκέμβριο. Ε, ο πρόεδρος Γιούκερ έκανε κάποιε δηλώσει ε, στο Στρασβούργο στην ομιλία για την κατάσταση τη Ένωση. και είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τον τελευταίο λόγο σε αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε. Προφανώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο πολύ σωστά για όλη τη διαδικασία. Επομένω, λείπει ε, μία εξήγηση από τον Επίτροπο των Αρμόδιων για τα Γεωργικά, τον κύριο Χόγκαν. Ακούσαμε την κυρία Γκαλίνα. Ε, οι προβλέψεις που είχε θέσει η Κομισιόν, ε, γιατί δεν τηρήθηκαν ε, μέχρι τον Δεκέμβριο. Ποιο στέει για την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, το Μερκοσούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαπραγματευτική διαδικασία στον Buenos Aires Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από το Μερκοσούρ ε, μία αύξηση 1% ε, και των γεωργικών μεταποιημένων προϊόντων. Ε, αν δεν το είχε ζητήσει αυτό θα είχε κλείσει γρήγορα η διαπραγμάτευση. μην ξεχνάτε τη σημασία της υπουργική διάσκεψης που θα γίνει. τι παίζεται ακριβώς, θέλουμε να ξέρουμε Και με βάση τις ε, τελευταίες προφορίες που μας έδωσε η Γκαλίνα, επιφυλάσσομαι να ξαναπάρω το λόγο. Πάντως θέλω να εκφράσω ήδη το σεβασμό για την πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει σε αυτό το πλαίσιο. Τελευταίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έστειλε μία επιστολή του κ. Κατάινεν, ε, της Μάστρομ και του κ. Χόγκαν, έχει δεσμευτεί για τα θέματα πρόσβαση στην αγορά. Ε, φαντάζομαι αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Πολλά ερωτήματα. Πρώτα θα μιλήσουν οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, τηρήστε το χρονοδιάγραμμα 1,5 λεπτό κατά κεφαλήν. Ο κύριος Ντάντε είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπω στο ψητό κατευθείαν και θα ζητήσω από την κυρία Γκαλίνα κάποια πράγματα θα τη ρωτήσω για αυτή την συμφωνία. Για πρώτη φορά διάβασα το κείμενο και το είδα συνολικά. Θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία. Καταρχάς, ε, διαγωνισμοί την εθνική μεταχείριση των Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών την, έχουμε, την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά. Έχουμε εξασφαλίσει όλες τις εγγυήσεις για τους διαγωνισμούς σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μάλλον τα έχουμε εξασφαλίσει εγγυήσεις σε ομοσπονδιακό και τώρα έχουμε περάσει στο υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, σε πολιτιακό δηλαδή επίπεδο, για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Μας είπατε, κυρία Γκαλίνα, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θέλω να καταλάβω πόσο βαραίνει ε, το θέμα της συνύπαρξης πολλαπλών γεωγραφικών ενδείξεων. Έχουμε αναγνωρίσει πολλές γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, έχουν αναγνωριστεί μάλλον ήδη. Και εμείς είμαστε ετοιμένοι να γνωρίσουμε τις δικέ τους γεωγραφικέ ενδείξει. Υπάρχουν όμω μερικέ φορέ ε, προβλήματα ονομάτων. Οικονομικά, πόσο μετράνε αυτές οι γεωγραφικέ ενδείξεις, α πούμε, έτσι, για να καταλάβουμε, ας πούμε, γιατί έχουμε παρόμοια ή ταυτόσιμα ονόματα κτλ. Ε, ένα σημαντικό τομέα κατ' είναι ο τομέας ε, των υποδημάτων. Εμείς έχουμε, αντιμετωπίζουμε το φάσμα πολύ ψηλών δασμών για να μπούμε στο Μερκοσούρ, στην αγορά του Μερκοσούρ, όπως στην Αργεντινή Φερρυπίν. Πολύ ψηλοί δασμοί για τις δικέ μας εξαγωγέ. Ε, για τους κανόνες ε, καταγωγής. Καταγωγής συζητούνται ακόμα το θέμα, αυτό το θέμα για τα κλωστοκοδοτικά και τα υποδήματα. Και τέλος, τι θέλω να καταλάβω. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, θα υπάρξει η περίπτωση διαφυγής όλη αυτή η δουλειά που έγινε. Αν δεν φτάσουμε σε συμφωνία, όπως προβλέπετε, δεδομένων και των προεκλογικών εκστρατιών ε, στην, ε, στις χώρες. Έχουμε μία ε, πόρτα διαφυγής. Έχουμε πλάν B. Ο κ. Σταμπάτη. η ε, ε, συμφωνία με τη Μερκοσούρ προφανώς είναι ιδιαίτερα πρόσδεκτη. Γνωρίζουμε το τι συμβαίνει με τέτοιου είδους συμφωνίες. Εδώ όμως φτάσαμε σε ένα ορόσημο και βρισκόμαστε κοντά στην επιτυχή έκβαση αυτή τη διαπραγμάτευση. Η χρονική συγκυρία είναι κατάλληλη, καθώ οι Αμερικάνοι έχουν απομακρυνθεί λίγο. Οπότε εμεί μπορούμε να αποτελέσουμε το νέο επίκεντρο, αν τη δραστηριότητα σε σχέση με τη συνεργασία με την κυρία. Με, με, τη, με, με Αλλά μόλι τώρα άκουσα από την κυρία Μαστρόμ ότι ε, ουσιαστικά έχει ρουστικοποιηθεί η σχετική συμφωνία. Αλλά ε, θέτω και εγώ μαζί με τον κύριο Σαραφράγκα το ερώτημα ποια είναι, ποιες είναι οι εκκρεμότητες. Η ε, έκθεση δηλαδή που μας έκανε η κυρία Γκαλίνα ε, ουσιαστικά μας δείχνει ότι υπάρχει εδώ, υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά ακόμα βρισκόμαστε μέσω διαπραγματεύσεων, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Και επίσης ε, ένα ζήτημα που αναφέρθηκε είναι ειδικότερο αγροτικό τομέα. Εξαιρετικά σημαντικό. Ε, σε σχέση με αυτό το τομέα θα ήθελα να ξέρω πιο συγκεκριμένα πού βρισκόμαστε στι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Σαράντσοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ θα ήθελα να θαρρύνω την Επιτροπή να αξιοποιήσει την όθηση ε, που έχει δοθεί σε αυτέ τι διαπραγματεύσει όντω ώστε να τι οριστικοποιήσουμε, γιατί ε, παλαιότερα πραγματικά δεν γίνονταν ε, αρκετά γρήγορα. Τώρα λοιπόν έχουμε την κατάλληλη όθηση, α την αξιοποιήσουμε. Γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή τα επιθετικά και τα αμυντικά συμφέροντα τη Ένωση. και γι' αυτό θα ήθελα να να την καλέσω να επιταχύνει τη διαδικασία. Γιατί δεν είμαστε οι μόνοι στους οποίους ενδιαφέρει η περιοχή της Μαρκούσου. Η κυρία Γκαλίνα τώρα εξέθεσε ε, τις ε, κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις διαπραγματεύσεις, αναφέρθηκε εκεί ε, στους κανόνες καταγωγής, οπότε θα ήθελα να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, θα ήθελα να τη ζητήσω λοιπόν να μας ε, δώσει λίγες παραπάνω πληροφορίες. Ε. Και επίσης ε, ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε εδώ θα έχουμε δυνατότητα να ανοίξουμε ένα μπουκάλι σαμπάνια ώστε να γιορτάσουμε την επιτυχή έκβαση. Αλλά εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ίσως θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια εξαιρετική συνεδρίαση τη Επιτροπή μα, έτσι ώστε να καλέσουμε εδώ και του συναδέλφου συμμετέχοντε στι διαπραγματεύσει, όπω ανέφερε ήδη ο κ. Φράγκα. Κάτι τώρα ακόμα σε γενικότερες γραμμές ε, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε είναι ενδεχομένως η δυνατότητα του να έχουμε ε, συγκεκριμένες ε, μελέτες σε ό,τι αφορά ευαίσθητους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι δηλαδή έκθεση σε ό,τι αφορά μια συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά εκθέσεις σε ό,τι αφορά επιμένους κλάδους και τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου σε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Σάντρα Γκαλίνα για αυτέ τι ε, πληροφορίε που μα έδωσε ω προ το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσει. Ε, και θεωρώ και εγώ πω ε, η ποιότητα θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε τέτοιου είδου συμφωνίε και όχι προφανώ στο χρονοδιάγραμμα, καθώ η συμφωνία θα έχει και σημαντικέ επιπτώσει στη ζωή των ανθρώπων. Τώρα, αναφερθήκατε με θετικά λόγια στο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση λοιπόν με αυτό, μπορεί να μας διαβεβαιώσει η Επιτροπή ότι δεν θα χρησιμοποιείται γλυφοζάτη στις εκτάσεις εκείνες όπου θα καλλιεργούνται εξαγωγικά προϊόντα που θα προορίζονται δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δηλαδή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αναλάβει τη δέσμευση εντός ε, πέντε ετών να καταργήσουμε τη χρήση της κλειφοζάτης και πρόκειται βέβαια για ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα διασφαλιστεί αυτή η απαγόρευση και στο πλαίσιο ε, του εμπορίου με τις λατινοαμερικανικές χώρες. Ε, ποια είναι δηλαδή τα προϊόντα ε, που χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες. Γιατί βέβαια θα πρέπει να διασφαλίσουμε εδώ και την προστασία των οικονομικών πολιτών, της υγείας τους. Δεύτερο ερώτημα πώς ε, θα ρυθμίσετε το κανονιστικό πλαίσιο ε, σε σχέση με τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή πώς θα διασφαλίσετε την, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις όπως αυτές που είχαμε, όπως για παράδειγμα αυτά που είδαμε με τα Panama Papers. Δεν θέλουμε δηλαδή σε καμία περίπτωση αυτή η συμφωνία να οδηγήσει τελικά ή να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την φορά που φύγει. Σα ευχαριστώ. Αν Μαρή Voorzitter, ehm, in het voortgangsrapport naar aanleiding van de laatste onderhandelingsroe. Ευχαριστώ. Ε, στην έκθεση πρόοδο μας είπατε ότι σχεδόν έχει υπάρξει συμφωνία για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα θέλω να γνωρίζω αν η Κομισιόν μπορεί να μας πει ποια κεφάλαια παραμένουν ανοιχτά και μήπως ήταν υπερβολικά φιλόδοξη. Έπειτα μιλάτε και επίση για μια ρήτρα όπου λέγεται ότι πρέπει να συνεργαστούμε κατά των κλιματικών αλλαγών. Αυτό ας πούμε λέγεται στην συμφωνία με την Ιαπωνία. Και θα προσθεθεί και αυτό ε, ε, και στις συμφωνίες με το Μερκοσούρ κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και προηγουμένως. Μπορεί η Κομισιόν να μας εγγυηθεί ότι η συμφωνία με τη Μερκοσούρ δεν θα οδηγήσει στην αύξηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντισταθεί σε αυτά τα μέτρα που μπορεί να επιφέρουν βλάβη στο περιβάλλον, ακόμα και αν είναι οι αντιπροσωπεύουν ε, συγκεκριμένη επένδυση. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και μέσα από τις επενδύσεις και έπειτα θα ήθελα να ζητήσω αυτές οι ενδιάμεσες εκθέσεις να είναι λιγότερο σύντομες γιατί θα έπρεπε να χρησιμεύουν για να ενημερώνουν τους πολίτες και να ε, επικρατεί διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Αντρικένα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτές οι διαπραγματεύσεις, όπως γνωρίζουμε για αυτή την εμπορική συμφωνία συνεχίζονται εδώ και δύο δεκαετίες ε, σχεδόν. Έχουν τελματοθήσει οι διαπραγματεύσεις και μπορούμε να σε συγχαρούμε για μια πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά... Ε, γνωρίζουμε ότι τον Οκτώβριο έγινε πρόταση Ε, για κατάργηση συγκεκριμένων αδασμών και τελικά όμως οι χώρες του Μερκοσούρ είπαν ότι ε, ήταν πολύ χαμηλή η προσφορά και τελικά την αποσύραμε θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά βοηού. Κυρία Γκαρλίνα, αλλά υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα και όχι μόνο το βοηού κρέας, όπως η πρόσβαση για τα γεωργικά και τα βιομηχανικά αγαθά, όπως αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και θέματα προέλευσης γεωγραφικών ενδείξεων και ευκαιριών για τις ε, υπηρεσίες ε, ναυσιπλοείας. Ερώτησή μου λοιπόν απλή. Είστε αισιόδοξοι ότι οι διαπραγματεύσει θα ολοκληρωθούν φέτος. Ο κύριος Γουάς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, στην, στην, στην, ε, στην Επιτροπή στην αντιπροσωπή Ευρωπαϊκή Ένωση με Βραζιλία. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε κοινέ αξίε, γλώσσα, ταυτότητα, κοινέ ε, δημοκρατικέ αρχέ και αρχέ του κράτου δικαίου. Και θα προβώ στην ερώτηση Με το τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων και τι ε, πολιτικέ εξελίξει που ε, επέρχονται. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε πω υπάρχει κάποιο διαπραγματευτικό άνοιγμα για συμβαστική συμφωνία κοινωνία στους ευαίσθητους τομείς που όλοι γνωρίζουμε ώστε να καταστεί δυνατό να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Καρολή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη Χιλή, η σχετική συμφωνία δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Θα υπάρξει δημοσίευση αντίστοιχη και αυτή με τη Μερκοσούρ για λόγου διαφάνεια. Επίση, κάτι δεν άκουσα σχετικά με την προστασία των επενδυτών. Υπάρχει κάτι σχετικά ε, στη συμφωνία. Ε, και αν ναι, ε, ποια είναι η άποψη των εταίρων μα από τη Μερκοσούρ σε σχέση με το ICS. E Επίση, η συμφωνία αυτή θα είναι σε τα πλάσια, για να το πούμε έτσι. Υπάρχει μεν ρήτρα αναθεώρηση, αλλά από εκεί και μετά Ε, ε, ποια είναι η θέση των εταίρων μας σε ό,τι αφορά και την ενδεχόμενη επιβολή ε, κυρώσεων από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τα πρώτα εργασία έχουν ήδη κυρωθεί. Σε ό,τι αφορά τη φοροαποφυγή υπάρχει σχετικό κεφάλαιο και επίση ο ρόλο τη οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Και εδώ έχει προβλεφθεί κάτι επίση σε ό,τι αφορά τι αγροτικέ δραστηριότητε σε σχέση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία αποκλείσαμε αυτούς ε, τους ε, ιδιαίτερα ευαίσθητους ε, τομείς. Κάτι τέτοιο θέλετε να κάνετε και σε σχέση με την Μερκοσούρ. Ευχαριστώ. Είμαι το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Γκαλίνα για την προσπάθεια που κάνει, αλλά και τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Εγώ νομίζω πως ακόμη μια φορά πρέπει να επιμείνουμε για τη στρατηγική σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Νότια Αμερική η υπογραφή μια καλή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρο. Όμως με ανησυχεί το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω πως θα ήταν απαραίτητο να φτάσουμε σε καλή συμφωνία και μάλιστα πριν να ξεκινήσει η προεκλογική διαδικασία στη Βραζιλία και να εμποδίσει την ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας. Όμως με ανησυχεί αυτό που άκουσα, κυρία Καλίνα, τόσα πολλά εκκρεμή ζητήματα. Πώς ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε συμφωνία το Δεκέμβριο. Υπήρξε κάτι κοντεύατε να επιτύχετε τη συμφωνία και κάνατε πίσω μετά. Συνέβη κάτι. Γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμα σε κρεμότητα. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς θα εγγυηθείτε τον έλεγχο των φυτογενομικών από πλευράς της Βερεσλίας ε, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Βραζιλία. Ποιος εγγυάται το φυτογενομικό έλεγχο, έπειτα θεσμική δομή ε, για την ε, συγκεκριμένο έλεγχο και για τη διαφάνεια. σαν οι διαπραγματεύσεις το 1997. Είναι παράδεκτο παράδεκτο και είναι ντροπή που δεν έχουμε κάνει ακόμα τη συμφωνία. Δεν πρέπει να αρχίσει ούτε μία μέρα να μην περάσει ακόμα χωρίς να δημοσιευθεί αυτή η εντολή. Και έπειτα, με τόσο καιρό που έχει περάσει μέχρι σήμερα, με όλες τις προόδους που έχουν σημειωθεί στην πνευμορική πολιτική και για να βελτιωθεί η, το εύρος και το πεδίο εφαρμογή ε, αυτών των συμφωνιών, θα έπρεπε η εντολή να μεταβληθεί. Θα έπρεπε να ενταχθεί εκεί μια ρήτρα αναθεώρησης, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να επιτύχουμε ε, στο, τον, την συμφωνία που επιθυμούμε, χωρίς να έχει μετατραπεί και η αρχική εντολή. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά καλωσορίζω τον επικεφαλής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Μερκοσούρ και τον εισηγητή της ΑΦΕΤ, τον κύριο Ασίσκου, και του δίνω το λόγο. agradecer as informações que nos foram prestadas pela Galina, mas eu creio Ευχαριστώ την κυρία Γκαλίνα για, τις, ε, για τα όσα μας ε, είπε ενημερωτικά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, αλλά έχουμε φτάσει σε μια ε, κέρια φάση τώρα των διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι Υπουργοί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τελικά το αν θέλουν μια συμφωνία ή όχι ε, με τη Μερκοσούρ. Έχω ακούσει δηλαδή επανειλημμένα στο παρελθόν την κυρία Γκαλίνα, αλλά και την Επίτροπο. Ε, και να μας ενημερώνουν επανειλημμένα σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό που ακούμε κάθε φορά είναι ότι βρισκόμαστε στο παραπέντε των εισαγωγικών ε, πριν από την ε, οριστικοποίηση της ε, συμφωνίας, αλλά δεν φτάνουμε ποτέ σε αυτήν την οριστικοποίηση. Άρα λοιπόν, η δική μου εντύπωση είναι ότι σε αυτή την ιστορική χρονική συγκυρία η πλευρά της Μερκοσούρ έχει κάνει πολύ πιο συγκεκριμένα βήματα ε, προς την οριστικοποίηση, προς τη σύναψη της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι αντίθετο με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Γιατί τώρα δηλαδή ε, το πρόβλημα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την επίτευξη προόδου ε, έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στην πλευρά της Μερκοσούρ. Άρα λοιπόν εδώ τίθενται μια σειρά από ε, σημαντικά ζητήματα, αλλά το κυριότερο από αυτά είναι θέλουμε τελικά ένα τέτοιο σύμφωνο ή όχι. Ε, και νομίζω πως ε, αυτό το σύμφωνο έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για από άποψη οικονομική, αλλά σε ό,τι αφορά και γενικότερα τα ζητήματα ανάπτυξη και τα εμπορικά ζητήματα. Αλλά πέραν αυτών των εμπορικών δηλαδή και οικονομικών ζητημάτων υπάρχει και μια διάσταση πολιτική και στρατηγική η οποία ακριβώς ε, ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να λάβουμε αυτή την απόφαση να, να, να φτάσουμε στη σύναψη τη συμφωνίας. Άρα λοιπόν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία ε, με τη Μερκοσούρ ουσιαστικά είδαμε να μεταβάλλονται οι τοποθετήσει, δηλαδή από το να, είναι ε, πιο, ε, να, να ακολουθούν μια προστατευτική ε, στάση, οι εταίρε μα τη Μερκουσούρ έχουν αρχίσει να ανοίγονται, να θέλουν να προβούν σε ένα σύμφωνο και τελικά εμεί είμαστε εκείνοι που δεν θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Όμω δεν είμαστε μοναδικοί εναλλακτικοί για αυτέ τι χώρε. Έχουν και άλλου σημαντικού εταίρου ανά τον κόσμο, του οποίου θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία. Άρα λοιπόν θεωρώ πω αποτελεί σφάλμα με άγνωστε συνέπειε προ το βανόν το να μην προβούμε στη σύναψη μια τέτοια συμφωνία και να αφήσουμε η Μερκοσούρ να στραφεί ε, προ άλλε περιοχέ του κόσμου. Άρα λοιπόν ε, ε, σε εμά έγκυται τελικά το να αποφασίσουμε. Επιθυμούμε ή όχι συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Και όχι μόνο σε σχέση με τα ζητήματα τη Βραζιλία, αλλά και με βάση δηλαδή, τα δικά μα χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να δούμε ε, αν πραγματικά τώρα θα, ε, θα, θα επιτύχουμε τη σύναψη τη συμφωνία ή όχι, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να συναυθεί μετά στα επόμενα χρόνια. Η συγκυρία πολυ δυσκολο να διαβιβαστεί αυτό είναι σωστή. Οπότε θα ήθελα να διαβιβαστεί αυτό το μήνυμα. Ότι δηλαδή πραγματικά σε αυτή τη φάση εμεί, η ευρωπαϊκή πλευρά, είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να κάνουμε τα τελευταία ε, βήματα. Και στο μέλλον κανείς δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί αν δεν φτάσουμε σε μια ε, συμφωνία το γιατί δεν μπορέσαμε μέσα στο 2018 σε μια τέτοια χρονική ε, συγκυρία ε, να μην φτάσουμε σε μια συμφωνία μόνο και μόνο λόγω 30 εκατομμυρίων τόνων βόηου κρέατος. Πραγματικά θα πρέπει να αναλάβουμε μια ισχυρή δέσμευση προκειμένου πράγματι να φτάσουμε στη σύναψη αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φίλμαν, έχετε το λόγο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μας, για το Μερκοσούρ, είναι προνόμιο το να μπορούμε να μιλάμε σε αυτή την Επιτροπή και προσωπικά ε, πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση, το άκουσα με απόλυτη προσοχή, με ευχαρίστηση άκουσα τη θέση της κυρίας Γκαλίνα που κάνει μια δουλειά ε, όλο ζήλο και ενθουσιασμό. Μου άρεσε επίσης η παρέμβαση, οι παρεμβάσεις μάλλον των Ευρωβουλευτών. Ε, θαυμάζω τις γνώσεις τους και την δέσμευσή τους. Μου άρεσαν τα λόγια που είπαν, ε, που δείχνουν ότι αναγνώριζουν τη σημασία αυτής της συμφωνίας. Ε, υπόθηκε πολλές φορές πόσο σημαντικό θα είναι αυτή η συμφωνία όχι μόνο για, τις δικές μας, για τη δική μας και τη δική σας περιφέρεια, αλλά για όλες τις χώρες ε, που θέλουν πολυμερές εμπόριο που να βασίζεται σε κανόνες. Ε, όλες αυτές οι χώρες θέλουν ε, το Μερκοσούρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάσουν σε μια καλή συμφωνία. Αυτό σημαίνει ισορροπημένη συμφωνία και παράλληλα με ένα αποδεκτό επίπεδο φιλοδοξίας, ούτω ώστε το σύνολο των παραγωγικών μας δυνάμεων ε, να βρει σε αυτό το εργαλείο μία ευκαιρία για να αναπτυχθεί και να γιγαντωθεί. Θέλουμε ε, μία συμφωνία ε, με μία καλή προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γεωργικά. Δεν έχει νόημα αλλιώ. Πώς γίνεται για τη χώρα μου, την Παραγουάη, ε, που η γεωργία είναι το 25% του ΑΕΠ ετησίως, ε, και είναι το 85% της προσφοράς μας για τις εξαγωγές και δίνει τόσο πολλές θέσεις απασχόλησης στον ενεργό πληθυσμό. Για το Μερκοσούρ αυτές οι διαπραγματεύσεις σημαίνουν ε, και μια ειδική πρόκληση. Είναι οι πρώτες διαπραγματεύσεις που θα μας επιτρέψουν καλύτερη ενσωμάτωση και θα επιτρέψουν και στο Μερκοσούρ να ενσωματωθεί καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία. Πιστεύουμε ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται η δυνατότητα να καταφέρει ε, να πετύχει καλύτερες προτιμήσεις ε, που αφορούν 263 εκατομμύρια ανθρώπους σε τομείς βασικούς για τη βιομηχανία της και θα της επιτρέψει να παγιώσει την ανάπτυξή της, να αυξήσει τις θέσεις και να ε, σκοτώσει το φάσμα της ύφεση. Έγινε η συνάντηση στο Buenos Aires, ε, η συνάντηση αυτή υψηλού επίπεδου, η οποία αναφέρθηκε εδώ. Το Mercosur έδειξε ότι είναι αποφασισμένο με συγκεκριμένες προτάσεις ε, που φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων μας. Ε, σύντομα θα γίνει μια νέα συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο, εδώ στις Βρυξέλλες, όπου το Μερκοσούρ ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει το ίδιο ενδιαφέρον να πετύχει μια δίκαιη και λογική συμφωνία, κάτι το οποίο νομίζω επιθυμούμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με ρωτάτε αν είναι φιλόδοξη ότι θα τελειώσουμε φέτο. Είμαστε τον Ιανουάριο. Ε, έχουμε μήνε μπροστά μα. Αλλά ε, δράζεται κάπου αυτή η αισιοδοξία. Σε αυτή τη φάση έχουμε καταφέρει όλα τα θέματα να τα ρυθμίσουμε εκτός από τα δύσκολα. Ε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά τα καλά λόγια τα αξίζει όλη η ομάδα. Πολλοί άνθρωποι δούλεψαν για αυτό το θέμα, για αυτή τη συμφωνία και θα ήθελα να το πω αυτό δημόσια. Να ξεκινήσω καταρχάς με το ποιο στέει. Γιατί νομίζω ότι είναι καλό ε, να ψάχνουμε να βρούμε το φταίχτη. Δεν θα απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Είναι λάθος προσέγγιση. Σε μία διαπραγμάτευση όλοι και οι δύο πλευρές συμπασχετώσει προσπαθούμε να φτάσουμε ε, σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Το να λέμε εγώ φταίω, εσύ φταίς κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό πνεύμα και η σχέση με τους εταίρους του Μερκοσούρ ούτως ή άλλως είναι πολύ καλή, δεν βασίζεται σε αυτό το ποιο στέει. Θα μπω και σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να πω μια τελική γενική φράση που, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβετε την πολιτική σημασία του τι κάνουμε. Άκουσα διάφορα να λέγονται εδώ στην αίθουσα. Να σα πω λοιπόν το εξή. Ε, ας πάμε στις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε εθνική μεταχείριση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ρήτρα. Περιμένουμε μια σαφή προσφορά που θα ικανοποιεί την ευρωπαϊκή πλευρά. Γιατί οι εταίροι του Μερκοσούρ όταν δημοσιεύονται μια συμφωνία δημοσίων προμηθειών μεταξύ του πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ του. τι μπορούν να προσφέρουν μεταξύ του. Τώρα για το ομοσπονδιακό επίπεδο, ο κατασκευαστικό τομέα λείπει, λείπουν κάποια στοιχεία ε, σε ό,τι αφορά τι ΔΕΚΟ. Σεβόμαστε απόλυτα ότι θέλουν να σεβαστούν, να διατηρήσουν κάποιες ΔΕΚΟ. Για το υπομοσπονδιακό επίπεδο πρέπει να δούμε λιγάκι περί τίνο πρόκειται. Δεν έχουμε φτάσει κάτι συγκεκριμένο για τι γεωγραφικές ενδείξει. Επίτευγμα. Το μείζον επίτευγμα είναι αυτό, γιατί Θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία, TRIPS συν 23, TRIPS 23 μάλλον plus, πιο συγκεκριμένα. Τώρα τι δημιουργεί πρόβλημα. Το γεγονός ότι πολλοί έφυγαν από την Ευρώπη. Ε, το θέμα δεν είναι ότι πήγαμε στην ε, Ιαπωνία. Πολλά, πολλά, δηλαδή εμπορικά σήματα φύγανε. Δεν πήγαν στην Ιαπωνία, αλλά πήγαν στον Καναδά κτλ. Τώρα πρέπει να βρούμε ε, λύσεις για αυτές τις συγκρούσεις, για αυτές τις διαφορές. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αντιπαραθέσεων πριν διαμορφώσουμε άποψη. Πάντως δεν υπάρχει βασικό θέμα γιατί υπάρχει βούληση για να τελειώσουμε με αυτό σε ό,τι αφορά τα υποδήματα, την, την υπόδηση και άλλα θέματα που λείπουν. Η απελευθέρωση για κάποιους τομείς στην ευρωπαϊκή προσφορά, διαβάστε το, βασιζόμαστε στην αμοιβαιότητα, έτσι. Δεν απελευθερώνουμε τα δερμάτινα υποδήματα στην Ευρώπη αν δεν απελευθερώσετε και εσείς το δικό σας τομέα. Θα είναι δύσκολο για σας, γιατί ο, ο, ο, ο όγκος εξαγών που έχουμε στο Μερκοσούρ είναι μηδέν. Επομένως, μπορείτε να βάλετε κάτι εκεί πέρα, μια και λείπει εντελώ. Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στην προσφορά σας του Μερκοσούρ, σκεφτείτε ότι βασιζόμαστε στην ε, αμοιβαιότητα, ειδικά για τα ευαίσθητα θέματα. Είμαστε στο μέσον ή στο τέλος. Πού είμαστε. Θέλω να το πω ε, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει plan B. Γιατί το υπενηχθήκατε ορισμένοι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια στρατηγική εξόδου, δεν υπάρχει plan B, πρέπει να το τελειώσουμε αυτό, πρέπει να τελειώσουμε αυτή τη συμφωνία και τώρα, γιατί αλλιώς θα κλείσει το παραθυράκι ευκαιρίες. Τι πρέπει να εξετάσουμε. Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά. Για μας κάτι που δεν είναι ικανοποιητικό ακόμα είναι το αίτημα ε, που έχουμε για τα αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων δεν μας έχετε απαντήσει. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μας δώσετε κάποια στιγμή κάποια απάντηση. Ε, το Μερκοσού θα μας δώσει, γιατί είναι βασικό στοιχείο της συμφωνίας για μας. Το ίδιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, όπως ανέφερα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι το τμήμα αυτής της πυρηνικής συμφωνίας, ε, στο, στον πυρήνα είναι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το 1% που τέθηκε στο, στο τραπέζι το Δεκέμβριο δεν συμπεριλάμβανε τα γαλακτοκομικά. Για τα άλλα θέματα. Κεφάλαιο TSD. Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ φιλόδοξο. Κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε. Δεν θα σας απογοητεύσει το αποτέλεσμα, γιατί είχαμε καλή υποδοχή των τιμάτων μας από τους εταίρους. Φόρο αποφυγή, ξέπλυμα χρήματος. Οι χώρες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στον περίφημο μαύρο κατάλογο που υπάρχει, να το πούμε αυτό, και παράλληλα έχουμε ε, το στοιχείο της φορολογικής συνεργασίας ε, στη συμφωνία. Το, αν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα εναπομείναντα θέματα. Είμαστε στην εξής φάση. Τώρα χρειάζομαστε κάποια πολιτική δέσμευση. Τα τελευταία που θέλω να σας πω είναι ότι σας άκουσα όλους και με χαρά βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένας έτσι πολιτικός ενθουσιασμός για αυτή τη συμφωνία που είναι πολύ σημαντικό για να διαπραγματευτεί. Να βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον το οποίο ξεπερνάει ε, τη μερκαντιλιστική προσέγγιση και ανταλλαγή. Αυτό που είπε ο κύριος Αζής είναι σωστό. Κανένας δεν έχει ε, καλές απαντήσεις. Εάν πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί δεν την τελειώσαμε τη συμφωνία τώρα, ας πούμε. Είναι δύσκολη η χρονική στιγμή, ειδικά για το βόλιο κρέας. Ε, οι γεωργοί μας ξέρουν ε, το θέμα του Brexit και μπορεί το βόλιο της Ιρλανδίας να επηρεαστεί. Δεν είναι καλύτερη χρονική στιγμή να μπούμε στη συμφωνία για το βόλιο. Υπάρχουν στιγμές που μετράμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να πετύχουμε. Και διάφορα μέτρα που μας δίνουν την ε, βεβαιότητα ότι η συμφωνία θα είναι καλή, αυτό, σε αυτά εστιάζουμε. Ε, SPS, ε, επενδύσεις. Καταρχάς δεν έχουμε τις επενδύσεις για τη συμφωνία αυτή. Μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θα υπάρξει τέτοιο κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Για το SPS, φυτογενομικά μέτρα. Σας τονίζω ότι θα είναι θαυμάσιο κεφάλαιο ε, με αμοιβαιότητα. Έχουμε ένα από τα κεφάλαια που θα, αν υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο θα είμαι περήφανη, θα είναι αυτό. Τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε γεωργική συμφωνία χωρίς τα φυτεογειονομικά. Η πολιτική, πραγματικό το πολιτικό πλαίσιο είναι σημαντικό. Ε, έχω μία έκκληση. Εγώ είμαι τεχνοκράτης, κάνω ό,τι μπορώ για να πιέσω τα πράγματα και με την υποστήριξη των εταίρων φτάνω σε μία ιονή πολιτική συμφωνία. Ε, υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν πήγαν πολύ μακριά. Έχω πολύ καλούς εταίρους που μπορούν να με βοηθήσουν, ειδικά με το κείμενο ε, σημειώσαμε πρόοδο, αλλά τώρα για το θέμα της πρόσβασης στην αγορά χρειαζόμαστε μια πολιτική ένδειξη, πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές. Γιατί τα εναπομείναντα θέματα πρόσβασης στην αγορά, στην αγορά για μας είναι τα αυτοκίνητα, απογοητευτικό θέμα και απαιτούν πολιτική επιλογή από το Μερκοσούρ. Και εμείς χρειαζόμαστε από πλευρά μα μια πολιτική βούληση για το θέμα των αυτοκινήτων και τη πρόσβαση στην, αγορά των αυτοκινήτων. χρειάζομαι βοήθεια πολιτική. Αλλιώ θα πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση και να απαντηθεί το ερώτημα τελικά γιατί δεν θέλουμε αυτή τη συμφωνία. Πάντως αυτή η συμφωνία θα είναι πολύ σημαντική γεωπολιτικά. Αλλά εγώ δεν έχω την πολιτική απάντηση να σα δώσω. Είμαι απλή τεχνοκράτη. Αλλά έχετε και επιρροή, ε. Κύριε Σαλαφράγκα. Eh. Μάλιστα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή σας και για τον άποψή τους για αυτή την κατάσταση των διαπραγματεύσεων που νομίζω σαφώς αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ ε, με όλο το σεβασμό που δείχνω και με την αρχική μου εισήγηση για την εργασία που κάνει η κυρία Καλίνα, νομίζω ότι Αυτή τη στιγμή πολιτικός ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι που λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι το Ευρωκοινοβούλιο ε, στην Επιτροπή ε, και είναι δική μας υπόθεση αν θέλουμε να δώσουμε σημασία ή όχι και είναι λογικό το να ρωτάμε γιατί δεν επιτυχάνονται οι στόχοι. Έχω θέσει τρεις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε και δεν πήρα καμία απάντηση. Ρώτησα αν ο γύρος στο υπουργικό επίπεδο ε, αν έγινε προσπάθεια για τα γεωργικά προϊόντα ε, για 1% παραπάνω είναι προφανές πως έγινε κάτι τέτοιο. Έπειτα σημαντική ερώτηση για το αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε γραπτός για να διαβελτιώσει την ε, προσφορά της είναι προφανές ότι Υπήρξε αυτή η θέληση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επιθυμητό να κάνουν λοιπόν και οι χώρε του Μερκοσούρ μια προσπάθεια για να ανταποκριθούν στι δικέ μα ανησυχίε. Και κύριε Πρόεδρε, νομίζω πω έχουμε κοινή αίσθηση εδώ στην Επιτροπή μα ε, ότι ο χρόνο είναι ένα παράγοντα που παίζει καθοριστικό ρόλο. Η Επίτροπος Μάλστρο μας εξήγησε πριν από λίγο ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ισχύω τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Οι διαδικασίε είναι γρήγορε, ταχείε και όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν συναυθεί αυτή η συμφωνία σύντομα, η έναρξή τη θα αναβληθεί και επαόριστα. Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε λοιπόν ε, την ουσία με τα επουσιώδη, γιατί ε, έτσι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω πως όλοι έχουμε την ευθύνη να πιέσουμε οι εθνικές κυβερνήσεις, γιατί κάποιες φορές υπάρχουν κάποια κρατημέλη τα οποία πραγματικά καθυστερούν τη διαδικασία. Ε, ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να καταστήσουμε σαφές πως το Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά επιθυμεί την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Γιατί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που έχει ανοίξει. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους για αυτή την συζήτηση και ευχαριστώ και τον πρέσβη που ήταν εδώ και τώρα περνάμε στο επόμενο μας σημείο που είναι το υπαριθμό 25. Πρόκειται για την έκθεση για την παρακολούθηση Έχουμε τη Είχαμε κάποιες ομάδες παρακολούθησης, μία για τη Χιλή, Συζητήσαμε με τον πρέσβη της διαπραγματεύσεις με την Χιλή. Δεν έγινε τίποτα σημαντικό. Για την Ιαπωνία μόλις κάναμε τη συζήτηση με τον επικεφαλ... επικεφαλής. Νότια Ασία. Υπήρξε μια ομάδα παρακολούθησης δραστηριοτήτων με μια αντιπροσωπεία ε, μελών του Πακιστανικού Κοινοβουλίου και θα τους ε, συναντήσω νομίζω αύριο. Ούτε εδώ έχει, γίνει, έχει υπάρξει κάτι το σημαντικό και υπήρξε και μια ομάδα παρακολούθησης ε, για τη συμφωνία για τις επενδύσεις και για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Um, uh, Canada will meet on the για τις, 24 ε, θα, συναντηθούμε με τον πρέσβη του Καναδά και για τις σχέσεις με τον Καναδά που τώρα πάμε στο η φάση εφαρμογής της Συμφωνίας ΣΥΤΑ. Η Ήρμα θέλει να πει κάτι για τη Χιλή. Μισό λεπτό και, η ομάδα παρακολούθησης για το Μαρόκο θα συναντηθεί επίσης στις 24 και θα ε, μιλήσει για την κατάσταση πρόοδου των διαπραγματεύσεων καθώς και για τα αγαθά που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Χιλή. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε να πω μόνο για ενημέρωσή σας ότι έγινε μια συνεδρίαση της ομάδας ε, παρακολούθησης μετά από την έναρξη του γύρου διαπραγματεύσεων. Έγινε η πρώτη συνεδρίαση λοιπόν και μιλήσαμε για το χρονοδιάγραμμα ε, και για το ποιε είναι οι φιλοδοξίες του Ευρωκοινοβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαμε εγκρίνει το ψήφισμά μας ε, το Σεπτέμβριο Πιστεύω πως ε, πληρώνται οι όροι για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε σε καλή συμφωνία. Συγκεκριμένα αυτή τη βδομάδα γίνεται ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων και θα μπούμε περισσότερο στην ουσία. Να τονίσω ότι υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση από και από τις δύο πλευρές και γι' αυτό και αναζητούμε θέσεις όσον αφορά το επενδυτικό δικαστήριο για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά και έναν μηχανισμό που βασίζεται, όπου θα περιλαμβάνονται κυρώσει όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών αυτά και να αναγνωρίσουμε ότι είναι πρόσδεκτο το ότι δημοσιεύθηκε η εντολή του Συμβουλίου δύο μήνες αφού συνέφθη ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια και δεν έχει δημοσιευθεί εντολή για το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε με αυτή την έκθεση σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε των ομάδων παρακολούθηση. Περνάμε στο σημείο 26, ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 2016. Εισηγητή εδώ είναι ο κύριο Λούνε, αλλά θα τον αντικαταστήσει σήμερα ο κύριο Ταρπάτ παρακαλώ. Ευχαριστώ. το συγγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου, ο οποίο ε, χρειάστηκε τελευταία στιγμή να αποχωρήσει. Και έτσι, τελευταία στιγμή μου ζήτησε και εμένα να πάρω το λόγο αντί αυτό. Οπότε θα διαβάσω προ το μόνο το κείμενο. Ε, χαιρετίζω το γεγονό ε, ότι ε, η Επιτροπή μπορεί να τοποθετηθεί επ' αυτής της έκθεσης της ετήσιας δραστηριότητας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, και γνωρίζουμε πως πρόκειται για ένα ίδρυμα το οποίο βέβαια διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για μακροπρόθεσμα στρατηγική σημασία σε επενδυτικά έργα και τα οποία συμβάλλουν βέβαια στην πρόοδηση των συμφωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι το 90% των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λαμβάνει χώρα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η τράπεζα δραστηριοποιείται ε, στο πλαίσιο των υπολείπων 10% εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ε, μέσω και τη αντίστοιχη εντολής που έχει για ε, δράσεις στην αλοδαπή Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή είναι σημαντικός χρηματοδότης και σε άλλα μέρη ε, του κόσμου. Άρα λοιπόν ε, θεωρώ σημαντικό ε, το ότι η λόγω έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται και σε αυτές τις δραστηριότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς ε, οι, αυτές οι επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδιαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι τέτοιο βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει εν λόγω αυτέ οι ε, επενδυτικέ δραστηριότητε ε, τη τράπεζα να ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Επίση, ε, γίνεται μία αναφορά ε, στην έκθεση ε, στην προτεραιότητα που δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, η καλύτερη δηλαδή χρηματοδότηση τέτοιου είδους επιχειρήσεων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση, η πρόσβαση σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Η τράπεζα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίζει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να εντοπίσει και να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Θα πρέπει δηλαδή να δρομολογήσει ορισμένα προγράμματα ακριβώ διευκόλυνση αυτή τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να είναι πιο ε, προσβάσιμε οι χρηματοδοτήσει τη ε, και να συμβάλλουν στι ε, παγκόσμιε αλυσίδε παραγωγή αξία, προωθώντα ταυτόχρονα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο του externalizing, θα ήθελα επίση να προτείνω και την υποστήριξη της δυνατότητας άμεσων ξένων επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χώρους της Ασίας, για παράδειγμα. ένα ακόμα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ο σημαντικός ρόλος που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων ως προς την καταπολέμηση των γενεσιουργών αιτιών της μετανάστευσης. Κατά τελευταία χρόνια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της μαζικής ανάπτυξης ε, στα δικά μας σύνορα και στο μέλλον η πίεση αυτή ενδεχομένως θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Λόγω δηλαδή και των ε, δημογραφικών εξελίξεων αλλά και λόγω των περιφερειακών σειράξεων των Άρα λοιπόν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωση να συνεργαστούμε με τις χώρες εταίρους μας έτσι ώστε να επιτύχουμε στις εν λόγω χώρες ε, μια σταθερότερη και πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εδώ μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο η τράπεζα, ε, παρέχοντας όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και την απαραίτητη έμπειρο γνωμοσύνη προς επιχειρήσεις και επενδυτές έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερε και να αξιοποιηθούν οι φυσταμένε εμπορικέ και επενδυτικέ ευκαιρίε που υπάρχουν σε αυτέ τι χώρε. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θέλει να ε, τονίσει ο συναδελφό Ελούνε. Αναμένω προφανώ ε, με ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδέλφων και την οικοδομική συνεργασία που θα κάνουμε στο πλαίσιο των τροπολογιών που θα ακολουθούν σε σχέση με αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Πρόεδρο. Ο λόγο τώρα στου οικειώδει εισηγητέ για το ΕΛΚ Ραμόνα Μανέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Το κείμενο που ετοιμάσε ο εισηγητής είναι βάση, καλή βάση, για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στο εξωτερικό και την αύξησή τους, ειδικά για την ενσωμάτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παγκόσμια αξίδα αξιών. Ε, είναι θετικό και το μέσο διευκόλυνσης ε, για τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Ε, είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι η, χρηματοδότηση. αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες τις ρίζες της μετανάστευσης, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα οικονομικά κίνητρα για ανάπτυξη και τα ανθρωπιστικά θέματα, αλλά και την ε, ανάπτυξη των υποδομών θα παρακολουθώ το θέμα με ενδιαφέρον και προσοχή και θα υποβάλω και τροπολογίε. Ε, θέλω ευκολότερη πρόσβαση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, στη χρηματοδότηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υποστηρίξει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο εξωτερικό και μέσω του προγράμματο του προγράμματος χρηματο, ε, διευκόλυνση του εμπορίου. Θα πρέπει οι δραστηριότητε τη τράπεζα να εφηγραμμιστούν με τους στόχους ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Ε, είναι ο οικονομικός βραχίωνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω θα πρέπει να είναι ε, σε φάση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση πρέπει να υποστηρίξουμε τι τις επιχειρήσει και κυρίω τι επενδύσει του, ειδικά στην κινέζικη αγορά. οι Ευρωπαϊκέ επιχειρήσει πρέπει να είναι πιο παρούσες στο εξωτερικό και ειδικά στην Ασία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χρειαζόμαστε γρήγορη προσαρμογή της τράπεζας στις τρέχουσες ε, διεθνείς προκλήσεις και στη μετανάστευση ε, και έναν ενεργό και στατικό ρόλο της τράπεζας για να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της μετανάστασης, όπως είπε και ο εισηγητής. Η τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη ε, της, την, στρατηγική για το εμπόριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβει υπόψη τι ισχύουσε εμπορικέ συμφωνίε αλλά και τι μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε ε, υποστηρίζοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του εξωτερικού, ε, δίνοντας προτεραιότητα στις χώρες που έχουν ήδη εμπορικές συμφωνίες, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και να τις υποστηρίξει και η τράπεζα βέβαια. Ε, είμαι σίγουρη για την καλή συνεργασία με τον εισηγητή και θα προσπαθήσω και εγώ όσο μπορώ να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Από το φιλελεύθερους η Πατρίτσια La Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Η Επιτροπή μας κάνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2016. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη δουλειά που κάνει η Τράπεζα ε, και τα δάνεια, το σύνολο των δανείων που δίνει εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 έδωσε ε, το 16 8,4 εκατομμύρια, το προηγούμενο το 7,8. η ε, προτεραιότητα για το 16 της τράπεζας είναι η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και η καταπολέμηση των βασικών αιτίων της ε, μετανάστευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι δύο διακυβέρματα βασικά για την παγκόσμια κοινότητα και η μετανάστευση προς την Ευρώπη ε, δεν ήταν πολύ δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικό πρόβλημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όσο σήμερα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο άξονε προτεραιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικοί που και αλληλένδετοι. Η γνωμοδότηση του εισηγητή είναι σωστή και είναι προ κατεύθυνση και ω κοιόδη των φιλελεύθερων θα ήθελα να συμπληρώσω την έκθεση με τα εξή στοιχεία. Θα προτείνω βεβαίω και τροπολογίε. Πρώτον, Είμαι πεπισμένη ότι οι δραστηριότητε τη τράπεζα σε διεθνέ επίπεδο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια ε, βιώσιμη και στρατηγική ανάπτυξη, δηλαδή σε αρμονία με τι πολιτικέ τη Ένωση και βεβαίω θα πρέπει να δώσει στον Ευρωπαίο επενδυτή ευκαιρίε στο εξωτερικό. Προ αυτήν την κατεύθυνση συμφωνώ με την ιδέα του εισηγητή για τι δραστηριότητε τη τράπεζα ε, που θα πρέπει να είναι πολύ πιο έντονε στην Ασία, κυρίω ε, στην Ινδία και στην περιοχή Αζεάν Επίσης, ε, στην άμεση γειτονία μας, που είναι η Αφρικανική Ήπειρο, προτεραιότητα και αυτή θα πρέπει να είναι. Λυπάμαι που η περιοχή των ΑΚΕ, ε, η περιοχή ΑΚΕ είναι αυτή που έχει τα λιγότερα χρήματα, παρά το γεγονό ότι έχουμε πάρα πολλά προγράμματα και έργα εκεί. Ε, θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω για τα, τα project ε, για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί ο οικονομικό ιστό και να δώσει ε, διεξόδου σε επιχειρήσει και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ξέρουμε ότι συχνά είναι δύσκολο να καταλήξουν αυτά τα έργα. Δεν καταλήγουν στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα project που λειτουργούν και να εντοπίσουμε και να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές. Σε ό,τι αφορά τις χώρες ΑΚΕ και τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να αξιολογούμε την επίπτωση των ε, project που γίνονται σε τοπικό επίπεδο ε, και, για το, και κατά πόσο επωφελεί για τις τοπικές κοινότητες. Οι συμφωνίες Κοτονού μας ε, συνδέουν με τους εταίρους μας ΑΚΕ. Θα πρέπει το 2020 να ανανεωθούν. Θα ήθελα ο μηχανισμός που υπάρχει για τη χρηματοδότηση project εκεί να μην τροποποιηθεί, ε, ως προς το πώς λειτουργεί, γιατί ανταποκρίνεται καλά στην ανάγκη χρηματοδότησης των δικαιούχων. Τέταρτον, η πρωτοβουλία για την οικονομική αντοχή που ξεκίνησε το 2000, ανθεκτικότητα για το 2006, για να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης, είναι κινείται προ σωστή κατεύθυνση, προ σωστό άξονα. Πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ικανότητα της ε, τράπεζα να παίρνει ρίσκα και να διαχειρίζεται το ρίσκο για διάφορα τέτοιου τύπου project και αν χρειαστεί να ανανεώνονται ε, τα project αυτά, γιατί μετά από πέντε χρόνια πούμε, μπορεί να χρειαστεί να ανανεωθούν. Επίση, οι ανταλλαγέ ε, απόψεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και των ε, Ευρωβουλευτών να είναι πολύ πιο συχνέ κτλ. για να ασκούμε σωστό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί να μην δημιουργήσουμε και μια ομάδα εργασία, α πούμε, πολύ πιο περιορισμένη σύνθεση για το θέμα αυτό. Ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Σάντερ ε, Λούνας ε, για αυτήν την ε, έκθεση. Πραγματικά αναφέρει μία σειρά από σημαντικά ζητήματα, ζητήματα τα οποία πραγματικά άξιζαν να αναφερθούν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί και μας ενδιαφέρουν όλους. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρει σωστά ε, την ε, ανάγκη της ένταξης των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις γενικότερες δράσεις εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Και αυτό είναι σωστό βέβαια. Γιατί οι αρμοδιότητε για αυτήν την εξωτερική πολιτική είναι κατοχυρωμένε και στις συνθήκες. Αλλά ταυτόχρονα ναι, εδώ σα. Ε, θα ήθελα να σας προτείνω να συμπληρώσετε και την ε, αναπτυξιακή πολιτική. Ε, γιατί οι δράσεις ακριβώς της ε, Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να κατευθυνθούν και προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του 2030. Και με αυτό τους λέω ότι δεν θα πρέπει να προωθεί εξαγωγές, για παράδειγμα, στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και επενδύσεις στην, στις υποδομές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ε, περιφερειακές ε, και τοπικές υποδομές ε, εμπορίου, εμπορικών ροών. Και αυτό αφορά ειδικότερα στις παραγράφους 5 και 6. Δηλαδή, στις περιοχές ιδιαίτερα όπου ο επενδυτικός κίνδυνος είναι αυξημένος και οι επενδυτές ακριβώς για αυτό το λόγο διστάζουν να προβούν σε επένδυση, εκεί θα μπορούσε η Τράπεζα Επενδύσεων να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Ειδικότερα δηλαδή αυτό αφορά την Αφρική η ε, Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναπτύξει όλο ένα και περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη ως προς την αξιολόγηση των κοινωνικοπολιτικών επιπτώσεων αυτών των επενδύσεων. Και γι' αυτό λοιπόν η συγχρηματοδότηση ε, κοινών project θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή συγχρηματοδότηση από την Τράπεζα ε, από κοινού με άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Γιατί είδαμε για παράδειγμα ε, πόσο λανθασμένα ήταν κάποια project ε, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εξόριξη λιγνίτη σε ορισμένε ανατολικοευρωπαϊκέ χώρε. Κάτι τέτοιο είναι εσφαλμένο. Και θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε ποιε είναι οι δυνητικέ συνέργειε τη συγχρηματοδότηση από διαφορετικέ αναπτυξιακέ τράπεζε εδώ. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το εργαλείο τους ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Τώρα σε ό,τι αφορά την ε, παράγραφο 4 αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες, ε, οι επενδυτικές ε, των επιχειρήσεών μας στην Κίνα. Πράγματι τέτοιου είδους επενδύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη από μια δημόσια τράπεζα επενδύσεων, οι επιχειρήσει μπορούν να προβαίνουν από μόνο του επενδύσει εκεί που το επιθυμούν. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αξιοποιείται η τράπεζα επενδύσεων προκειμένου να ε, ε, εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις αυτές, για παράδειγμα μεσοπαίδιο, οι οποίες ακόμα βρίσκονται σε φάση ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση πάντως ε, χαίρομαι για την συζήτηση και την εμβάθυνση αυτών των ζητημάτων που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ, λέω. Πρόεδρος. Κύριος Σταρτμαντ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομα και σαφερό Με βάση τον εισηγητή εδώ στην παράγραφο 1 διαβάζω ότι το 10% ε, των, ε, της ε, νολικής, των συνολικών δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αφορά περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την τελευταία φορά που έριξα εγώ μια ματιά υπήρχε και ένα σημαντικό ποσοστό πέραν αυτού που κατευθύνθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω, ε, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί ε, ως έχει ή ε, προτίθεται να την επαναξετάσει. Δεύτερο ζήτημα. γύρω στο 16% που αντιστοιχεί σε 9 δισεκατομμύρια ευρώ ε, αναλογούσαν τελευταία φορά που έριξα μια ματιά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από επιχειρησιακής λοιπόν άποψης, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το, το, χάσμα που θα προκύψει στο ό,τι αφορά το μετοχικό τη ε, ε, μερίδιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μετά τον Brexit. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Δεν μα μένει πολύ χρόνο μέχρι τι και μισή, οπότε δίνω το λόγο κατευθείαν στην Επιτροπή και μετά στην Τράπεζα Επενδύσεων για να απαντήσει στα ερωτήματα. Πολύ σύντομη θα είναι η Επιτροπή. Οι λειτουργίε τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν αποκτήσει μεγάλη ορατότητα. Ε, χαιρόμαστε που μιλάει και λέει την άποψή τη και αυτή η Επιτροπή εδώ. Ε, τη βασική ε, Επιτροπή την έβγαλε η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή, που είναι η Επιτροπή Ελέγχων των Προπολογισμών. Για τι εξωτερικέ δραστηριότητε. Ε, ε, υπάρχει το, με βάση το ELM το οποίο έχει αναθεωρηθεί πέρυσι και λαμβάνουμε μεταξύ άλλων υπόψη και τους βασικούς λόγους μετανάστευσης ε, σε θέματα εξωτερικού δανεισμού. Μάλιστα. Πολλές ερωτήσεις τώρα απευθύνθηκαν προς την ίδια την τράπεζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Να αντιδράσω στις τελευταίες ε, δύο ερωτήσεις. Για το μερίδιο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πόσο κομμάτι από το κεφάλαιό της το δίνει για δανειοδοτικέ επιχείρησει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση που έχουμε είναι η εξή. Το 10% των δραστηριοτήτων μας ε, αφορά ε, δραστηριότητε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπε και η Κομισιόν, ξέρετε ότι οι πολιτικέ διαπραγματεύσει για την εξωτερική δανειστική εντολή έχουν οριστικοποιηθεί. Αυτό είναι το ELM. Ε, οριστικοποιήθηκε στι 7 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια, του Κοινοβουλίου και η Τράπεζα επίση ετοιμάζει μια νέα πρόταση ε, να υπάρχει δηλαδή μία ε, θηγατρική τράπεζα, ευρωπαϊκή τράπεζα, ε, σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη. Να υπάρχουν επίσης διάφορες υπηρεσίες αναπτυξιακές που θα συνεργάζονται για να ενισχύσει το, την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει project εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η τράπεζα με την υποστήριξη βεβαίω για να υποστηρίξει τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που το Ούτω ή άλλω αυτό το έχουμε στο μυαλό μα όταν επεμβαίνουμε είτε στο εξωτερικό, παρεμβαίνουμε στο εξωτερικό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω θα έχουμε ένα φορέα ειδικό, μία θηγατρική εντό τη τράπεζα που θα μα επιτρέπει να παίρνουμε περισσότερα ρίσκα. Αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο και στο παρελθόν. Αν λαμβάνουμε ούτω ώστε με αυτόν τον τρόπο να προωθούμε και να δημοσιοποιούμε περισσότερο τι δραστηριότητέ μα. Ε, για να υπάρχει μια καλύτερη κατανομή ε, στο χαρτοφυλόκιό μας ανάμεσα στις δανειοδοτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Τώρα, για την επίπτωση του Brexit. Είναι προφανές ότι μετά το Μάρτιο του 2019 η τράπεζα θα χάσει ένα μεγάλο μέτοχο. Θα χάσουμε το 16% του κεφαλαίου μας, των μετοχών μας. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Υποστηρίζουμε φυσικά τις ε, ομάδες ε, διαπραγματεύσεων όταν χρειάζεται. Όταν ε, υπάρχει κάποιο σημείο στη διαπραγμάτευση του Brexit που συνδέεται με την τράπεζα. Φυσικά για την τράπεζα το, το γεγονός ότι το δημοψήφισμα έδωσε αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό και θα έχουμε μεγάλες απώλειες εμείς στην τράπεζα σε κεφάλαιο. Θα δούμε μετά το Μάρτιο 2019 πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κλείσαμε τη συζήτηση. Ε, για να υποβάλουμε τροπολογίες έχουμε μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. 6 η ώρα το απόγευμα. Πάμε πάρα αυτά. Στο 27 έχουμε 6 λεφτά. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας για τη συνεργασία και αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνιακά θέματα. Ο κύριος Μόστερ ε, τον κύριο Κασπάρη. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ο κύριος Κασπάρης, δεν συγγνώμη που δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν, μου ζήτησε να παρουσιάσω αυτή την έκθεση εξ ονόματός του και προς χάρη ακρίβειας θα διαβάσω το σημείωμά του. Ο εισηγητής θα ήθελε να ζητήσει από την Επιτροπή ήταν να εγκρίνει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία για τη συνεργασία και την αμοιβαία ε, αρρωγή σε τελωνιακά θέματα που υπεγράφηκε στις 3 Ιουλίου 2017. Γενικό στόχος της συμφωνίας είναι να αναπτύξει και να εντατικοποιήσει τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνεργασία στα τελωνιακά θέματα ανάμεσα στην Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία. Θεσπίζει συγκεκριμένα νομική βάση για πλαίσιο συνεργασίας που στόχο έχει να εξασφαλίσει την αλυσίδα ανεφοδιασμού καθώς και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή της ε, τελωνιακή νομοθεσίας και να προβλέψει και να αποτρέψει την ε, διάρρηξη της, την ρήξη μάλλον, την παραβίαση της ε, τελωνιακής νομοθεσίας εν ώψη της μελλοντική διαπραγμάτευσης για Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών όπου εγκρίθηκε ως ιδέα από το Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2017, αυτή η συμφωνία μπορεί να σημαίνει μια εμβάθυνση του ίδιου όριμου της όριμης εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο εταίρους, δημιουργώντας μια πιο φιλική, ένα πιο φιλικό περιβάλλον για το εμπόριο. Ε, συνεργασία επιτευχθεί και με την Νότια Κορέα, το Καναδά, το Χονγκ Κόνγκ, τη ΣΥΠΑ, την Ινδία, την Κίνη και την Ιαπωνία. Ο εισηγητή λοιπόν πιστεύει πως είναι κατάλληλη στιγμή για σύναψη τέτοια συμφωνίας με έναν αξιόπιστο και στενό συνεργάτη όπως η Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των Σοσιαλιστών σύντομα η Καρολίνα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα είμαι, γιατί πραγματικά έτσι κι αλλιώς σε σχέση με αυτό το ζήτημα το Κοινοβούλιο έχει μόνο ε, δικαίωμα σύμφωνη νόμη. Σημαντικό πάντω ε, παραμένει να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μα με την Ζηλανδία. Οπότε δεν νομίζω πω υπάρχει κάποιο λόγο ε, για αμφιβολίε. Οπότε κατά τη δική μα άποψη, ναι, είμαστε υπέρ του να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο Πρόεδρο. Υπάρχουν άλλα σχόλια, υπάρχουν σχόλια από την Επιτροπή. Όχι καλός. Οπότε ανακοινώνω απλώς την ε, προθεσμία για την υποβολή ανθρωπολογιών. Α, ο κύριος Ντάρτμαθ, το λόγο, παρακαλώ. Νομίζω πως ε, θα ήθελα να αναφέρω ουσιαστικά δύο, α, δύο Ε, καταρχήν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε μια εμπορική συμφωνία, προτού δηλαδή προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 1973-1974 με τη Νέα Ζηλανδία. Ε, ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το, η Νέα Ζηλανδία έχει μια ε, συμφωνία εμπορική με την Κίνα. Οπότε δεν υπάρχει μια βιώσιμη ελπίδα του να συναυθεί μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα στο σε μέλλον εντάξει, με βάση αυτά τα δύο στοιχεία μπορεί κανεί να λύσει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, αλλά εντάξει, δεν θα επεκταθώ παραπάνω και σα ευχαριστώ για την μόνη σα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. 30 Ιανουαρίου στι 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την αποβολή τροπολογιών. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, 28 της ημερήσια διάταξη στα διάφορα, το αγαπημένο μου σημείο που τη ημερήσια διάταξη. Α, βλέπω κάτι υπάρχει. κύριο Δάρπαου. Ναι, ένα σημείο τη διαδικασία για να το λάβετε υπόψη σα. Σήμερα το πρωί διακόψαμε γύρω στις 12, λίγο νωρίτερα, ε, ενώ ε, σήμερα το απόγευμα ε, ήταν τόσο φορτωμένη η Μερσέντα που χρειάστηκε να ξεκινήσουμε και νωρίς ε, και παρόλα αυτά, πολλοί από τους προσεκριμένου ομιλητές μας, ε, παρότι ήρθαν από μακριά, δεν είχαν δυνατότητα να πούν όσα ήθελαν να πούν. Οπότε εκείνο που θα ήθελα να ζητήσω από τη γραμματεία της Επιτροπής είναι να, να ε, διαμορφώνουν λίγο πιο σοβαρά την ημερήσια διάταξή μας, ε, έτσι ώστε το πρωί να μην είναι τόσο άδεια και το απόγευμα να μην είναι τόσο φορτωμένο. Πρόεδρος. Ναι, ε, το πρόβλημα είναι όμως ε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιο, ποια από τα μέλη ε, θα είναι παρόντα και πότε. Γιατί αν μπορείτε να μου εγγυηθείτε την παρουσία των μελών, τότε ναι, μπορώ να σας πω ακριβώς. Εκεί θα μπορούμε να υπολογίσουμε το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό που σημαίνει συνήθως δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη, δεν ζητάνε όλα τα μέλη τον λόγο και ορισμένες φορές υπάρχουν πολλά μέλη που παρευρίσκονται και ζητάνε και πολλά μέλη το λόγο και βέβαια ε, ξεφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο από το χρονοδιάγραμμά μας. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, εγγυόμαστε την τήρηση του χρονοδιαγραμματός. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα από τα διάφορα. Επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 19 και 20 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.